Guten Morgen, meine Damen und Herren, liebe Kolleginnen, liebe Kollegen. Ich äh, möchte ganz pünktlich beginnen. Θέλουμε να αρχίσουμε στην ώρα μας. Παρόλο που δεν είμαστε όλοι εδώ, αλλά έχουμε μια ημερησία διάταξη πάρα πολύ βαβαρημένη και σήμερα και αύριο και γι' αυτό θα πρέπει να εκμεταλλευτούμε το χρόνο μας κατά το καλύτερο δυνατόν. Θα ήθελα στην αρχή να σας πω, παρόλο που είναι σε λίγη να το ακούσουμε, ότι έχουμε 20 λεπτά για κάθε σημείο της μερικής διάταξης. Θα το φροντίσω αυτό, γιατί αλλιώς θα είμαστε μέχρι και το Σάββατο εδώ και δεν νομίζω θα ενδιαφέρεστε πάρα πολύ για κάτι τέτοιο. Έχουν αλλάξει κάποια σημεία της ημερησίας διάταξης. Δεν θα σας τα αναφέρω όλο αυτό, το έχετε όμως το χαρτί μπροστά σας. Και αυτό ε, οφείλεται στο γεγονό ότι κάποιοι συνάδελφοι με παρακάλεσαν γιατί θα έρθουν αργά, θα φύγουν νωρί ή κάτι τέτοιο τέλο πάντων. Οπότε δεν χρειάζεται να αναφερθώ σε αυτά. Εντάξει. Λοιπόν, ε, γίνεται δεκτή η ημερησία διάταξη όσο έχει δεχ... τροποποιηθεί. Ωραία, δεν διαφωνεί ημερησια διαταξη οσο εχει τροποποιηθει ωραια δεν διαφωνει κανενα Σαν εκείνο που είχα να σα πω, τι έκανα. Πάει και αυτό πρακτικά το το στις 20 Νοεμβρίου, 9 10 Νοεμβρίου και 2 3 Δεκεμβρίου. Τα έχετε στο φάκελό σας, δεν βλέπω να διαφωνεί κανένας. Εντάξει, οπότε μπορούμε να περάσουμε στη συζήτηση. Αν δεν κάνω λάθος, το πρώτο σημείο είναι το σημείο 7. Κοινό πρόγραμμα έρευνας και ανάπτυξης στη Βαλτική θάλασσα. Η συνάδελφος ΕΚ είναι παρούσα, υπεύθυνη και έχει και το λόγο. Παρακαλώ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Αυτή η έκθεση αφορά τη Βαλτική θάλασσα που είναι ένα από τα μεγαλύτερα σώματα υδατός που έχει μεγάλη επίπτωση στα ευρωπαϊκά κράτη που την περιτυχίζουν. Υπάρχουν πάρα πολλές πιέσεις στο ε, σώμα νερού αυτό λόγω της υπερτροφίας, της ε, αλλαγής της κλιματολογικής κλπ. Αυτό μειώνει τη δυνατότητά της αηφορία και προσφορά υπηρεσιών σε όλου. Έχει επίπτωση στην υγεία των κατοίκων γύρω από τη Βαλτική, έχει επιπτώσεις στην περιφερειακή ανάπτυξη των περιοχών γύρω από τη Βαλτική, έχει σημαντικές επιπτώσεις στην Αλία στον τουρισμό και ούτω καθεξής. Η προστασία της Βαλτικής θάλασσας η συνεργασία μεταξύ των χωρών της Βαλτικής έχει μακρό ιστορικό. Ήδη το 1974 7 χώρες υπέγραψαν την σύμβαση του Ελσίνκη. Αυτό ανέφερε ότι όλες οι πηγές μόλις της θάλασσας θα υπάρχουν σε μία σύμβαση. Από τότε οι χώρες αυτές προσπάθησαν να δημιουργήσουν ένα σύστημα διαχείρισης για να διατηρήσουν την αηφορείο και αηφοροχρήση του συστήματος της Βαλτικής. Αν κοιτάξετε τη γεωγραφία θα δείτε ότι οι κύριες ε, πλημμύρες και τα κύρια σώματα ε, ποταμών έχουν επίδραση μακρά μέσα στα κράτη τα ίδια. Εδώ και πολλά χρόνια η Βαλτική έγινε μια εσωτερική θάλασσα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και απαιτεί κοινή δράση στο ευρωπαϊκό επίπεδο για να αντιμετωπιστεί αυτή η ευρωπαϊκή πρόκληση και να υποστηριχθούν οι περιοχές γύρω από τη Βαλτική. Πολλές ερευνητικές δραστηριότητες γίνονται στην περιοχή αυτή Παρ' όλα αυτά, πολλές από τις αυτές δεν είναι συντονισμένες, είναι καταδεκαιρματισμένες και εξαρτώνται από τις ε, πενιχρές δυνατότητες ε, των περιφερειών και της τοπικής αυτοδιόδεσης. Γι' αυτό χρειάζεται μια συντονισμένη δράση για ένα πρόγραμμα κοινό. Για να πετύχουμε μια εφόρη συνεργασία και συντονισμό μεταξύ των ε, χωρών που είναι γύρω από τη Βαλτική, Οκτώ χώρες, Βαλτική, Δανία, Εστονία, Φιλανδία, Γερμανία, η Λετωνία, Λιθουανία, Πολωνία και η Σουηδία, ξεκίνησαν ένα κοινό πρόγραμμα έρευνας για τη Βαλτική με συμμετοχή της κοινότητας βάσει στο άρθρο 169 της Συνθήκης. Και το πρόγραμμα αυτό λέγεται Bonus 169. Αυτό το πρόγραμμα θέλει να συντονίσει την έρευνα και την ανάπτυξη των συμμετοχουσών χωρών σε ένα κοινό πρόγραμμα για την επιτύχηση των περιβαλλοντικών στόχων της στρατηγικής για την Βαλτική που αποφασίστηκε το περασμένο έτος. Ένας από τους κύριους στόχους του προγράμματος είναι να βοηθήσει την διαμόρφωση της ε, περιφέρειας και το πρόγραμμα Bonus 169 ακολουθεί το Bonus Aeronet και το Aeronet Plus αυξάνοντας το ποσοστό ολοκληρώσης και εξελίφοντας τα εμπόδια μεταξύ των συμμετεχόντων κρατών. Ξέρετε ότι αυτό δεν είναι εύκολο. Το ξέρουμε όλοι ότι δεν είναι εύκολο. Αλλά παρόλα αυτά είναι σημαντικό. Και βέβαια θα μπορέσει να συμμετάσχει και η Ρωσία, μια που η Ρωσία είναι πάρα πολύ σημαντική, μια που μολύνει πάρα πολύ τη Βαλτική. Όπως είπα, το πρόγραμμα Bonus βασίζεται στο άρθρο 169, γι' αυτό αποκαλείται Bonus 169, που προβλέπει συμμετοχή κοινή στα προγράμματα έρευνας των κρατών μελών συμπεριλαμβανομένους και τη συμμετοχή στις δομές για την εκτέλεση των προγραμμάτων αυτών. Δεύτερον, οι στόχοι του πόνους είναι σύμφωνη με τους κύριους στόχους του εβδομου προγράμματος πλαισίου και ειδικών προγραμμάτων συνεργασίας για να μπορούν να συμβάλλουν στην αηφόρο ανάπτυξη και συγκεκριμένα προγράμματα περιβαντολογικής έρευνας. Οι συμμετέχουσες χώρες συμφώνησαν ότι η δομή της ε, πραγματοποίησης του πόνους θα βασίζεται σε μια ευρωπαϊκή οικονομική ομάδα που λέγεται ε, Bonus EIT e <clears throat> και που έχει ιδρυθεί στη Ελσίνκι στην Φιλανδία. Η Κομισιόν υποσχέθηκε και το χαιρετίζουμε αυτό να συμβάλλει μέχρι 50 εκατομμύρια ευρώ για όλη τη διάρκεια του μπόνους για τα επόμενα δηλαδή 7 χρόνια. Και νομίζω ότι πραγματοποιώντας κάτι τέτοιο θα πρέπει να προσπαθήσουμε να πετύχουμε τους στόχους μας και αυτό να είναι κατά δυνατόν αποτελεσματικό και να αποφύγουμε την πλεονασματική γραφειοκρατία. Δεν πιστεύω ότι θα πρέπει να ε, εισαγάγουμε νέα δημοκρατικά, ε, γραφειοκρατικά μέτρα των αντίον. Και είδαμε στην ε, μήνυα ακρόαση το φθινόπερο ότι όλα τα πανεπιστήμια και όλες οι οργανώσεις και τα σώματα που συμμετείχαν τόνισαν ακριβώ αυτά τα προβλήματα. Διαμακρών μάλιστα. Η πρόταση Κομισιόν για τη συμμετοχή της κοινότητας στον πόνους είναι σύμφωνη και με την πολιτική γραμμή του Κοινοβουλίου για την ε, βελτίωση του συνολισμού των ερευνητικών δραστηριοτήτων, πράγμα που έχουμε συζητήσει πλιστάκι. Εάν εφαρμόσουμε το πρόγραμμα αυτό σωστά, θα μπορούσε να αποτελέσει πρότυπο για άλλε μορφέ ε, περιφερειακή συνεργασία, παραδείγματο χάρη, νο... Βόρεια Θάλασσα, Μεσόγειο και ούτω καθεξής. Έχουμε λοιπόν την δυνατότητα να προσφέρουμε έτσι ένα μοντέλο για περιφερειακή συνεργασία. Είναι πάρα πολύ σημαντικό λοιπόν τι θα κάνουμε με τον πόνους γιατί θα μπορεί να είναι παράδειγμα για άλλες περιοχές. Υπάρχουν δύο κυρίως προβλήματα που θα πρέπει να συζητήσουμε και τα οποία συζητηθήκαν στο Συμβούλιο και στην Κομισιόν. Το πρώτο είναι η δομή δύο σταδίων. Στην πρώτη της Κομισιόν το πόνος θα πρέπει να εφαρμοστεί σε δύο φάσεις. Στο παρελθόν η συζήτηση αυτή για τις δύο φάσεις αφορούσε την εφαρμογή. Τώρα η Κομισιόν θέλει να εισαχθεί μια δομή στην έρευνα με δύο φάσεις. Καταρχήν στρατηγική φάση. Τα πρώτα δύο χρόνια θα πρέπει να γίνει διαβούλευση και να καθοριστούν οι πλατφόρμες για τους ενδιαφερόμενους, να προετοιμαστεί η σχετική ατζέντα έρευνας και ο τρόπος εφαρμογής. Και κατόπιν θα υπάρχει μια φάση εφαρμογής 5 ετών όπου θα λάβει χώρα η έρευνα. Και εκεί θα υπάρχουν ε, διάφορα συγκεκριμένα προγράμματα που θα αντιμετωπίζουν και θα προσπαθούν να βρει λύσει για τους στόχους της πρωτοβουλίας. Έχοντας κατά τη μακρά ε, ιστορία συνεργασία στον τομέα της έρευνας, Υπάρχει ήδη μία ε, δομή για τη χρηματοδότηση και άλλα θέματα και θα πρέπει να τα συζητήσουμε αυτά αναλυτικά και θα χαρώ πάρα πολύ να ακούσω τις απόψεις σας. Κατά τη διάρκεια της το δίκτυο χρηματοδότηση, το EIG, συμφώνησε με την πρώτη Κομισιόν για την διτή αυτή ε, προσέγγιση, για τις δύο αυτές φάσεις. Υπάρχουν όμως διαφορετικές ερμηνείες της αρχής, γι' αυτό πρέπει να το συστήσουμε το θέμα. Μετά από την πρώτη φάση, η Κομισιόν θα αξιολογήσει την οριμότητα και την προετοιμασία της πρωτοβουλίας και αν τα αποτελέσματα της είναι θετικά θα προχωρήσει στην συμφωνία εφαρμογής με το Πόνος ΑΕΓ. Αυτή δεν θα είναι μια απόφαση ναι ή όχι, γιατί είμαστε σίγουροι ότι θα πρέπει πραγματικά να πραγματοποιηθεί το πόνος. Η αξιολόγηση λοιπόν θα πρέπει να έχει σαν στόνο την αποτελεσματικότητα της δομής. Δεν θα είναι μια απόφαση κατά πόσον θα πραγματοποιηθεί ή όχι αυτό το πρόγραμμα. γιατί αλλιώς θα χάσουμε τη συμμετοχή των ερευνητών και θα χάσουμε και χρόνο και ορμή. Το άλλο θέμα που θα πρέπει να συζητήσουμε είναι πώς θα πρέπει να πραγματοποιηθεί η χρηματοδότηση. Και εδώ προβλέπεται ένα σύστημα κοινών μερών. Στην πρόταση της Κομισιόν όλες οι συμμετέχουσες χώρες θα πρέπει να συμβάλλουν σε ένα κοινό ταμείο. Ξέρουμε ότι τα διάφορα κράτη-μέλη έχουν διαφορετική συμμετοχή. Ε, ο τρόπος δηλαδή χρηματοδότηση θα μπορεί να γίνει διαφορετικά. Με χρήματα, με άτομα, με υποδομές, με οτιδήποτε τέλος πάντων. Γιατί χρειάζεται ένα κοινό ταμείο. Γιατί από σκοπιά της Κομισιόν είναι καλύτερο γιατί ίσως σε κάποιες ασυμμετέχουσες χώρες έχουν προβλήματα νομικά ή ε, διοικητικά και δεν μπορούμε να περιμένουμε να αλλάξει το σύνταγμα σε κάποια από τις συμμετέχουσες χώρες για να μπορέσουμε να προχωρήσουμε με το πρόγραμμα και γι' αυτό θα πρέπει να βρούμε κάποιο κοινό τορβανά αν θέλετε στο οποίο θα συμβάλλουν όλοι και από το οποίο θα μπορέσουν να συμβάλλουν από εκεί και πέρα στην χρηματοδότηση των διαφόρων σχεδίων. Πρέπει να έχουμε μία εφαρμόσιμη λύση βέβαια, να αποφύγουμε τα νομικά προβλήματα. Ταυτόχρονα όμως θα πρέπει να εξασφαλιστούν οι κοινοτικοί στόχοι της πρότασης. Τούτων εχθέντων δεν θα ήθελα να μακρηγορήσω, γι' αυτό θα σταματήσω εδώ και θα ακούσω με ενδιαφέρον τις απόψεις των συναδέλφων. Γιατί αυτό το σχέδιο είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό πρόγραμμα όσον αφορά το περιεχόμενο και τους στόχους, αλλά και η μορφή του θα μπορούσε να είναι ένα παράδειγμα για περιφερειακή συνεργασία. Σας ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρο. Εγώ σας ευχαριστώ, κύριε συνάδελφε. Συνάδελφος και έχει το λόγο. Ε, Ευχαριστώ πολύ. Είναι σαφές ότι συζητάμε για ένα πολύ σημαντικό πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Τι είναι η Βαλτική θάλασσα? Η Βαλτική δεν είναι ακριβώς η φάλμηρη λιμνοθάλασσα, είναι κατά προσέγγιση η φάλμηρη θα έλεγα. Και το πρόβλημα είναι ότι πολλές φορές ε, παγώνει και πάγωνε κατά το παρελθόν σε μεγάλο βαθμό. Άρα δηλαδή εκεί ε, εντοπίστηκαν ανθρωποειδοί. Και ού αυτό, αλλά στις ε, εκβολές προς τη θάλασσα υπήρξαν εξωγενή, ε, ε, διαπιστώθηκαν εξωγενείς, ε, εξωγενή μορφώματα. Γι' αυτό λοιπόν θεωρώ ότι θα πρέπει τελικά να καταλήξουμε στο τι είδους νερά είναι αυτά που καταλήγουν μέσω του ποταμού Όντερ στη θάλασσα. Η Ρωσία συμβάλλει και αυτή στη μόλυνση στη ρήπανση της ε, λιμνοθάλασσας. Μπορεί λοιπόν να πει κανείς ότι κατά 90% είναι λιμνοθάλασσα της Ευρωπαϊκής ε, και της Ευρώπης και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά υπάρχει και αυτό το 10% της Ρωσίας. Η Ρωσία λοιπόν σύντομα θα κατασκευάσει ε, τον αγωγό της Βαλτικής θάλασσας το ύψος της επένδυσης έχει ήδη καθοριστεί και νομίζω ότι σε αυτό το πρόγραμμα η Ρωσία θα διαδραματίσει σημαντικό ρόλο. Έχω κατά νου τη συνεργασία ανάμεσα στην ε, Ευρωπαϊκή Ένωση και τη Ρωσία και αυτό είναι κάτι που πρέπει να το λάβουμε υπόψη μας. Όσον αφορά τώρα τη χρηματοδότηση αυτού του προγράμματος, εγώ θέλω να κάνω τέσσερις παρατηρήσεις επ' αυτού. Real Common Pot, όπως ε, αναφέρεται στα αγγλικά από το 7ο πρόγραμμα πλαίσιο γνωρίζουμε ότι η γραφειοκρατία οδηγεί σε μεγάλες καθυστερήσεις και γι' αυτό φοβούμεθα ότι τα κονδύλια αυτά τα οποία εμείς θα διοχετεύσουμε σε αυτή την κοινή δεξαμενή, σε αυτό το ε, κοινό καζάνι αν θέλετε, δεν θα τύχουν σωστής εκμετάλλευσης. Γι' αυτό λοιπόν προτείνουμε ένα μείγμα χρηματοδότησης ή ένα virtual common pot όπως θα το αποκαλούσα στα αγγλικά. Αυτή είναι η πρώτη μου παρατήρηση. Δεύτερη παρατήρηση αφορά σε αυτές τις δύο φάσεις ε, της μεταβατικής περίοδου. Κατά την πρώτη φάση πρέπει να λάβουν χώρα αναλύσεις και να ληφθούν αποφάσεις. Θα πρέπει όμως να λάβει χώρα και μία περαιτέρω ανάλυση, ένα είδος ορόσημου όπως αποκαλείται, ε, ένα ορόσημο το οποίο θα οδηγήσει σε μία παράταση του χρονικού διαστήματος ερευνών μέχρι να περάσουμε στη δεύτερη φάση. Και εδώ θέλω να προσθέσω ότι κατά το παρελθόν υπήρξαν παρεμφερή προγράμματα ρυθμίσεις ε, για περισσότερο ηλικιωμένα άτομα, για μικρομεσαίες επιχειρήσεις, ε, ρυθμίσεις για τη μέθοδο. Θεωρώ λοιπόν ότι θα ήταν ε, σκόπιμο το σύνολο της τεκμηρίωσης να έχει μια ενιαία μορφή, γιατί αυτό θα αποτελεί διευκόλυνση. Και τώρα η τέταρτη παρατήρηση εκ μέρους μου κατατέθηκε μία πρόταση να υπάρξει προσπελάσιμη υποδομή για τις χώρες εκείνες που θα συμμετέχουν στη χρηματοδότηση. Πρέπει να πω ότι η πρόταση αυτή είναι και λεπτομερής και περιοριστική. Η κοινή χρήση της ε, προσπελάσιμης υποδομής, κατά τη δική μου άποψη, είναι κάτι το οποίο χρήζει περαιτέρω συζητήσεων. Και νομίζω ότι η γραμματεία της Επιτροπής που είναι αρμόδια για αυτό το πρόγραμμα των πόνους θα πρέπει να μας δώσει τις απαραίτητες ε, λεπτομέρειες. Ο κύριος Μπαλσίτης ε, παρακαλώ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Πράγματι, ε, θα ήθελα να εκφράσω τη χαρά μου για το γεγονός ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποδίδει ιδιαίτερη σημασία στη, στο πρόγραμμα για τη Βαλτική θάλασσα. Με το πρόγραμμα αυτό βελτιώνει κατάσταση στο σύνολο της περιοχής. Θα ήθελα λοιπόν να συγχαρώ την κυρία Εκ, γιατί η κυρία Εκ ε, πραγματικά παρουσίασε μια θαυμάσια έκθεση, επεξεργάστηκε ένα τεκμηριωμένο έγγραφο και θέλω να ελπίζω ότι το έγγραφο αυτό θα καταστεί εύκολο να εφαρμοστεί στην πράξη. Και επιτρέψτε μου να κάνω κάποιες παρατηρήσεις από αυτού. Πρώτα απ' όλα, θα ήθελα να αναφερθώ σε δύο φάσεις, σε δύο χρονικά διαστήματα. Ε, δηλαδή, δεν ήθιστε το, τα προγράμματα να ε, διαχωρίζονται αυστηρά σε δύο φάσεις. Και όταν μιλάμε για ανεξάρτητους εμπειρογνώμονες και για τη δική τους την ανάλυση. Εγώ πιστεύω ότι το χρονικό διάστημα που προβλέπετε είναι πολύ αυστηρό και θεωρώ ότι θα αρκούσε ε, τα κράτη-μέλη να μιλήσουν ε, από κοινού για τα ερευνητικά προγράμματα και αργότερα στη φάση υλοποίησης του προγράμματος εκεί τα κράτη-μέλη μπορούν με τους εμπειρογνωμονές τους να συζητήσουν ή να συζητήσουν και μεταξύ τους και αυτή η συζήτηση θα μπορούσε να συμβάλλει έτσι ώστε ε, πολλά κράτη-μέλη να εφαρμόσουν την ίδια χρονική στιγμή το πρόγραμμα. Και δεύτερη παρατηρήσή μου σε αυτό το ε, την κοινή δεξαμενή, το κοινό ταμείο θέλετε. Δεν θέλω να επαναλάβω αυτά που είπαν οι συνάδελφοί μου ή τα κονδύλια που θα διοχετευθούν σε αυτό το κοινό ταμείο βεβαίως και θα συμβάλλουν στην επίλυση πολλών προβλημάτων. Από την άλλη βέβαια πλευρά υπάρχουν πολλά ε, νομικής φύσεως ε, κολλήματα σε ορισμένα κράτη-μέλη και είναι αδύνατο να διοχετεύσουμε κονδύλια χωρίς στόχο, χωρίς συγκεκριμένο σκοπό, έτσι γενικά και αόριστα. Αυτό ε, δεν θα συμβάλλει στην υλοποίηση του προγράμματος. Νομίζω λοιπόν ότι η Κομισιόν πρέπει να λάβει υπόψη της αυτές τις δύο παρατηρήσεις και να καταρτήσει τη στρατηγική της με τέτοιο τρόπο έτσι ώστε να ε, μπορεί να εφαρμοστεί η στρατηγική αυτή το συντομότερο δυνατόν. Ο κύριος Βανίς Σήμερα, ε, ε, θα κάνουμε την πρώτη ανταλλαγή απόψεων και αργότερα μπορούμε ίσως ε, να επανέλθουμε. Θα ήθελα λοιπόν ε, να μιλήσω για την για την προσέγγιση αυτή. πρέπει πράγματι να υπάρχει μια, ένα σωστό αρχιτεκτονικό οικοδόμημα για την έρευνα. Αλλιώς η έρευνα θα είναι κάπου στον αέρα ε, χωρίς να υπάρχει και επίλυση των ε, προβλημάτων. Θα πρέπει λοιπόν να ασχοληθούμε όχι μόνο με την ε, βασική έρευνα αλλά να δούμε λιγάκι ευρύτερα το πρόγραμμα και το πρόβλημα μάλλον της Βαλτικής. Θεωρώ λοιπόν ότι η πρώτη φάση είναι πολύ δύσκολη. Ε, υπάρχουν τα κονδύλια τα οποία διοχετεύονται σε ένα ταμείο αλλά πρέπει να μεριμνήσουμε να χρησιμοποιηθούν σωστά αυτά τα κονδύλια. Η λιδία λήθος ε, σε όλο αυτό το πρόγραμμα είναι κατά πόσον η συνεργασία στη Βαλτική οδηγεί πράγματι σε κοινή χρηματοδότηση και στην επεξεργασία προγραμμάτων τα οποία πρέπει να εφαρμοστούν. Πρόκειται για κοινή χρηματοδότηση και συζητάμε για πράγματα τα οποία σχετίζονται με την περιφερειακή πολιτική, με επενδύσεις ε, Ε, αναφέρθηκε και προηγουμένως, ε, χρήματα υπάρχουν. Το θέμα είναι μόνο ε, πού θα διοχετευθούν τα κονδύλια αυτά. Γι' αυτό λοιπόν είναι πολύ σημαντικό να αναλυφθούν και κάποιες υποχρώσεις. Και νομίζω ότι είναι καλύτερα να μιλήσουμε διεξοδικά, να δαπανίσουμε περισσότερο χρόνο στις συζητήσεις πριν ο καθένας καταλήξει στην εκταμείωση των κονδυλίων. Εγώ λοιπόν τάσομαι υπέρ της διατήρησης των δύο φάσεων. Και θα ήθελα επίσης να πω το εξής. Οι επιπτώσεις από αυτές τις δύο φάσεις είναι πολύ σημαντικές για τη φάση εκτέλεσης του προγράμματος. Γι' αυτό λοιπόν σας προειδοποιώ να μην ε, επιταχύνουμε και να βιαστούμε να λάβουμε αποφάσεις οι οποίες μετά δεν θα μπορούν να εφαρμοστούν. Αυτό είναι πολύ σημαντικό και δεν θα πάψω να το τονίζω. Ε, κατά τα άλλα υπάρχουν και άλλες ε, λεπτομέρειες που αφορούν στην εφαρμογή εγώ συμφωνώ ότι η Βαλτική πράγματι αποτελεί ε, μία περιοχή πρότυπο. Το κοινοβόλιο τάχθηκε υπέρ αυτού και το θέμα που τίθεται είναι πώς ακριβώς μπορούμε να συμμετάσχουμε σε καινοτόμα προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και όχι μόνο αυτό, αλλά πώς ε, η Κομισιόν θα δραστηριοποιηθεί στην περιοχή. Μακροπρόθεσμα θεωρώ ότι η περιοχή αυτή μπορεί να αποτελέσει το παράδειγμα για πολλές άλλες που θα ακολουθήσουν. Φοβάμαι ότι ε, θα μπορούσαμε να συζητάμε στο δινεκές ε, χωρίς να καταλήγουμε σε συγκεκριμένα προγράμματα. Ε, και αν θέλουμε να συμπεριλάβουμε και τη Ρωσία σε αυτό το πρόγραμμα, γιατί όχι. Και η Ρωσία σε τελική ανάλυση θα πρέπει να ενδιαφέρεται και θα μπορούσε να προκύψει μια περαιτέρω συμφωνία ανάμεσα στη Ρωσία και την ε, Ευρωπαϊκή Ένωση. Έχω ε, άλλη μία... Ε, άλλος ένας έχει το λόγο για να παρέμβει, ο κύριος Ματή από την Κομισιόν. Σας ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θα ήθελα καταρχήν να ευχαριστήσω την εισηγήτρια για την έκθεση αυτή για το πρόγραμμα Πόνιους. Θα ήθελα να τονίσω ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στηρίζει έντονα την πρόταση. Ήταν αντικείμενο η πρόταση αυτή μια συσβάθος ανάλυσης και μια συνεχούς εργασίας εδώ και δύο έτη. Μια εργασία η οποία έγινε από κοινού με την ε, ομάδα Bonus που είναι στο Ελσίνκι. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σκέφτηκε πάρα πολύ πάνω στον τρόπο να προχωρήσει και θα ήθελα να τονίσω τη στρατηγική σημασία της πρώτης φάσης, της λεγόμενης στρατηγικής φάσης δηλαδή, που επιτρέπει να αναπτυχθούν με τους συμμετέσχοντες ε, οι στρατηγικές ατζέντε ε, έρευνας που θα υποστηρίξουν την ευρωπαϊκή πολιτική. Και θα ήθελα να πω επίσης ότι το πρόγραμμα Bonus είναι σημαντικό για την ε, Βαλτική, αλλά είναι πάρα πολύ σημαντικό επίσης για τη δομή του Ευρωπαϊκού Χώρου Έρευνας. Είναι λοιπόν ένα παράδειγμα που θα μας χρησιμεύσει για το μέλλον. όσον αφορά αυτό το κοινό ταμείο, το κοινό τορβανά αυτό, το... θα ήθελα να πω ότι βασίζεται και σα... Ε, έχουμε και άλλες φορές βασιστεί στο άρθρο 169, έκθεση Φανβέλτζεν, παραδείγματος χάρη, όπου η Κομισιόν αποδίδει ιδιαίτερη σημασία στις, ε, στα συμπεράσματα της έκθεσης Φανβέλτζεν και γι' αυτό ακριβώς προτείνουμε την εφαρμογή του προγράμματος αυτού που θα βασίζεται σε ένα κοινό ταμείο γιατί έτσι θα μπορέσουμε πιο γρήγορα να, να εφαρμόσουμε το πρόγραμμα. Σας ευχαριστώ Πρόεδρε. Danke sehr, Monsieur Audi. Eine Minute. Wir müssen jetzt auf die Zeit gucken. Euh, για να αναρωτηθώ για το ρόλο των κρατών μελών ε, για τις κοινωτικές πολιτικές ε, όπως αυτή. Η σύγκριση γίνεται με τη Μεσόγειο είναι μία από τις πιο μολυσμένες θάλασσες ε, του κόσμου και πρέπει να προσέξουμε και στην αρχή ε, αναφερόμαστε στα κράτη-μέλη ε, που βρέχονταν από τη Μεσόγειο, ενώ τώρα αναφερόμαστε στα κράτη που συμμετέχουν ε, στην Ευρωμεσογειακή διάσκεψη. Τώρα, Ποιος είναι ο ρόλος των κρατών μελών, αυτό πρέπει να αναρωτηθούμε. Πρέπει ε, να ασχοληθεί το σύνολο της Ένωσης τελικά με το θέμα αυτό ή πρέπει να ασχοληθούν μόνο τα κρατημέλη της Μεσογείου. What? Will die Präsidentschaft auch noch was an der Rat? No. It's your turn. Nobody wants. No. Okay. Ε, σας ευχαριστώ. Κοιτάξτε, θα ήθελα να ευχαριστήσω όλα τα μέλη για τις πολύ χρήσιμες παρεμβάσεις τους σε αυτή τη συζήτηση. Πρώτα απ' όλα, όσον αφορά στη Ρωσία, όλοι μας αναγνωρίζουμε τον ιδιαίτερα σημαντικό ρόλο της Ρωσίας. Όχι μόνο λόγω του ότι η Ρωσία είναι γεωγραφικά μία από τις χώρες ε, γύρω από τη Βαλτική, αλλά και διότι ένα μεγάλο τμήμα της ρήπανσης προέρχεται από τη Ρωσία. Επίσης, ε, η ε, Ρωσία στη Βαλτική είναι μια χώρα που εξάγει μεγάλες ποσότητες ενέργειας, όχι μόνο αερίου. Και υπάρχει και αυτή η έντονη κίνηση του στόλου στη Ρωσία και στη Βαλτική. Άρα δηλαδή η Βαλτική ε, δίνει τη δυνατότητα στη Ρωσία να συνδεθεί ε, τόσο με ε, κονδύλια όσο και με το να προσφέρει στην υποδομή και αυτό είναι πάρα πολύ καλό. Αυτό λοιπόν είναι ένα θέμα που είναι κοινό, ορίζεται ως τέτοιο και είναι πάρα πολύ σημαντικό ε, είναι ένα θέμα όπου πραγματικά πρέπει να προχωρήσουμε. Και εδώ πρέπει να υπάρχουν τρία προγράμματα που βασίζονται στο 169. Ε, το ένα είναι αφορά το περιβάλλον, το δεύτερο αφορά το πρόγραμμα για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και το τρίτο αφορά σε ε, μετρήσεις μετερολογίας. Ε, εδώ βλέπουμε ότι η Κομισιόν προτείνει μια διαφορετική υποδομή σε ένα τέταρτο πρόγραμμα που είναι μεγαλύτερη υποδομή, που καλύπτει περισσότερες περιοχές, που είναι πολύ πιο δύσκολη η υποδομή αυτή. Ίσως λοιπόν θα ήταν σκόπιμο να σκεφτούμε σε βάθος ε, το θέμα της ε, στρατηγικής και το πώς ακριβώς πρέπει να οργανώνεται η συνεργασία για να καλύπτονται οι στόχοι του προγράμματος Bonus. Τώρα, όσον αφορά τη δράση μας. Αν ανοίξουμε μια ματιά στην κατάσταση που υπάρχει στις ε, χώρες ε, και στην ε, περιοχή, στις χώρες που περιβάλλουν τη Βαλτική, κυρίως στις νέες χώρες, θα διαπιστώσουμε ότι εκεί υπάρχει ανάγκη οικονομικής βελτίωσης και απομόλυνσης, απορρίπανσης της περιοχής. Ε, βλέπουμε ότι αυξάνεται συνεχώς ε, η ρήπανση. Αυτό είναι ένα μεγάλο πρόβλημα. Για την ε, αλία η κατάσταση είναι ιδιαίτερα οξία. Βλέπουμε λοιπόν τη Βαλτική θάλασσα που είναι μια μοναδική θάλασσα, αντιμετωπίζει ιδιαίτερα έντονα προβλήματα και οι άνθρωποι που ζουν στην γύρω από τη Βαλτική πραγματικά χρειάζονται το να υπάρξει βελτίωση για να βελτιωθεί τη υγεία τους, ε, να βελτιωθεί το επίπεδο της διαφύωσής τους, να υπάρξει ε, περιφερειακή οικονομική ανάπτυξη και τέλος να αντιμετωπιστεί και το πρόβλημα του ε, περιβάλλοντος. Και θέλουμε και πρέπει να δούμε και τι συμβαίνει με το υδάτινο, το πρόβλημα ύδατος στη Βαλτική. Είναι λοιπόν πολύ σημαντικό όλα αυτά να γίνουν με το σωστό τρόπο, με πρακτικό και αποτελεσματικό τρόπο, να χρησιμοποιούνται ε, λοιπόν ε, οι πόροι ε, σωστά, ε, αυτό προφανώς είναι πρώτη προτεραιότητα της Κομισιόν και της έρευνας. Ε, θεωρώ ότι η βελτίωση θα μπορούσε να αποτελέσει παράδειγμα για το μέλλον. Ο πρόεδρος αναφέρθηκε στο χρονοδιάγραμμα. Εγώ θα ζητήσω να υπάρξει μια συνάντηση με τους ε, συντονιστές κατά προτίμηση στο Στρασβούργο όπου θα μπορέσουμε να δούμε λιγάκι το κείμενο. Η έκθεση θα σταλεί για μετάφραση την Παρασκευή της επόμενης εβδομάδας. Έχουμε λοιπόν ένα πολύ σφιχτό χρονοδιάγραμμα και αν τελικά συμφωνήσουμε πάνω σε ένα καλό κείμενο, πράγμα το οποίο ε, ελπίζω διακαώς, θα μπορέσουμε να ψηφίσουμε τον Ιούνιο ή το αργότερο τον Ιούλιο, έτσι ώστε να ε, μπορέσουμε να προχωρήσουμε με το να καλύψουμε τις ανάγκες στη Βαλτική και ε, τις ανάγκες των ανθρώπων που ζουν γύρω από τη Βαλτική. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, λέει ο Πρόεδρος. Είπατε τα σημαντικότερα. Εγώ θέλω μόνο να προσθέσω κάτι. Εχθές ε, είχα συζητήσεις ε, με την Ισπανική Προεδρία, η οποία με παρακάλεσε οριζόντια ε, σε όλες τις θήσεις που θα έχουμε ή δυνατόν να επιτύχουμε συμφωνία κατά την πρώτη ανάγνωση. Εγώ βέβαια πιστεύω ότι πρέπει να ακολουθήσουμε την πεπατημένη και η συμφωνία στην πρώτη ανάγνωση είναι η εξαίρεση, αν κάτι δηλαδή πιέζει χρονικά. Και εμείς αυτό να κάνουμε, αυτό να ακολουθήσουμε. Αν βέβαια υπάρξει κάτι έκτακτο θα επιδείξουμε ευελιξία. Και εσείς είπατε είπατε, να προχωρήσουμε γρήγορα, αλλά να αφήσουμε και τον χρόνο που χρειαζόμαστε. Η Κομισιόν άφησε τον εαυτό τη χρόνο για να προετοιμαστεί, το ίδιο σκοπεύουμε να πράξουμε κι εμεί. Αυτή είναι η δική μου παράκληση. Σα ευχαριστώ πάρα πολύ. Ε, από πλευρά ε, χρόνου τώρα του δικού μα προδιαγράμματο, κλείσαμε με το θέμα αυτό και αν προχωρήσουμε σήμερα όπως σήμερα, κοίταξε για τώρα ε, χρησιμοποίησαμε διπλάσιο χρόνο από ό,τι έπρεπε και αν συνεχίσουμε έτσι δεν θα μπορέσουμε να συζητήσουμε τουλάχιστον δύο-τρει εκθέσεις. Γι' αυτό λοιπόν ξανά παρακαλώ να προχωρήσουμε με μεγαλύτερη ταχύτητα. Επόμενη εκθέση είναι η ενδιάμεση επισκόπηση των Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων Δορυφορικής Πλήγησης. Ο συνάδελφος κ. Ρέμεκ είναι ο συγητή, ο οποίο έχει και το λόγο. Παρακαλώ. Ε, ε, ε, Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Έχουμε τη δυνατότητα τώρα από τη Βαλτική να πάμε στο διάστημα και ελπίζω ότι στη συνέχεια θα μπορέσουμε να επανέλθουμε στη γη, να προσθαλασσοθούμε αν θέλετε. Νομίζω ότι είναι πλεονέκτημα να δούμε αυτά τα διαφορετικά συστήματα και πώς μπορούμε να τα χρησιμοποιήσουμε ε, είτε σε χερσαίο είτε σε θαλασσιοπίπεδο. Αγαπητοί συνάδελφοι, η δική μου έκθεση παρουσιάζει κάποιες πτυχές. Θα προσπαθήσω εγώ να επικεντρωθώ στα πιο σημαντικά θέματα. Θέλω να πω ότι η έκθεση αυτή περιλαμβάνει, βασίζεται μάλλον σε μία σειρά εγγράφων. Υπάρχει επίσης ε, και η έκθεση του κ. Γκλάν και του κ. Τωσονοφσκή. Βασιζόμαστε και στις εκθέσεις αυτές. Και νομίζω ότι αυτό το σύστημα συνεργασίας με τους δύο εισηγητές είναι εξαιρετικό. Πιστεύω ότι μία σειρά ατόμων γνωρίζουν ήδη τα έγγραφα αυτά και θα συμμετάσχουν και στο δικό μου έγγραφο, στη ζήτηση για το δικό μου έγγραφο. Νομίζω ότι αυτό είναι καλό για να υπάρχει συνέχεια στις εκθέσεις μας. Προσωπικά θεωρώ ότι είναι πολύ σημαντικό να έχουμε αυτό το έγγραφο όχι μόνο για το Κοινοβούλιο αλλά και για το σύνολο των δραστηριοτήτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης καθώς το και προγράμματα πλοήγησης αποτελούν τμήμα φιλόδοξων σχεδίων υποδομών και όπως βλέπετε για πολλούς ε, βουλευτές ε, τέτοια θέματα θεωρούνται ε, αμφίσιμα και σε ό,τι αφορά τη χρηματοδότηση αλλά και στο ότι θέλουμε να δείξουμε στους πολίτες ότι όχι μόνο μπορούμε να φανταζόμαστε προγράμματα, αλλά τα θέτουμε και σε εφαρμογή και θέλουμε να φτάσουμε σε ένα στάδιο από το οποίο θα μπορούσαν να αποφεληθούν τα κράτη. Αυτό λοιπόν επιφέρει πολύ μεγάλο πλεονέκτημα για την Ευρωπαϊκή Ένωση και είναι ευθύνη μας ως Ευρωβουλευτές να προωθούμε τα προγράμματα αυτά. Υπάρχουν και κάποια φιλοσοφικά στοιχεία στο έγγραφο αυτό, παραδείγματος χάρη το θέμα της, ε, πέρα από τα φιλοσοφικά μάλλον υπάρχει και το θέμα της χρηματοδότησης και να δούμε πώς μπορούμε να συνεχίσουμε τη χρηματοδότηση αυτού του προγράμματος και τις ε, διάφορες δραστηριότητες. Χρειαζόμαστε επαρκή χρηματοδότηση για να συνεχιστεί το πρόγραμμα στο μέλλον. Υπάρχουν και οι δαπάνες που τίθενται υπό έλεγχο, αλλά θα πρέπει να δούμε τι θα γίνει στο μέλλον και πώς θα συνεργαστούμε με τον ιδιωτικό και με το δημόσιο τομέα. Πρόκειται λοιπόν για ένα νέο είδος μοντέλο που αναπτύσσεται. Πρέπει να δούμε ποιες είναι οι δυνατότητες διεθνούς συνεργασίας και με τρίτες χώρες από άλλες υπήρους ή με άλλες χώρες στην Ευρωπαϊκή Ήπειρο. Πρέπει να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε ε, σε σχέση και με όσα γίνονται με παρόμοια προγράμματα που γίνονται στην Κίνα, στη Ρωσία, στη ΣΥΠΑ. Και θα πρέπει να εκπονήσουμε μια στρατηγική σε ευρωπαϊκό επίπεδο προκειμένου να μπορέσουμε να προωθήσουμε την ανταγωνιστικότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεν ε, πρόκειται για κάτι απλό. Γνωρίζουμε ήδη τα αποτελέσματα του Γαλιλαίου και Όλα αυτά θα είναι δύσκολο να ολοκληρωθούν, καθώς ε, το σύστημα θα λειτουργήσει όταν θα έχει ολοκληρωθεί το δίκτυο. Μόνο τότε θα μπορέσουμε να προσφέρουμε εξειδικευμένες υπηρεσίες. Πρέπει λοιπόν να λάβουν χώρα ακόμα μια σειρά εξελίξεων και δεν ε, έχουμε ακόμα ε, όλες τις δυνατότητες. Υπάρχουν μια σειρά προβλημάτων που πρέπει να επιληθούν. Αυτά λοιπόν ε, είναι κάποια σχόλια που ήθελα να κάνω. Νομίζω ότι πρέπει να προχωρήσουμε σε αυτή την αξιολόγηση και σε ένα διάμεσο στάδιο. Αλλά επίσης είναι σημαντικό να επιδιώξουμε την υλοποίηση αυτού του προγράμματος. Και πέρα από το 2013 να επικεντρωθούμε στη χρηματοδότηση, στα τεχνικά χαρακτηριστικά και στην εφαρμογή θα πρέπει να συνεχίσουμε να αναπτύσσουμε το σύστημα γιατί διακυβεύεται το γόητρο τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Ελπίζω να μπορώ να βασιστώ στη δική σα υποστήριξη και στη δική σα συνεργασία και αναμένω τα σχολιά σας. Ο κύριος ε, Μπρεζίνα, ευχαριστώ πρόεδρε. Όπως και ο θα ήθελα να πω και εγώ ότι αυτό το ευρωπαϊκό πρόγραμμα είναι πάρα πολύ σημαντικό. Θα αποτελέσει μια πηγή καινοτομία επιστημονικών ανακαλύψεων. Ουσιαστικά θέλουμε εδώ να προσφέρουμε υπηρεσίες που αποτελούν υπεραξία. η σημασία είναι τόσο μεγάλη που το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα πρέπει με προσοχή να παρακολουθήσει ε, το σύνολο ε, των διαδικασιών και θα πρέπει να ενημερώνεται το Κοινοβούλιο για τη θέση σε εφαρμογή του συστήματος αυτού. Είναι απαραίτητο να αποφύγουμε επιπλοκές όπως είχαμε στην αρχή με το πρόγραμμα Γαλιλαίο γιατί υπήρξε ένα είδος ε, κατάρρευσης, ε, αν θέλετε, της εταιρεία που είχε αναλάβει, υπήρξαν, ε, του εγχειρήματος μάλλον, και υπήρξαν προβλήματα. Έτσι λοιπόν το Κοινοβούλιο πρέπει να παρακολουθεί προσεκτικά τις εξελίξεις και ίσως ε, μπορεί να χρειαστεί και παρέμβαση των πολιτικών μας θεσμών, ακόμα και του δικού μας κοινοβουλίου. Βασίζομαι στο ότι είναι σε εξαιρετικά χέρια η έκθεση αυτή, γιατί ο κύριος Ρέμεκ είναι ο μόνος ε, ίσως στην αίθουσα αυτή που έχει τη δυνατότητα να χρησιμοποιεί τέτοιου είδους συστήματα. Έτσι λοιπόν, ε, ο κύριος Ρέμεκ έχει τις ε, απαραίτητες ε, ικανότητες και εγώ φυσικά θέλω να τον βοηθήσω ώστε το δυνατό περισσότερο. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Χόλ. Um, ευχαριστώ. Νομίζω ότι όλοι κατανοούμε ότι το Γαλιλαίο έχει να διαδραματίσει σημαντικό ρόλο γιατί παράσχει θα παράσχει υπηρεσίες στην Ευρώπη ανεξάρτητα από τα συστήματα κυβέρνησης. Επομένως, δεν μας εκπλήσει ότι το αξιολογούμε ιδιαίτερα. Αλλά είναι σημαντικό να γνωρίζουμε τι συμβαίνει και να μην υποστηρίζουμε τυφλά το Γαλιλαίο, όσο και μεγάλη πολιτική σημασία να έχει σε εμά του Ευρωπαίου, θέλω να αναφερθώ σε κάποια θέματα που προέκυψαν κατά τη διάρκεια των ακροάσεων. Ακούσαμε τον εκπρόσωπο της Κομισιόν, τον κύριο Ταϊχάν, και είπε ότι ε, υπάρχουν λιγότερα προβλήματα από ότι στον Καλλιλέο. Υπάρχουν διάφορα θέματα, αλλά θέλω να αφαιρθώ σε δύο συγκεκριμένα. Ίσως ε, ο εισηγητής να τα έχει σκεφτεί. Τι γίνεται με την ε, Κίνα, η οποία αυτή τη στιγμή μπλοκάρει το φάσμα επί το οποίου θα λειτουργήσουν οι δορυφόροι και δεν φαίνεται να είναι πρόθυμη να επιλύσει το ζήτημα αυτό. Ο κύριος Σταχανή είπε ότι συνεχίζεται ο διάλογος με την Κίνα και ο πρόεδρος Βαρόσο έστειλε επιστολή στην Κίνα και παραδέχτηκε ότι υπάρχουν προβλήματα αναρμόνισης. Και αναρωτιέμαι τι πιστεύει ο κύριος Ρεμέκο ότι θα πρέπει να κάνουμε αν καταληξούμε σε πολιτικό αδιέξοδο γιατί α, τελικά αυτή τη στιγμή πρέπει να διαβάζουμε ε, ουσιαστικά κάτω από τις γραμμές και και το θέμα του κόστους. Η Κομισιόν παραδέχτηκε ότι το συνεχιζόμενο καθαρό κόστος θα είναι 500 ε, εκατομμύρια ευρώ το χρόνο και ε, φαίνεται να είμαστε σε πολύ δύσκολη θέση σε ό,τι αφορά τη χρηματοδότηση. Ήδη έχουμε χρησιμοποιήσει πάνω κάτω τα κονδύλια που έχουν εκτομιευτεί για να ε, ε, χρηματοδοτήσουμε το σύστημα στο στάδιο της, ε, της έγκρισης. Επομένως, τι πρόκειται να κάνουμε αν ανακαλύψουμε ότι το κόστος του Γαλιλαίου τελικά ξεφεύγει από τον ελεγχό μας. Θα ήθελα να ακούσω πολύ ενδιαφέρον την άποψη του κύριου Ρέμεκ Δηλαδή πότε τελικά πρέπει να θέσουμε τέρμα στη διαδικασία αυτή. Danke sehr, Kollegin Herzog. Συνάδελφος κυρία Herzog. Elnök úr, szeretnék csatlakozni az előttem szólókhoz az előző európai parlamenti ciklusban. Αγαπητοί συνάδελφοι, κατά την τελευταία ε, θητεία Όλες οι επιτροπές στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και όλα τα πολιτικά κόμματα ε, κατέβαλαν κάθε δυνατή προσπάθεια έτσι ώστε να διατηρηθεί το πρόγραμμα Γαλιλαίος και να ενταχθεί στον Ευρωπαϊκό Προπολογισμό. Είναι ένα ιδιαίτερα σημαντικό ε, πρόγραμμα για μας και είμαστε πεπισμένοι ότι συνεπάγεται πάρα πολλά ωφέλη για τους Ευρωπαίους πολίτες. Είναι όμως εξίσου σημαντικό να μην εκτροχιαστεί το κόστος. Γι' αυτό λοιπόν ε, πρέπει στην ενδιάμεση έκθεση να αναφέρουμε με σαφήνεια ότι δεν πρέπει να υπάρξουν ε, απρόβλεπτοι κίνδυνοι, να μην χάσουμε το χρόνο, αλλά μην ξεχνάμε ότι πρέπει να υπάρξουν και πολλές θυσίες αναγκαστήκαμε και υπήρξαν θυσίες. Αναγκαστήκαμε να απαρατηθούμε από πολλά ερευνητικά υποπρογράμματα για να διατηρηθεί το πρόγραμμα Γαλιλαίος. Είναι σημαντικό ε, να έχουμε υποσχέσεις και ανάληψη ευθυνών, αλλά να παραμένουμε και προσγειωμένοι. Ας σκεφτούμε το πρόγραμμα ITER ή άλλα προγράμματα, στρατηγικές επενδύσεις ε, στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αν λοιπόν θέλουμε να διαβιβάσουμε ή αν διαβιβάσουμε τελικά στους Ευρωπαίους πολίτες το μήνυμα ότι δεν είμαστε αξιόπιστοι, τότε και οι πολίτες δεν θα εμπιστεύονται την έρευνα και την ανάπτυξη, παρότι αυτή θεωρείται πολύ σημαντική για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Για μένα είναι πολύ σημαντικό η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να συνεργαστεί με την Επιτροπή Κοκομπύ και με εμά ε, έτσι ώστε να μπορέσουμε να βελτιώσουμε την εικόνα μα κυρίω την εμπιστοσύνη μα απέναντι στους ε, Ευρωπαίους πολίτες. Ο κύριος Λάμπερτ. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Θα ήθελα να κρατήσω λίγο κάποιε ανησυχίες. Ήταν ε, καλή αρχικά η πρωτοβουλία του Γαλιλαίου, γιατί θέλαμε τελικά να έχει μερίδιο ε, η Ευρώπη σε μια υπηρεσία που παρήχαν μόνο οι Ηνωμένες Πολιτείες ε, και υποστηρίξαμε. Τώρα όμως βρισκόμαστε σε μια δύσκολη κατάσταση, τουλάχιστον αυτή είναι η γνώμη μας. Λόγω δημοσιονομικών αιτιών καταλήξαμε σε αυτό το σύστημα, το οποίο τελικά δεν έχει και πολύ μεγάλη αξία σε σχέση με τις υπηρεσίες που διατίθεται σήμερα. Δηλαδή το να έχουμε ένα ακόμα παγκόσμιο σύστημα ραδιοπλοήγησης δεν έχει κανένα νόημα, εκτός αν υπάρξει κρίση με τις Ηνωμένε Πολιτείε. Και είτε πρέπει να διασφαλίσουμε ότι ο Γαλιλαίο παρέχει υπηρεσίε που δεν διατίθενται σήμερα ή εφαρμογές που δεν είναι διαθέσιμες σήμερα και τότε θα έχει προσθέμενη αξία βεβαίω, αλλά αυτό σημαίνει ότι θα μπορεί να λειτουργεί πλήρω και κανονικά ή τελικά θα έλθουμε αργά σε μία αγορά η οποία θα έχει ξοδέψει πολύ, πολλά χρήματα για ένα σύστημα που τελικά δεν έχει ε, αξία ιδιαίτερη. Αυτή είναι η κατάσταση. Πρέπει να δούμε ποιες είναι οι δυνατότητές μας. Ε, γιατί, γιατί κάθε ευρώ που ξοδεύουμε θα μπορούσαμε να το ξοδέψουμε για κάτι άλλο και όχι για αυτό το σύστημα. Και αυτό που περιμένουν οι πολίτες από εμά είναι να εξετάσουμε στενά τι γίνεται με τον Γαλιλαίο και να πιστούμε πως ό,τι και να κάνουμε έχει προσθέμενη αξία. Δεν έχω τις απαντήσεις στο στάδιο αυτό. Αλλά νομίζω ότι δεν πρέπει να ξεφεύγουμε από τα δύσκολα ερωτήματα σε αυτή την ενδιάμεση αναθεώρηση ακόμη και αν οι απαντήσεις ε, μας ε, κάνουν να φαινόμαστε κάπως σκεπτικιστές. Ε, έχουμε καθυστερήσει, είχαμε κάνει διάφορες επιλογές που δεν μας οδήγησαν πουθενά και τελικά καταλήγουμε σε μια κατάσταση που δεν είναι ικανοποιητική. Έτσι λοιπόν θα ήθελα να έχουμε συζήτηση εις για το θέμα αυτό, ακόμη και αν αυτό σημαίνει ότι θα βγούμε κάπως από τα πλαίσια. Ευχαριστώ. Θα ρωτήσω αν θέλει η Κομισιόν το λόγο. Κύριος Φερχόφ ή ποιος θέλει το λόγο. Παρακαλώ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ κυρίε και κύριοι. Καταρχήν ευχαριστήσω τον κύριο Ρένακ ε, για την πρωτοβουλία να συντάξει έκθεση για το θέμα αυτό. Η επόμενη φάση, το επόμενο στάδιο του Γκαλιλαίου και το έγνωση είναι πάρα πολύ σημαντικές. Όπως ε, είπατε, είναι ένα πολύπλοκο πρόβλημα, είναι πολύ μεγάλου μεγέθους ε, και πρώτη φορά ε, άμεσα αναλαμβάνουν τη διαχείριση τα όργανα και θα πρέπει να λειτουργήσουμε με ένα πολύ συντονισμένο τρόπο. Να πω δύο λόγια για το τι έχουμε κατά νου εμείς ε, και ίσως να μπορέσω και να δώσω και κάποιες απαντήσεις ε, στα σχόλια που ακούστηκαν από τα μέλη. Καταρχήν, συμφωνία με το Συμβούλιο και το Κοινοβούλιο ήταν ότι η Κομισιόν θα ξεκινούσε ε, με μία συνεισφορά στο Γαλιλαίο και θα έθετε παράλληλα σε λειτουργία το έγνος και θα υπήρχε και μία συζήτηση παράλληλα με το πώς θα προχωρήσουμε με το σύστημα μετά από το 2013. Ξέρετε ότι μας ζητήθηκε να παρουσιάσουμε φέτος προτάσεις. Ολοκληρώσαμε σχεδόν ένα χρόνο μελετών εις βάθος για το τι πρέπει να γίνει στο μέλλον και προβλέπουμε να παρουσιάσουμε τις προτάσεις μας τον επόμενο μήνα. Είναι ε, επίγουσες οι προτάσεις αυτές κατά κάποιο τρόπο. Γιατί, τι πρέπει να κάνουμε, να έχουμε μια πολιτική συμφωνία μεταξύ Συμβουλίου και Κοινοβουλίου και Κομισιόν για το πώς θα προχωρήσουμε. Αυτή η πολιτική συμφωνία πιθανότατα πρέπει να μεταφραστεί σε ένα κανονισμό, δηλαδή πρέπει να προταθεί επίσημα και να ε, υπάρξει θεσμική συζήτηση και συμφωνία και στη συνέχεια όποιες διευθετήσεις, ε, σε όποιες τη συμφωνήσουμε θα πρέπει να τεθούν σε εφαρμογή και όλα αυτά θα πρέπει να λειτουργούν στις αρχές του 2014. Δηλαδή δεν έχουμε και πολύ χρόνο στη διάθεσή μα, μόνο λίγα χρόνια. Και φυσικά για ένα τέτοιο σύστημα με το επιχειρησιακό κόστος, το λειτουργικό κόστος που έχει, δεν θα ήταν καλό να έχουμε και ούτε στη διαχείριση ούτε στη χρηματοδότηση από το 2013 και μετά τα θέματα που θίξατε. Να σας δώσω κάποιες απαντήσεις. Ε, ποιος θα διαχειριστεί το σύστημα, πώς θα χρηματοδοτήσουμε ε, τη συντήρηση, την αναβαθμίση του συστήματος, ποια θα είναι η συμμετοχή του δημοσίου τομέα, τι αναμένουμε από τον ιδιωτικό και πώς τα συμφέροντα της Ένωσης ε, θα διασφαλιστούν ποιο είναι το νομικό πλαίσιο που απαιτείται ε, για τη χρησιμοποίηση από τους ε, χρήστες. Ε, κοιτάξτε, αν και το σύστημα είναι ακριβό, το οικονομικό ενδιαφέρον έγκυται στις εφαρμογές. Επομένως, πρέπει να διασφαλίσουμε ότι θα λειτουργούν τα δίκτυα. Έχω πει κάποιες φορές, δεν μπορούμε μόνο να συστήσουμε ένα δίκτυο κινητών ε, στα πλαίσια της υποδομής, ε, δηλαδή ως υποδομή χωρίς να κάνουμε κάτι για τους χρήστες, να μην δημιουργήσουμε διεπαφές με τους χρήστες, έτσι ώστε να αρχίσει να χρησιμοποιείται η υποδομή. Τους επόμενους μήνες, όπως σας είπα, θα προωθήσουμε τις προτάσεις μας. Οι προτάσεις μας θα εξετάσουν τι έχει γίνει τα τελευταία δύο έτη που βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή και θα απαντούν και στις μελλοντικές προκλήσεις. Να πω κάτι για το μέλλον. Θα εξετάσουμε το μακροπρόθεσμο μέλλον, γιατί εμείς θέλουμε σταθερότητα για τα προγράμματα για τις επόμενες δεκαετίες. Φυσικά πρέπει να δούμε τι πρέπει να γίνει με το δημοσιονομικό πλαίσιο από το 2013 έως το 2020, αλλά κατανοείται ότι η σταθερότητα ενό τέτοιου επιχειρησιακού προγράμματος πρέπει να διασφαλιστεί μακροπρόθεσμα και οι χρήστες δεν θα επενδύσουν ε, σε εξοπλισμό έρευνας και ανάπτυξης και εφαρμογέ αν δεν υπάρχει μια λογική εγγύηση ότι το σύστημα μακροπρόθεσμα θα λειτουργεί. Έτσι λοιπόν, ανυπομονούμε να συνεργαστούμε με τον κύριο ρεμέ και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για να εξεύρουμε μια κοινή προσέγγιση και να συζητήσουμε όλα αυτά τα θέματα. Να πω και δύο λόγια για το που βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή. Χθε το βράδυ υπεγράφηκαν συμβάσει ε, ε, με ε, τη βιομηχανία για 14 δορυφόρου για υπηρεσίε στήριξη συστήματο 1,1 δι. Τώρα έχουμε συμβάσεις που ετοιμάζονται για το υπόλοιπο, το του συστήματος κοντά στο 1 δισεκατομμύριο για φέτος επίσης και γνωρίζετε από όσα είπε ο Επίτροπος Ταγιάννη δεν αρκεί ο προπολογισμό για να καλύψουμε όλο το σύστημα. Όμως το σημαντικό είναι ότι τώρα έχουμε ε, δεσμευτεί συμβατικά, έχουμε δέσμευση για την ημερομηνία παράδοσης και έναρξης. Το σύστημα θα περιλαμβάνει 18 δορυφόρους. Έχουμε ήδη του 4 υποκατασκευή, είναι του 14 που παραγγείλαμε. Θα έχουμε λοιπόν ένα σύνολο 18 δορυφόρων, ε, θα υπάρχουν το 2014 και θα μπορέσουμε να παράσχουμε τρεις υπηρεσίες, ανοιχτή υπηρεσία Open Service που ισοδυναμεί με την υπηρεσία GPS που χρησιμοποιούμε σήμερα και προσφέρουν η Είναι σημαντικό να πούμε ότι είναι συμβατή αυτή η υπηρεσία με την υπηρεσία GPS και, και με μελλοντικά εργαλεία, στις μελλοντικές συσκευέ δεν θα βλέπετε διαφορές. Ε, έτσι λοιπόν θα βλέπουν οι χρήστες πολύ περισσότερους δορυφόρους από τους 18 δορυφόρους Γαλιλαίο. Αυτό είναι σημαντικό γιατί αυτό αυξάνει σημαντικά τη διαθεσιμότητα ε, συνδυασμένου του Γαλιλαίου και του GPS έτσι λοιπόν αυτό αποτελεί σημαντική πρόδρο. Η άλλη υπηρεσία που θα περάσουμε το 2014 είναι μια υπηρεσία έρευνας και διάσωσης. Ε, τώρα ε, τα σημερινά συστήματα πλοήγησης ε, δεν προσφέρουν μια τέτοια υπηρεσία. Μόνο η Ευρωπαϊκή Ένωση θα προσφέρει μια τέτοια υπηρεσία στο μέλλον. Είναι πολύ σημαντική υπηρεσία. Συνεργαζόμαστε πολύ στενά με τη σχετική κοινότητα για να θέσουμε σε εφαρμογή αυτή την υπηρεσία. Και η τρίτη υπηρεσία που θα αρχίσουμε να παράσχουμε είναι PRS, είναι η δημόσια ρυθμισμένη υπηρεσία που ε, θα ε, παράσχεται στα ίδια τα κράτη-μέλη και σε όσους έχουν λάβει άδεια από τα κράτη-μέλη. Οι άλλες δύο υπηρεσίες που προβλέπονται είναι η ασφάλεια της ζωής και η εμπορική υπηρεσία. Ε, θα μπορέσουμε να τις περάσουμε το 2014. Μάλλον από το 2014 θα μπορούμε να έχουμε επιδείξεις αρχικές αυτών των υπηρεσιών, αλλά θα πρέπει να έχει τεθεί σε εφαρμογή, να λειτουργεί το σύνολο των δορυφόρων για να παρασκευθούν αυτές οι υπηρεσίες. Όπως είπε και ο Επίτροπος, ε, είναι κάπως ε, πολύπλοκο το δημοσιονομικό θέμα αυτή τη στιγμή, πρέπει να αντιμετωπίσουμε δύο τινά: Το κόστος ε, για το στάδιο IOV ε, που διαχειρίζεται ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Διαστήματος ε, και από ό,τι φαίνεται είναι ανώτερο το κόστος από αυτό που περιμένουμε. Έχουμε 500 ε, εκατομμύρια προ το κόστο και έχουμε τα κράτη-μέλη που δεν μπόρεσαν στον ΕΟΔ να το χρηματοδοτήσουν και μα ζήτησαν να βρεθούν άλλα κονδύλια το κάναμε αυτό γιατί ήταν αναπόφευκτη η απόφαση. Αν δεν την είχαμε λάβει, τότε το στάδιο Β θα είχε σταματήσει και το σύστημα δεν θα υπήρχε. Η άλλη πραγματικότητα που πρέπει να αντιμετωπίσουμε είναι οι τιμές ε, για τους εκτοξευτές παγκοσμίως. έχουν ανέβει 60 ως 80% ε, τα τελευταία δύο έτη και αυτό μας ε, προκαλεί ένα επιπρόσθετο κόστος 500 εκατομμυρία ευρώ. Τώρα ε, για τα υπόλοιπα είμαστε στα επίπεδα που είχαμε εκτιμήσει, έτσι λοιπόν δεν έχει αυξηθεί τόσο πολύ το κόστος, αλλά υπάρχουν κάποιοι εξωτερικοί παράγοντες που δεν έχουμε προβλέψει, που δεν είχαμε προβλέψει. Ανυμονούμε, Πρόεδρε, για τη διεξαγωγή αυτής της συζήτησης επιθυμείτε και όπω και στο παρελθόν ελπίζουμε να μπορέσουμε να ε, ευθυγραμμιστούμε το Κοινοβούλιο και να συμφωνήσουμε για το πώς θα προχωρήσουμε. Ευχαριστώ. Εγώ σας ευχαριστώ. Θέλετε ξανά το λόγο, παρακαλώ. Ναι, σας ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θα είμαι πάρα πολύ σύντομος, γιατί ε, μου υπευλήθησαν κάποιες ερωτήσεις. Η συζήτηση μου επιβεβαίωσε ότι πρόκειται για ένα πολύπλοκο πρόγραμμα. Δεν πρόκειται μια έκθεση πρωτοβουλίας απλώς. Ταυτόχρονα θα ήθελα να ευχαριστήσω την Κομισιόν. Αν θέλετε να δώσω τις απαντήσεις σε όλες τις ερωτήσεις που ε, ε υποβλήθησαν, δεν θα έπρεπε να είμαι στο Κοινοβουλίο, θα έπρεπε να είμαι κάπου αλλού, μου φαίνεται, αν ήμουν τόσο υπερογνώμονας. Όσον αφορά τις ερωτήσεις ε, της κυρίας έχω να πω ότι και εγώ όσα ξέρετε τους ξέρω κι εγώ. Τα προβλήματα σε σχέση με τον Καλλιλέο υπήρχαν πράγματι, πολλά προβλήματα μάλιστα. Στην αρχή υπήρχε από την Αμερική έντονη πίεση να μην χρησιμοποιηθεί αυτό το σύστημα στην Ευρώπη. Παρ' όλα αυτά με τις διαπραγματεύσεις πετύχαμε να επιβάλλουμε αυτό το σύστημα. Και ο παραλληλισμός των συστημάτων είναι επίσης ενδιαφέρον γιατί δεν θα πρέπει ο τελικός χρήστης να πρέπει να ασχολείται με το ποιον δορυφόρο με ποιον δορυφόρο επικοινωνεί αυτή τη στιγμή. Για την Κίνα τώρα, ο κύριος Μπαρόσο στράφηκε προς την Κίνα, προς την κινέζικη ηγεσία δηλαδή, και θα πρέπει να ακολουθηθεί εκεί η διπλωματική οδός. Όσον αφορά όμως πολλά τεχνικά σχέδια, βλέπουμε ότι υπάρχουν και ε, εναλλακτικές τεχνικές λύσεις. Δεν θέλω να επισέλθω σε όλες τις λεπτομέρειες. Κατά τη γνώμη μου όμως, τα προβλήματα μπορούν να επιληθούν. Την απάντηση θα τη δούμε βάσει των αποτελεσμάτων των διαπραγματεύσεων. Τώρα, όσον αφορά το οικονομικό θέμα, την απάντηση στην έδωσε ήδη ο πρόσωπος της Κομισιόν. Εγώ χαίρομαι για τη συνεργασία, για τις τέτοιες καταστάσεις όπου υπάρχουν κάποιες αμφιβολίες και όπου υπάρχουν απόψεις από διαφορετικές ε, πλευρές έχουμε ταυτόχρονα την ευκαιρία να πετύχουμε πολύ καλά αποτελέσματα. Εξακολουθώ να είμαι πεπισμένος ότι πραγματικά αξίζει η Ευρώπη αυτό το πρόγραμμα. Γιατί, Γιατί η Ευρώπη μέχρι στιγμής ήταν ένα πάρα πολύ καλό παράδειγμα ότι μπορούσε με σχετικά λίγα χρήματα να πετύχει να ευθυγραμμαστεί με τις μεγάλες δυνάμεις όσον αφορά την, το διάστημα. Τον αντίον μάλιστα έχει ένα πλεονέκτημα γιατί δεν ε, ζητά να καθιδρύσει ένα στρατιωτικό ε, σύστημα. Έχει ένα σύστημα που έχει μόνο στόχους ειρηνικούς, πολιτικούς. Αυτό είναι ε, πραγματικά πολύ χαρακτηριστικό γιατί στη ΣΥΠΑ έχουν φτάσει σε ένα σημείο όπου το αρχικά στρατιωτικό σύστημα μπορεί να χρησιμοποιηθεί και για μη στρατιωτικούς σκοπούς. Και στην Κίνα θα υπάρχει κάτι παρόμοιο. Γιατί και η Κίνα θα είναι προσεχώς ε, μία από τις μελλοντικέ μεγάλες δυνάμεις. Θέλουμε να είμαστε ανεξάρτητοι. Δεν θα εξαρτηθούμε από αυτές τις υπηρεσίες. Κατά τη γνώμη μου λοιπόν αυτό το σύστημα είναι πάρα πολύ σημαντικό. Ευχαριστώ κύριε Γιάννη ε, Ρέμεκ λέει ο πρόεδρος. Ε, ολοκληρώνονται εδώ οι διαπραγματεύσεις για σήμερα. Ξανατονίζω παρακαλώ, προσπαθήσουμε να τηρήσουμε το 20 λεπτά για κάθε σημείο της ημερησίας διάταξης, για αλλιώς δεν θα προφτάσουμε όλα. Έχουμε ήδη περίπου μισή ώρα καθυστέρηση. Τι να κάνω κι εγώ. Όλοι πρέπει να βοηθήσετε. Το επόμενο σημείο. Αηφόρο μέλλον για τις μεταφορές. Ο συνάδελφος Κάντσιαν έχει το λόγο. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Ε, το μέλλον, το αηφόρο μέλλον για τις μεταφορές, κατά την άποψή μου, είναι ένα σημαντικό θέμα, το οποίο κατά την αμέσως επόμενη περίοδο θα μας απασχολήσει. Ε, το 2001 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκνε τη Λευκή Βίβλο για το μέλλον των μεταφορών ε, που κάλυπτε ε, το χρονικό διάστημα μέχρι το 2010 <clears throat> και εντωμεταξύ το 2006 αναθεωρήθηκε. Τώρα λοιπόν έχει φτάσει η στιγμή που θα κατατεθεί η νέα Λευκή Βίβλος και βεβαίως ε, όλα αυτά τα οποία ακολουθούν κατά κανόνα ως εκ τούτου εγώ θεωρώ ότι η Επιτροπή αυτή θα πρέπει απαρέγκλιτα να ε, δείξει κάποιο σκεπτικό, να παρουσιάσει κάποια επιχειρηματολογία ολοκληρωμένη μάλιστα, για να αντιμετωπίσουμε το θέμα με σοβαρότητα. Ο στόχος λοιπόν της Λευκής Βίβλου 2010 είναι η υλοποίηση ενός συστήματος μεταφορών, ε, το οποίο θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη του τις οικονομικές ανάγκες, μα κυρίως ε, τις ε, κοινωνικές και περιβαλλοντικές της κοινωνίας. Και θεωρώ ότι εδώ το καθοριστικό σημείο είναι η ένταξη των διαφόρων μέσων μεταφοράς, η διαλειτουργικότητα, η χρήση της νέας τεχνολογίας, της επικοινωνίας, η περιβαλλοντική αηφορία και επίσης και η ανταγωνιστικότητα των υπηρεσιών και των ευρωπαϊκών τεχνολογιών στην παγκόσμια αγορά. Τα προγραμματικά μέσα που διατίθενται είναι οι πολιτικές μέσω των οποίων όλοι οι στόχοι αυτοί μπορούν να υλοποιηθούν αλλά επιμένω στην ε, ένταξη των υποδομών στη διατροπικότητα. Η ανάπτυξη των πράσινων τεχνολογιών, την δημόσια και ιδιωτική οικονομική υποστήριξη μέσω των ΣΔΙΤ, υποστήριξη της έρευνας ε, και ενημέρωση των πολιτών. Οι προκλήσεις για το μέλλον ε, είναι εξή. Πρέπει να λάβουμε ε, υπόψη ότι αυξάνονται συνεχώς με ηλικία. Έχουμε γύρανση λοιπόν του πληθυσμού και οι μεταναστευτικές ε, ροές θα φέρουν περισσότερους εργαζόμενους και επιβάτες στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Ένωση πρέπει να επιδιώξει τους στόχους της περιβαλλοντικής αποδοτικότητας. Πρέπει να λάβουμε υπόψη την εξάντληση των ορυκτών καυσίμων και πρέπει να επικεντρωθούμε στον ενεργειακό ανεφοδιασμό. Πρέπει να λάβουμε υπόψη στις δημογραφικές τάσεις στις πόλεις, στα αστικά κέντρα και η παγκοσμιοποίηση μας επιβάλλει να εξετάσουμε τις διαστάσεις όχι μόνο στο εσωτερικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης αλλά και τη σύνδεση προς ε, το εξωτερικό και προς τις τρίτες χώρες. το οποίο θα ήθελα να επιστήσω την προσοχή σας αφορά δύο πτυχές. Ένα που αφορά τη βιομηχανία και την μόλυνση και την εξοικονόμηση ενέργειας που παρά τις προσπάθειες που έχουν υλοποιηθεί γνωρίζουμε ότι πρέπει να επιμείνουμε στην εφαρμογή τεχνολογιών που να μας βοηθούν να μειώσουμε την κατανάλωση ε, καυσίμων και τις βλαβερές εκπομπές η χρήση των μέσων ε, μεταφοράς αυξάνεται συνεχώς και αυξάνεται η κυκλοφορία στους δρόμους. Αυτό αποτελεί ε, αντικείμενο διεθνών συμφωνιών και θα πρέπει να εντάξουμε σε αυτές τους διάφορους τρόπους μεταφοράς και να προβλέψουμε την εισδοκεύση των ε, εξωτερικών πόρων και να ευνοήσουμε το πέρασμα σε μέσα που μολύνουν λιγότερο. Δεύτερη πτυχή, σε ό,τι αφορά την τεχνολογία της ενημέρωσης ε, που έχει να κάνει με τα μέσα μεταφοράς, εφαρμογή αυτής της τεχνολογίας πληροφοριών ε, και επικοινωνιών για τις ε, ροές, τις μεταφορές. Θα μας επιτρέψει να ελέγξουμε και να διαχειριστούμε καλύτερα την κινητικότητα. Αυτό θα επιφέρει πλεονεκτήματα και στη μεταφορά των επιβατών αλλά και των εμπορευμάτων έτσι ώστε να μειωθεί η συμφόρηση και να υπάρχει μεγαλύτερη ασφάλεια. Τέλος, τα προγράμματα ε, ε μέσω δορυφόρων που συζητήσαμε ακριβώ πριν μα επιτρέπουν την συλλογή και διαχείριση πληροφοριών σε σχέση με την κυκλοφορία και με όλα τα προγράμματα που αναπτύσσουν αυτά τα έξυπνα συστήματα μεταφορών που πρέπει να στηριχθούν και να χρηματοδοτηθούν και πρέπει λοιπόν να δοθούν κίνητρα στην έρευνα στους τομείς αυτούς. Ορίστε πρόεδρε και συνάδελφοι, εγώ προσπάθησα να προβώ σε μία σύνθεση, όμως για λόγους ε, χώρου και χρόνου δεν μπόρεσα να αναπτύξω περισσότερο το θέμα ούτε στην ε, πρότασή μου. Θα ακούσω λοιπόν ε, τους συναδέλφους ε, και εγώ ίδιος θα αναπτύξω καλύτερα την πρότασή μου με τροπολογίες. Ε, έχουμε την εκδοχή σε όλες τις γλώσσες ε, στις 13 ε, Ιανουαρίου μέχρι τις 2 Φεβρουαρίου έχουμε την προθεσμία για τις τροπολογίες. Θα προσπαθήσω να τις λάβω υπόψη και θα προσπαθήσω να καταλάβω ποια είναι τα επιπρόσθετα επιχειρήματα που μπορούν να συνεισφέρουν οι συνάδελφοι λαμβάνοντας υπόψη το θέμα αυτό, όπως σας είπα στην αρχή, είναι σοβαρό, σημαντικό και θα αποτελέσει αντικείμενο της στρατηγική ε, της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το 2020. Ευχαριστώ. Thompson. Ευχαριστώ, συνάδελφο Τόμψον. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Χαιρετίζω το σχέδιο της έκθεσης της ε, ε, του εισηγητή για την επικείμενη αυτή λευκή βίβλο τη Κομισιόν που είναι τόσο σημαντική και που καθορίζει την πολιτική μεταφορά για τα επόμενα 10 χρόνια. Η μείωση των εκπομπών των, ε, του θερμοκηπίου είναι πάρα πολύ σημαντικό, όπως επίσης και η μείωση της ε, ηχορύπανσης, ιδίω στις αστικέ περιοχές. Έχουμε διάφορες νέες τεχνολογίες που θα μας βοηθήσουν, αλλά η πρόκληση είναι να επιταχυνθεί η μετάβαση στις νέες αυτές τεχνολογίες ορισμένου θα έλεγαν ότι θα πρέπει να αφήσουμε τα πράγματα στην αγορά και ότι είναι επικίνδυνο να επιλέξουμε εμείς ε, τους νικητές. Εγώ πιστεύω θα πρέπει να κάνουμε ό,τι μπορούμε για να βρούμε ποια είναι τα προβλήματα με τις νέες αυτές τεχνολογίες και να βοηθήσουμε το γλυγορότερο δυνατόν Χωρί να παραβλέπουμε καμία τεχνολογία. Θα πρέπει να μην ξεχνάμε ότι η εισαγωγή κάθε νέα τεχνολογία είναι ακριβή και γι' αυτό χρειαζόμαστε στην αρχή μια χέρα βοηθεία. Και εμείς εδώ στην Επιτροπή μας θα ήταν καλό να προτείνουμε την εξασφάλιση όρων πλαισίου για την προώθηση των ηλεκτρικών ε, οχημάτων που θα μπορέσουν να βοηθήσουν την καλύτερη χρήση ε, της ενέργειας, παραδείγματος χάνει και αιωλικής ενέργειας. Έτσι θα μπορούσαμε να μειώσουμε και τις εκπομπές του θερμοκηπίου και την ηχορύπανση τη φύλη και να αυξήσουμε την αποτελεσματικότερη χρήση ε, της ενέργειας και να μειώσουμε την εξάρτηση από το πετρέλαιο. Θα πρέπει να είμαστε κατά συγκεκριμένοι. Ποια είναι η ε, νομοθεσία που θα πρέπει να εισαχθεί ή να τροποποιηθεί τα επόμενα χρόνια για να είμαι σίγουρη ότι ο τομέας των μεταφορών θα είναι φόρος στο μέλλον και σύμφωνα με την οδηγία. Ευχαριστώ. Εγώ σας ευχαριστώ. Ο κ. Λάνε. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Και εγώ ευχαριστώ τον εισηγητή για το κείμενο που υπέβαλε και θέλω να το συμπληρώσω με δύο σημεία. Η πολιτική μεταφορών, κυρίε και κύριοι, είναι κεντρική σημασία για την βιομηχανία στην Ευρώπη. Για δύο λόγου. Γιατί καταρχήν, χωρί αποτελεσματικέ μεταφορέ, η βιομηχανία μα δεν μπορεί αποτελεσματικά να λειτουργήσει. Και κατά δεύτερον, η βιομηχανία της κινητικότητας είναι ο βασικός τομέας παραγωγής στην Ευρώπη. Αυτοκινητοβιομηχανία, σε δρομική βιομηχανία, ναυπηγική κλπ. Και γι' αυτό εκτός από τα θέματα της ε, μείωσης επιβάρυνσης του περιβάλλοντος θα πρέπει να λάβουν υπόψη μας και αυτές τις δύο πτυχές. Πρώτη πτυχή. Η οργάνωση της μεταφοράς για να μπορέσει να βελτιωθεί η παραγωγική διαδικασία. Εκεί χρειάζεται πράγματι μια ολοκληρωμένη ε, προσέγγιση για τις μεταφορές. Δεν βοηθάει πάρα πολύ αγαπητοί συνάδελφοι εάν αναπτύσσουμε νέες τεχνολογίες με το σύστημα Γαλιλαίο και έτσι έχουμε μια βελτιωμένη δυνατότητα να οργανώσουμε τη δυνατότητα για τα ε, φορτηγά, να απαγορέψουμε όμως τα φορτηγά αυτά να παίρνουν εμπόρευμα από άλλες χώρες εκτός από τη χώρα στην οποία προέρχονται. Αυτό σημαίνει ότι έχουμε περίπου 30% άδειε διαδρομές στην Ευρώπη των φορτηγών αυτών. Και αυτό δεν είχε κανένα νόημα. Για να το αντιμετωπίσουμε όμως θα χρειαστούμε μια ολοκληρωμένη προσέγγιση. Χρειαζόμαστε δηλαδή τον Γαλιλαίο για να είμαστε αποτελεσματικοί. Χρειαζόμαστε όμως και την άση των απαγορεύσεων καμποτάζ. Αυτή είναι λοιπόν η πρώτη μου πρόταση για συμπλήρωση. Να έχουμε πιο ολοκληρωμένη πολιτική στον τομέα των μεταφορών. Μπορεί να γίνει και στον τομέα των ε, εμπνευματικών συνδρομικών μεταφορών. Δεν έχει κανένα νόημα κυρίε και κύριοι ένα ε, ένα τρένο που κινείται από μέσα από διάφορα σύνορα στην Ευρώπη να κινείται με τόσο μικρές ταχύτητες. Η μία πτυχή που σας ανέφερα αφορά την ε, βιομηχανική παραγωγή. Θα πρέπει βέβαια να έχουμε σωστή ε, απόδοση και στο μέλλον θα πρέπει να δούμε πώς οι μεταφορές στο μέλλον, πώς η κινητικότητα στο μέλλον θα οργανωθεί. και θα πρέπει εκεί να περάσουμε την βοηθητική ε, βοηθητική πολιτική για την κινητικότητα. Υπάρχουν διάφορες προσπάθειες όσον αφορά και την έρευνα, αλλά όσον αφορά και πιο συγκεκριμένα σχέδια για να υπάρξει μεγαλύτερη πίεση και να πετύχουμε έτσι μία ευρωπαϊκή αναδιάρθρωση, ούτω ώστε οι θέσει απασχόλησης στον τομέα αυτό να είναι πραγματικά σίγουρες και για το μέλλον. Και κάτι ακόμα, ο Σνάλφας αναφέρθηκε στα ηλεκτρικά ε, οχήματα. Πολλές φορές ε, το πρόβλημα στην εισαγωγή καινοτομιών είναι ότι δεν υπάρχει επαρκής τυποποίηση. Πρέπει να ξέρουμε ποια είναι η δομή που θέλουμε τι πρίζες χρειάζονται. Πραγματικά θα πρέπει η βιομηχανία εδώ να εργαστεί προς την κατεύθυνση αυτή για να έχουμε καλή τυποποίηση για τα καινοτόμα προϊόντα. Σας ευχαριστώ πολύ. Πρόεδρος. Έξι έχουν ζητήσει το λόγο τώρα. Θα σας ήμουν ιδιαίτερα ευγνώμων να προσπαθήσετε πραγματικά να είσαστε κατά δυνατόν σύντομοι. Ο κ. Τσιτσίστερ έχει το λόγο πρώτος. Ο Μπαλτσίτης, συγγνώμη. Θα είμαι σύντομο. Ε, στην έκθεση αυτή αναφέρονται διάφορε από τι προτάσει Κομισιόν και εγώ θα τονίσω διάφορε από αυτέ. Καταρχήν, όσον αφορά το διοξείδιο του άνθρακα, ελέγχθησαν διάφορα, δεν θα επαναλάβω, αλλά η ε, αστιφιλία είναι πάρα πολύ ανησυχητική. Γιατί όσο πάει και περισσότεροι άνθρωποι συγκεντρώνονται στις αστικές περιοχές και θα συγκεντρωθούν ακόμα περισσότερο στο μέλλον και θα πρέπει γι' αυτό με την έκθεση αυτή να στείλουμε κάποια μηνύματα όσον αφορά τη μελλοντική πολιτική τιμών. Παραδείγματο χάρη ένα τέλος ρήπανσης. Παραδείγματο χάρη τα αστικά κέντρα, οι τοπικές αυτοδικήσεις θα πρέπει να σκεφτούν αυτό το θέμα. και θα πρέπει να δούμε ότι τα σχέδια αυτά είναι πάρα πολύ σημαντικά για την ανταγωνιστικότητα των κρατών μελών. Αυτό θα πρέπει να είναι μια προτεραιότητα για το μέλλον. Τα σχέδια αυτά είναι πάρα πολύ σημαντικά και όσον αφορά την ασφάλεια. Έχουμε τον στόχο του στη Λευκή Βίβλου που ήταν για το 2010 και που δεν έχουν επιτευχθεί ακόμα και γι' αυτό θα πρέπει η στρατηγική μας για το μέλλον να είναι τέτοια ούτω ώστε τα κράτη-μέλη να αναλάβουν περισσότερες υποχρεώσεις για την επίτευξη των προβλεπωμένων στόχων. Θα ήθελα επίσης να υποστηρίξω τους στόχους όσον αφορά τα καθαρά μέσα μεταφορών και θα ε, πρέπει να λάβουν υπόψη μας και τις σκέψεις του ε, Πρωθυπουργού Σαμπατέρα ότι τα συστήματα μεταφορών που δημιουργούνται θα πρέπει να είναι πτωχά όσον αφορά τι εκπομπές και να είναι συμβατά με το περιβάλλον. Παραδείγματο χάρη τα ηλεκτρικά οχήματα. Θα πρέπει πάντα να έχουμε κατά νου το μέλλον και τους ανθρώπους στο μέλλον και το πώς οι άνθρωποι μπορούν να αντικαταστήσουν τα μη οικολογικά με οικολογικά οχήματα. Ε, ευχαριστώ, Πρόεδρε. Πολλά καλά ελέγχθησαν. Θα ήθελα να συγχαρώ τον συνάδελφο Γκαντσιάν, τον κ. Χατζημαρκάκη, ε, που δεν μπορεί παρά να είναι κάπως ε, περιοριστικός, γιατί δεν έχει και τόσο πολύ χρόνο. Θα ήθελα να αναφερθώ στον κ. Λάγκερ. Οι μεταφορές είναι το μεγάλο μας ανταγωνιστικό πλεονέκτημα σε όλο τον κόσμο. Γιατί αν ξεκινήσουμε από τις δυνατότητες και δικαίως ο κ. Καντσιάν θέσει το θέμα της τεχνολογίας πληροφορικής ε, και ενημέρωσης ε, στο επίκεντρο, γιατί όσον αφορά τη δυνατότητα δικτύωσης, είμαστε ηγητές σε όλο τον κόσμο. Έχουμε 27 κράτη-μέλη και έχουμε 27 διαφορετικά συστήματα παραδείγματο χάρη σιδηροτροχιών, και δεν μπορούμε αυτό που έχουμε κατά νου να το πραγματοποιήσουμε γιατί υπάρχουν πάρα πολύ, ε, πολλά εθνικά συμφέροντα τα οποία θα πρέπει να ξεπεράσουμε και αυτό θα είναι αυτό που θα πρέπει να επιτύχουμε σαν Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ότι εδώ δηλαδή θα πρέπει να ζητήσουμε πιο έντονα ευρωπαϊκή πτυχή σε όλα αυτά αλλιώς δεν θα πετύχουμε να προωθήσουμε στην αγορά αυτό που έχουμε. Δεν επιτρέπεται ένα φορτηγό που πάει από την Κοπενχάγη στη Μαδρίτη κινείται με μέση ταχύτητα 17 χιλιόμετρων ανά ώρα. Έχουμε καλύτερα συστήματα. Δεν έχουμε κάνει αυτό που θα έπρεπε. Θα πρέπει να ξεπεραστεί. Γιατί όχι, και θα χαρεί ο κύριος Μπιουτικόφερ, αν είχαμε πράσινους διαδρόμους που προβλέπουμε, δηλαδή σχέδια πειραματικά, αλλά στις, στους κεντρικούς άξονες θέματα που έθιξε ο Ζαπατέρο, να προωθήσουμε δηλαδή την ηλεκτρικοποίηση της, ε, των μεταφορών με αηφόρο βέβαια ρεύμα και να έχουμε κεντρικούς άξινες, ε, αηφόρους, πράσινους όπως θέλετε πέσω του και αυτοί θα πρέπει να τους χρηματοδοτήσουμε από τους πόρους που έχουμε. Θα πρέπει η περιφερειακή πολιτική και η πολιτική συνοχή και η πολιτική για την υπεθρό να βασιστεί σε αυτό το κεντρικό θέμα. Δεν μπορούμε να αναφερόμαστε μόνο στο διοξείδιο του άνθρακα. Θα πρέπει να έχουμε σε κέντρο ε, τη συζήτηση και το θέμα τη κινητικότητα. 17 χιλιόμετρα ανά ώρα δεν είναι και τόσο θαυμάσιο. Θα πρέπει να το έχουμε αυτό υπόψη μα. Το Ζάφο Λάγκα αναφέρθηκε σε κάτι πάρα πολύ βασικό και δεν μπορώ παρά να το ξανατονίσω. Να καλέσω την Κομισιόν να θέσει πρότυπα δεν μας ωφελούν τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα που έχει ο, ε, προωθήσει ο Σαπατέρα στην Ισπανία, τα οποία όμως δεν μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε στο Βερολίνο. Θα πρέπει να υπάρχει τυποποίηση και επίση η μορφή ενέργειας θα πρέπει να προωθηθεί. Αυτά τα πρότυπα, αυτά, αυτή την τυποποίηση θα πρέπει να την κάνει η Κομισιόν τώρα. Η Κομισιόν πολλές φορές περιμένει πολύ την βιομηχανία. Η βιομηχανία έχει προχωρήσει όμως και αυτή τη στιγμή ε, προσπαθεί να ε, δηλώσει, να καταθέσει κάποια πρότυπα, αλλά θα πρέπει να γίνει αυτό. Αν δεν υπάρχει τυποποίηση, δεν θα μπορέσουμε να εκμεταλλευτούμε τις δυνατότητε του ανταγωνισμού που έχουμε. Ευχαριστώ. Άλλοι τέσσερι και άλλε τρει εκθέσει και σε θα έρθει ο Υπουργό. Παρακαλώ. Ε, θα ήθελα να είμαι Σύντομος, ε, κοιτάξτε το μυστικό της, του εξορθολογισμού στις ευρωπαϊκές μεταφορές αφορά την επιμελητία. Ε, Παραδείγματος χάρη ε, δεν είναι δυνατόν ε, οι μεταφορές με φορτηγά μάλλον τα φορτηγά να κινούνται στην Ευρώπη κατά τόν 1 τρίτον άδεια. Και πώς είναι δυνατόν να συμβαίνει κάτι τέτοιο. Το βασικό αίτιο είναι ότι παλαιότερα υπήρχε η απαγόρευση του καμποτάζ και έτσι λοιπόν πριν τελικά κατορθώσουμε τους κατασκευαστές να τους αναγκάσουμε να μεριμνήσουν για την μείωση των ρηπογόνων ουσιών, θα πρέπει να χρησιμοποιήσουμε τα μέτρα που έχουμε στη διάθεσή μας και πρέπει να εστιάσουμε την προσοχή μας στην απαγόρευση του καμποτάζ στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Θα ήθελα να συγχαρώ τον κύριο Κανσιάν για το έργο του και να επιμείνω στο ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν επενδύει τα μάλλα στο Ευρωπαϊκό Δίκτυο Μεταφορών. Αυτό είναι δραματικό πρόβλημα. Είναι οι ανάγκες μεταξύ 600 και εκατομμυρίων και ενός δισεκατομμυρίου. Δεν επενδύουμε τόσο πολλά. Έτσι λοιπόν ε, η ερώτησή μου είναι σήμερα τι επικρατεία θέλουμε και, έχουμε, ε, μια, και πρέπει να έχουμε μια πολιτική χωροταξία έτσι ώστε όλοι να εξυπηρετώνται από ε, τις μεταφορές και να ενώνουμε τα αστικά κέντρα με την επαρχία και να μην επικεντρώνουμε τις επενδύσεις μας στα αστικά κέντρα γιατί Όσο αντιμετωπίζουμε τα προβλήματα στις πόλεις, τόσο περισσότερο αυξάνουμε τη μόλυνση και οθούμε και τους πολίτες προσταστικά τα κέντρα. Έτσι λοιπόν αυτά τα στοιχεία των μεταφορών και της κινητικότητας είναι πάρα πολύ σημαντικά. Πρέπει να επενδύσουμε στη διασύνδεση των δικτύων μεταξύ των κρατών μελών. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Επόμενη ομιλήτρια. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Κοιτάξτε, οι δικές μου παρατηρήσει αφορούν ε, στις ε, προτάσει που κατατέθηκαν. Ε, στο σημείο υπαριθμών 6 ε, αναφέρονται τα πάντα, γίνεται λόγος για την ασφάλεια, για την επιμελητία, για τη ρήπανση, ε, για την έγκαιρη ολοκλήρωση των προγραμμάτων TET και επίσης και για την χρηματοδότηση των ε, μελλοντικών ε, καθαρών μεταφορών. Εγώ έχω να καταθέσω μία πρόταση. Πρώτον, θα πρέπει να αποδοθεί μεγαλύτερη σημασία στο μέλλον ε, των διαλειτουργικών προγραμμάτων και αυτό θα πρέπει να είναι ένα θέμα ε, που πρέπει να απασχολήσουν αδέλφους. Αυτή τη στιγμή, όπως αναφέρθηκε, δεν υπάρχουν αρκετές επενδύσεις και ε, ικανοποιητικός προγραμματισμός. Ε, να υπάρχουν ξεχωριστά προγράμματα. Αυτό πρέπει να υπογραμμιστεί. Η δεύτερη παρατήρησή μου αφορά το εξής. Ε, γίνεται λόγος ε, για την εφαρμογή της ε, ατζέντα της ε, Λισαβόνας. Εγώ, αν μου επιτρέπετε, εδώ θα ήθελα να προσθέσω στην ατζέντα της Λισαβόνας και στην πολιτική γειτονίας, έτσι ώστε η Ευρωπαϊκή Ένωση να συνδεθεί με όμορες χώρες και να μη στηρίζεται μόνο η συνθήκη της Λισαβόνας, αλλά και η πολιτική γειτονία που επίσης είναι σημαντική, γιατί εμείς επιθυμούμε ε, να συνεχίσουμε τις ε, καλές σχέσεις που έχουμε με τους γειτονάς μας, ε, γειτονάς μας, στο πλαίσιο εξωτερικής πολιτικής. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Χανά. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Για να τοποθετηθώ για το σχέδιο γνωμερώτηση τη Επιτροπή μα, είναι καταρχήν πρέπει να δούμε το τηλεκομισιόν ε, τώρα λέμε καταρχήν ότι ε, το άνοιγμα ε, των αγορών μεταφορών έχει οδηγήσει σε πτώση των τιμών και σε καλύτερη διασυνδεσιμότητα όμως δυστυχώς βλέπουμε ότι δεν ισχύουν αυτά γιατί υπάρχει υποβάθμιση του περιβάλλοντος, της ασφάλειας, μειονεκτήματα για τους εργαζομένους όμως βλέπουμε αντίθετα να έχουμε τεράστια κέρδη κέρδη από τις μεγάλες ε, ε, επιχειρήσεις ε, που εξαγοράζουν σαν να μιλάμε εδώ για μονοπόλιο. Αν θέλουμε πραγματικά να κάνουμε την επανάσταση στο εσωτερικό της Ευρώπης πρέπει τελικά να αναλάβουμε δράση αν δεν θέλουμε να καταλήξουμε σε άγονες δράσεις. Εμείς δίνουμε κίνητρα και ενθαρρύνουμε τα κράτη-μέλη να κάνουν διάφορα αλλά δεν υπάρχει τελικά καμία όθηση. Εδώ θέλουμε τελικά να έχουμε τις καλύτερες δυνατές συνθήκες σε ό,τι αφορά το περιβάλλον και την ασφάλεια και το Κοινοβούλιο θα πρέπει να επικεντρωθεί ε, στο θέμα του περιβάλλοντος, θα πρέπει να λάβουμε υπόψη τις ανάγκες των πολιτών, θα πρέπει να έχουμε προϊόντα ε, που θα διανέμονται, θα πρέπει να ε, επενδύουμε στη διατήρηση των υποδομών γιατί ο ευρωπαϊκός πολίτης δεν πρέπει να πληρώνει πάντοτε το κόστος όταν του ζητάμε να συμμετάσχει στην ε, διανομή των κερδών. Ε, πρέπει ε, να σταματήσουμε να δρούμε βάση μόνο συμφερόντων και αν η Ευρώπη δεν προβεί στην ανάπτυξη υποδομών για τις μεταφορές τότε δεν θα προχωρήσουμε ε, να σας αναφέρω και δύο παραδείγματα. Στους σιδηροδρόμους θα πρέπει επιγόντως, θα πρέπει να έχουμε μία ευρωπαϊκή δημόσια επιχείρηση ε, με δημόσιο κεφάλαιο, γιατί αυτό θα μας επιτρέψει να αποφύγουμε τη σημερινή κακοφωνία και θα μας επιτρέψει να υπάρχει πραγματική ε, ολοκλήρωση και διατροπικότητα μεταξύ των διάφορων ειδών τρένων, ΤΖΒ, ε, κτλ. Και θα πρέπει να ε, ε, έχουμε προγράμματα έρευνες για τα καθαρά αεροπλάνα του αύριο. Θα πρέπει να θέσουμε τέλος ε, στη χρήση των ορυκτών καυσίμων στην αεροπλοεία ε, θα πρέπει ουσιαστικά να δημιουργήσουμε ένα ευρωπαϊκή βιομηχανία έναντι των ανταγωνιστών από τη Ρωσία και την ε, Κίνα. Ε, επίσης, δυστυχώς η μόνη επιτυχία που έχουμε είναι το Airbus και μιλάμε για τεχνολογίες που έχουν αναπτυχθεί εδώ και 25 χρόνια και αυτό χάρη στο δημόσιο, στα δημόσια κονδύλια. Ευχαριστούμε πολύ εκ μέρου ε, τη ε, Κομισιόν. Ε, Σανταμάτο, πολύ σύντομα παρακαλώ αν είναι δυνατόν. Θα σας ήμασταν ευγνώμονε, αν μπορούσατε να είστε σύντομο. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Πρόεδρε. Και Ευχαριστούμε επίσης τον εισηγητή για την έκθεσή του, γιατί η έκθεσή του σε μεγάλο βαθμό συμβαδίζει με τη στρατηγική που έχει καταθέσει η Κομισιόν στην ανακοίνωσή της για ένα αηφόρο μέλλον για τις μεταφορές. Και αυτό είναι το πρώτο σημαντικό βήμα ε, στο δρόμο για την προετοιμασία της επόμενης Λευκής Βίβλου, η οποία έχει και θα έχει ως στόχο να βελτιώσει την ε, περιβαλλοντική απόδοση των ε, μεταφορών, των μέσων μεταφοράς, ε, να αποδώσει επίσης ιδιαίτερη σημασία στην έλλειψη πηγών και πρώτων υλών, κάτι που μπορεί να αποτελέσει πρόβλημα για το μέλλον. Ξέρετε ότι ο πρόεδρος κύριος Μπαρόζο παρουσίασε το στόχο που είναι να μην υπάρχουν εκπομπές διοξιδίου του άνθρακα από τις ε, πρώτε λύσει που χρησιμοποιούνται, από τα καύσιμα που χρησιμοποιούνται στις ε, μεταφορές. Αυτό λοιπόν είναι ένας ε, πολύ φιλόδοξος στόχος, ο οποίος προποθέτει την κινητοποίηση πολλών εργαλείων και θεωρώ ότι πάρα πολλά από αυτά που αναφέρθηκαν στη συζήτηση πράγματι ε, έχουν ε, συμπεριληφθεί και θα συμπεριληφθούν στην επόμενη Λευκή Βίβλο. Θα ήθελα λοιπόν να αναφερθώ στην έννοια της ε, διαλειτουργικότητας των μέσων μεταφοράς της τεχνολογίας που θα μας στηρίξει, τεχνολογία τόσο για εναλλακτικά καύσιμα, όσο και για τη συμπερίληψη της ε, πληροφορικής στη διαχείριση της ε, κυκλοφορίας και σε άλλες εφαρμογές. Αναφέρθηκε επίσης η πολιτική τιμολόγηση, το περαιτέρω άνοιγμα της ε, εσωτερικής αγοράς και Όλα αυτά μέσα σε ένα πλαίσιο ολοκληρωμένης προσέγγισης, όπως πολύ σωστά αναφέρθηκε. Γι' αυτό λοιπόν θεωρώ ότι όλα τα σχόλια που έγιναν συμβαδίζουν ε, με αυτά που πιστεύουμε και εμείς. Δεν χρειάζεται να συζητήσουμε περαιτέρω και εμείς ε, προσβλέπουμε στην ε, συμβολή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην επόμενη Λευκή Βίβλο. Πρόεδρο, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ο εισηγητής παρακαλώ. Πρόεδρε, πιστεύω ότι ακούστηκαν σημαντικά σχόλια τα οποία θα τα λάβω υπόψη και φυσικά περιμένω να στείλουν οι συνάδελφοι και γραπτές τροπολογίες ως τις 2 Φεβρουαρίου και ε, θα συνεισφέρω και εγώ με δικές μου πρωτολογίες ε, και θα υποβάλω τη γνωμοδότηση για τελική ψηφοφορία. Σα ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ο εισηγητή λοιπόν είπε ήδη 2 Φεβρουαρίου το μεσημέρι είναι καταληκτική ημερομηνία για την κατάθεση των τροπολογιών. Επόμενο ε, θέμα, τα γεωσκοπικά συστήματα. Να είστε σύντομο, παρακαλώ. Βεβαίω θα προσπαθήσω, Πρόεδρε, ε, κυρίες και κύριοι, αγαπητοί συνάδελφοι, υπάρχουν πάρα πολλές τροπολογίες που έχουν ε, κατατεθεί και τις οποίες εμείς εξετάσαμε. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τους ε, συντάκτες αυτών των τροπολογιών. Σε γενικές γραμμές, στην έκθεση αυτή δεν υπάρχουν έντονα επίμαχα θέματα. Όλες οι πολιτικές ομάδες αναγνώρισαν τη σημασία αυτού του θέματος και καταλήγουν σε ότι πράγματι πρέπει να προχωρήσουμε. Θα ήθελα να αναφερθώ σε ορισμένα σημεία των ε, τροπολογιών. Πρώτον, όσον αφορά ε, την ε, τροπολογία να συμπεριληφθεί σε αυτόν τον κανονισμό και η θάλασσα και η ατμόσφαιρα. Καλό αυτό, γιατί με τρόπο αυτό θα μπορέσουμε να έχουμε καλύτερη διαχείριση καταστροφών. το δεύτερο εδώ ε, πρέπει και εγώ λιγάκι να αυτοδιορθωθώ, δηλαδή ε, κανείς ε, δεν μπορεί να ισχυριστεί ότι δεν κάνει λάθη. Όσον αφορά αυτή την ανοιχτή πρόσβαση στα δεδομένα, πράγματι δεν μπορούμε να μιλάμε για δωρεάν πρόσβαση, αλλά να μιλάμε για ανοιχτή και διαφανή πρόσβαση στα δεδομένα, πράγμα που σημαίνει ότι για την επεξεργασία των δεδομένων προφανώς θα πρέπει να επιβάλλονται τέλη. Και στο μέλλον θα πρέπει να συζητήσουμε γι' αυτό. Ίσως θα πρέπει να έχουμε μια επιστροφή στην απόδοση, return on investment, όπως λέει ο μιλητής. Στο μέλλον να παραμείνουμε ανοιχτοί στο θέμα αυτό. Κατά τα άλλα, υπάρχουν τροπολογίες για την αποφυγή επικαλύψεων ε, στη συγκέντρωση δεδομένων. Υπάρχουν δεδομένα τα οποία έχουν ήδη συγκεντρωθεί ε, πράγματι ε, σωστό και αυτό. Εδώ βέβαια υπάρχουν και διαφορετικές απόψεις ε, όσων την τροπολογία, Πού θα πρέπει δηλαδή αυτό να ενταχθεί στον κανονισμό. Και εδώ θα ήμουν ευγνώμων αν η Κομισιόν μπορούσε να μας κάνει μια επικοδομητική πρόταση πού να θίξουμε αυτήν την επικάλυψη των δεδομένων και πού να κατατεθεί η τροπολογία. Γίνεται λόγος και για το Partners Board. Εδώ υπήρξαν ε, τροπολογίες ε, στην Επιτροπή Προπολογισμών. Δεν είναι κακή αυτή η ιδέα, αλλά θα πρέπει να δούμε ποιος θα μπορούσε να συμπεριληφθεί σε αυτό το είδος σύμπραξης, ας το πούμε έτσι, Partners Board. Ε, ποιος θα συμπεριλαμβάνεται στους παραγωγούς του συστήματος στο μέλλον. Υπάρχουν και κάποιες τροπολογίες που είμαι πάρα πολύ επιφυλακτικός. Παραδείγματος χάνει η πρόταση παράλληλα και πέρα από τις ε, τρεις ε, συστάσεις που υπάρχουν να προσθεθεί και μία ε, τέταρτη. Την άκουσα αυτή την πρόταση αλλά νομίζω ότι είναι πάρα πολύ προχωρημένη αυτή η παρατήρηση το να συμπεριλάβουμε και αυτό. Και τέλος υπάρχει πρόταση της επιστοποίησης των δεδομένων. Εκεί προτείνεται αυτό να γίνεται από την Κομισιόν. Εγώ έχω κάποιες επιφυλάξεις επ' αυτού αλλά η ίδια Κομισιόν πρέπει να μας πει κατά πόσο είναι σε θέση να προσφέρει κάτι τέτοιο. Δεν είναι λάθος η προσέγγιση. Καλή είναι, τα δεδομένα πρέπει να είναι αξιόπιστα και το θέμα που τίθεται μόνο είναι κατά πόσο η Κομισιόν είναι ο κατάλληλος φορέας για να πράξει κάτι τέτοιο. Κατά τα άλλα προτείνω το συντομότερο δυνατόν να ξανασυναντηθούμε σε μια ε, συνάντηση των ε, σκιωδών εισηγητών. Εγώ θα σας ε, καλέσω σε μια τέτοια συνάντηση για να προετοιμάσουμε συμβαστικές προτάσεις, τις οποίε μετά θα συζητήσουμε. Και κατά τα άλλα ε, παραμένει ανοιχτό ένα θέμα, όπως και στην προηγούμενη συζήτηση που έγινε για το πρόγραμμα Γαλιλαίο. Ε, το θέμα της χρηματοδότησης. Εχθές στην Επιτροπή Προϋπολογισμών συζητήθηκε το θέμα της ε, χρηματοδότησης από τους συναδέλφους και εχθές η Κομισιόν διαβεβαίωσε ότι θα μας δώσει έτσι μια γενική εικόνα για το από πού θα πάρει, από ποιους επιμέρους προπολογισμού θα πάρει τα κονδύλια για τα δικά μας τα προγράμματα. Πρέπει λοιπόν να έχουμε έχουμε τις απαραίτητες πληροφορίες και παράλληλα καλό θα ήταν η Κομισιόν να μας διαβεβαιώσει ότι θα αρκέσουν αυτά τα ε, κονδύλια. Γιατί κατά τα άλλα ε, θα πρέπει να καταθέσει τροπολογία να αυξηθούν τα κονδύλια. Και θα χαιρόμουν πάρα πολύ αν επί του θέματος αυτού επικρατούσε σε το στομό των Κατά τα άλλα θεωρώ ότι όλοι από κοινού είμαστε σε θέση και επιθυμούμε η έκθεση αυτή να κλείσει πριν από το καλοκαίρι. Πρόεδρος ε, και εγώ ευχαριστώ. Πρώτος συνάδελφος Νταντ Ευχαριστώ. Πρόεδρε. Εγώ εξέτασα το σύνολο των τροπολογιών ε, που κατατέθηκαν από τους συναδέλφους ε, και μπορώ να πω ότι χέρι συνένεσης ε, η έκθεση. Χαίρομαι που ορισμένοι κατέθεσαν τις ίδιες τροπολογίες που είχα καταθέσει και εγώ αναφέρουμε συγκεκριμένα στη σύσταση αυτού του Partners Board. Ε, άκουσα τα επιχειρήματά σας, ε, κύριε Κλίντε, για τη σύνθεση και για τη λειτουργία ε, του Συμβουλίου αυτού. Νομίζω ότι συμφωνούμε για τη σύσταση αυτού του Συμβουλίου και την καταλληλότητά του. Τώρα, για τα δεδομένα GMS, πρέπει να υπάρχει συντονισμό με το τι υπάρχει σε εθνικό επίπεδο. Υπάρχουν και σχετικέ τροπολογίε, άλλε τροπολογίε που κατατέθηκαν, που είναι ενδιαφέρουσε. Νομίζω ότι για αυτές θα ήταν ενδιαφέρον να συζητηθούν αυτές ε, από όλους τους εισηγητές όμως θα ήθελα να επανέλθω στο δωρεάν χαρακτήρα. Είχαμε συζητήσει το θέμα αυτό την περασμένη φορά για το δωρεάν, τη δωρεάν πρόσβαση στα δεδομένα. Νομίζω ότι υπήρχε η απαρχή κάποια συνένεση σε αυτό, όμως ε, ε κυρία Τυρκάου είχε, θέσει μία, είχε καταθέσει μια τροπολογία για την αρχή της, ε, του δωρεάν χαρακτήρα. Ε, εγώ νομίζω ότι ε, εδώ δεν πρέπει να είμαστε κάθετοι σε σχέση με το θέμα αυτό σήμερα. Στο στάδιο αυτό θα πρέπει να το εξετάσουμε το θέμα, αλλά θα πρέπει να έχουμε οπωσδήποτε ε, την αρχή της ελευθερής πρόσβασης στα δεδομένα GMS. Γι' αυτό έχω καταθέσει την τροπολογία 28 και την τροπολογία 37, γιατί η ελεύθερη πρόσβαση δεν σημαίνει δωρεάν. Είναι η συζήτηση που είχαμε και η αρχή της ελεύθερης πρόσβασης ε, και η αρχή της δωρεάν πρόσβασης όχι, μπορούμε να τη συζητήσουμε, όμως πρέπει να έχουμε την ελεύθερη πρόσβαση στα δεδομένα. Νομίζω ότι στο στάδιο αυτό πρέπει λοιπόν να διαφοροποιήσουμε ε, ξεκάθαρα το θέμα της ελεύθερης πρόσβασης και του δωρεάν χαρακτήρα των δεδομένων. Επίσης νομίζω ότι πρέπει να μην περιορίσουμε τις δυνατότητες του προγράμματος GMS, e το συζητήσαμε αυτό τη τελευταία φορά, ε, έτσι ώστε η αγορά να υιοθετήσει συζητήσει αυτές τις εξελίξεις. Ε, τώρα, το θέμα του δωρεάν χαρακτήρα θα το δούμε εσχάτως. Αναφερθήκατε και στο θέμα της πιστοποίησης των δεδομένων. Ε, ρωτήσατε αν η Κομισιόν μπορεί να το κάνει ή όχι. Νομίζω ότι είναι σημαντικό να ξέρουμε πώς εργαζόμαστε για την πιστοποίηση των δεδομένων που είναι απαραίτητη. Και να ξέρω ότι κάποιοι είναι αντίθετοι στην αρχή της γραπτής πιστοποίησης γιατί θα τεθεί θέμα ευθύνη. Έτσι λοιπόν πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί για την έννοια, τον ορισμό που θα δώσουμε στην πιστοποίηση των δεδομένων. Αναφερθήκα και σε άλλες πτυχές που έχουν να κάνουν για την για αναφορά. Νομίζω ότι και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Ε, αυτά που προτείνεται είναι πολύ ενδιαφέροντα γιατί είναι σημαντικά συγκεκριμένα θέματα και διακυβεύονται πολλά. για την αγορά που θα γεννηθεί μέσω του GMES. Αυτά τα σχόλια στο στάδιο αυτό, αλλά θεωρώ ότι ήταν πολύ ενδιαφέρον το έργο σας και μας επιτρέπει να βελτιώσουμε το κείμενο και να ανοίξουμε και νέες προοπτικές για το δημόσιο τομέα, για τις επιχειρήσεις μας, αλλά έχουμε και το θέμα της ελεύθερης πρόσβασης των πολιτών. Σας ευχαριστώ. Και εγώ σας ευχαριστώ, συνάδελφος Χολ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε και ευχαριστούμε και τον κύριο Γκλάντε για την ε, έκθεσή του, ε, την οποία όλοι μας ε, βρίσκουμε ιδιαίτερα χρήσιμη και επικοδομητική. Υπάρχουν κάποια θέματα που θέλω να θίξω. Όσον αφορά το κατά πόσον θα υπάρχει περιορισμένη πρόσβαση στα δεδομένα ή όχι. Εγώ προσωπικά ανησυχώ ε, με την τροπολογία που θέλει να περιορίσει την πρόσβαση ε, σε πολίτες Ευρωπαϊκής Ένωσης και σε ε, φορείς της, γιατί θεωρώ ότι αντιβαίνει στην αρχή της ε, διαλειτουργικότητας, κάτι το οποίο διασφαλίσαμε στο πρόγραμμα Galileo και για, τα, για το πρόγραμμα GPS. Πρέπει λοιπόν να είμαστε πολύ προσεκτικοί. Τώρα, καθαρά πρακτικά. Θεωρώ ότι κάτι τέτοιο θα αποτελούσε φραγμό για τη χρήση δεδομένων πλευρά τρίτων χωρών για να αντιμετωπίσουν προβλήματα όπως είναι η κλιματική αλλαγή. Ε, θέματα που αφορούν όμως και εμάς. Ως εκ τούτου πρέπει το όλο θέμα να το δούμε κάπως πιο ανοιχτά και όχι να θεωρούμε ότι υπάρχει ένα οχυρό που αποκαλείται Ευρώπη όσον αφορά τα δεδομένα. Και το ακαθόδε πρόβλημα τη ε, πρόσβαση δεδομένων αν θα είναι δωρεάν ή όχι. Σύμφωνα με την κυρία Ντατή, ότι πράγματι εδώ πρόκειται για ένα ύπουλο, περίπλοκο θέμα και το πιο σωστό είναι αυτή τη στιγμή να παραμείνουμε ευέλικτοι. Εγώ ε, βλέπω να υπάρχουν πολλά πλεονεκτήματα αν η ε, χρήση δεδομένων είναι ελεύθερη και θα έχει πολύ πιο εύκολη πρόσβαση και μεγαλύτερη χρήση η βιομηχανία, αλλά το θέμα είναι ότι ε, είναι πολύ άκαμπτο αυτό το να το γράψουμε στη νομοθεσία. Γιατί με τον τρόπο αυτό ε, δεν θα μπορούσαμε να καλύψουμε ενδεχομένως κάποιες νέες εξελίξεις τεχνολογία που θα μπορούσαν να προκύψουν στο μέλλον. Σας ευχαριστώ. Επόμενος ε, ο κυρία Καμπαλέρο. Κύριε Κρεβάλη, ευχαριστώ. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον εισηγητή και συμφωνώ με όσα συμπεριλαμβάνονται στην έκθεση, αλλά για να μένα το πιο ανησυχητικό έχει να κάνει με τη χρηματοδότηση. Φράχη πρόθεσμα για το 2011-2013 φαίνεται να είναι διασφαλισμένη η χρηματοδότηση και θα δούμε και τον πινακά με τα δεδομένα της Κομισιόν, αλλά πρέπει να εγγυθούμε και τη βιωσιμότητα μέσω πρόθεσμα και μακροπρόθεσμα για την περίοδο 2014-2020. Εγώ ε, φοβάμαι ότι οι αναγκαιότητες χρηματοδότησης του προγράμματος μπορεί να υπερβούν τα κονδύλια που έχουν προβλεφθεί. Και Επομένως, θα χρειαστεί να κάνουμε μια σωστή, μια ορθή αξιολόγηση των αναγκαιοτήτων και να διασφαλίσουμε ότι υπάρχουν πηγές χρηματοδότησης για τις επόμενες δημοσιονομικές προοπτικές. Με... Έτσι δηλαδή θέλουμε να υπάρχει απαραίτητη χρηματοδότηση για το πρόγραμμα GMES. Δεν θέλουμε να επαναλάβουμε καταστάσεις που προέκυψαν στο παρελθόν σε σημαντικά προγράμματα για το μέλλον της Ευρώπης. Δηλαδή είδαμε στο παρελθόν ότι υπήρχε χρηματοδότηση για τα αρχικά στάδια και στη συνέχεια ήταν πολύ προβληματική χρηματοδότηση για τα στάδια εφαρμογής και ολοκλήρωσης ε, των προγραμμάτων με επιτυχία. Έτσι λοιπόν ε, είναι πολύ σημαντικό να διασφαλίσουμε τη βιωσιμότητα αυτού του προγράμματος που είναι ζωτικό για την ανταγωνιστικότητα και για τους Ευρωπαίους. Ευχαριστώ. Äh, πρόεδρος, και εγώ ευχαριστώ πολύ. Η κυρία Μουλαρίλη από την ε, Κομισιόν, παρακαλώ. Με συγχωρείτε, λέει ο Πρόεδρος. Είναι κύριος. Ο Πρόεδρος έκανε λάθος. Είναι κύριος. Η Κομισιόν, παρακαλώ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Δεν υπάρχει πρόβλημα που μπερδέψατε ε, το όνομά μου. Είμαι αρμόδιο ε, για το GMS e από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Από ό,τι καταλαβαίνω, σα πιέζει ο χρόνο. Θα είμαι σύντομο. Θα ήθελα να αντιδράσω για ορισμένα θέματα που τέθηκαν ε, από τον συγγητή και από του βουλευτέ που πήραν το λόγο. Καταρχήν, να σα ευχαριστήσω για το ενδιαφέρον σα ε, ε, και εγώ θεωρώ ότι οι συνεισφορές ε, είναι συγκλίνουσες και θετικές ε, για το πώς όλοι μας θα συνεισφέρουμε στην πρόοδο της ζημίας. E Τώρα για την ερώτηση που τέθηκε από τον εισηγητή για ένα ενδεχόμενο συνδυασμό των τροπολογιών 33 και 43 για την βαέλτιστη ε, χρησιμοποίηση των υφισταμένων δεδομένων. Νομίζω ότι υπάρχουν κάποιες δυνατές επιλογές. σε Αυτό το θέμα μπορεί να ρυθμιστεί στο ίδιο το πεδίο εφαρμογής του κανονισμού, λόγου χάρη μέσω των διατάξεων που διευκρινίζουν την ε, δραστηριότητα της πρόσβασης στα δεδομένα και μπορεί να υπάρχει και μια συνδήλωση σε σχέση με την πολιτική που ακολουθείται για τα δεδομένα. Νομίζω ότι πρέπει να σκεφτούμε μία από τις δύο αυτές δυνατότητες, αλλά είμαι βέβαιος ότι υπάρχει τρόπος ε, να εξεύρουμε μια κατάλληλη νομική διατύπωση. Σε ό,τι αφορά τώρα το θέμα της πολιτικής που ακολουθείται για τα δεδομένα. Νομίζω ότι η συζήτηση που έλαβε χώρα είναι πολύ σοφή. Η πρόθεση της Κομισιόν ήταν να διασφαλίσει ανεκτή πρόσβαση στα δεδομένα στο βαθμό που το όχι που έχουμε στην πρώτη παράγραφο του άρθρου 8 της πολιτικής των δεδομένων ε, χρήζει μια τέτοια προσέγγισης ε, σήμερα στο μεταβατικό στάδιο για ορισμένα δεδομένα θα μπορούσαμε να τα έχουμε δωρεάν για τα δεδομένα ε, φρουρούς που χρηματοδοτούνται από τον ΕΟΤ και την Ευρωπαϊκή Ένωση έχουμε δωρεάν άδειες ε, όμως δεν φαίνεται ότι το σύνολο των τομέων που καλύπτονται από το GMS e ε, είναι τόσο ξεκάθαρο αυτή τη στιγμή. Γι' αυτό μία πιο ανοιχτή αρχή που ανάλογα με τα διάφορα θέματα στο χρόνο θα δούμε αν θα είναι ανοιχτή η πρόσβαση δωρεάν ε, είναι κάτι προτιμητέο κατά την απόψή μας. Τώρα για την πιστοποίηση των δεδομένων είναι ένα πολύ σημαντικό ζήτημα και συνδέεται με την αξιοπιστία του συστήματος. Ε, οι πληροφορίες που παράγονται από το GMS e πρέπει να είναι ποιοτικέ. Εμπνεούμαστε από το μετεωρολογικό μοντέλο. Θεωρούμε ότι πρέπει να διασφαλίσουμε υποχρέωση των μέσων, να δράσουμε έτσι ώστε τα δεδομένα να είναι ποιοτικά, ανιχνεύσιμα και να σέβονται μία σειρά προτύπων ε, και θεωρούμε ε, ότι οι χειριστές των υπηρεσιών GMES θα πρέπει ε, να διασφαλίζουν την υλοποίηση των προτύπων αυτών γύρω από τις ε, ιδέες αυτές μπορούμε να συνεργαστούμε εμπνεόμενοι από το επιχειρησιακό μετεωρολογικό μοντέλο για να ε, υιοθετήσουμε αυτή την προσέγγιση και στην εκπόνηση του κανονισμού. Όμως δεν νομίζω τώρα ότι η διατύπωση που ακολουθείται στον κανονισμό είναι η καλύτερη. Ε, τώρα δεσμευόμαστε να ε, σας ενημερώνουμε για τα διαθέσιμα ποσά και για το κόστος ε, στις μεταβατικές περιόδους. Πολύ σύντομα θα έχετε τις πληροφορίες αυτές στη διάθεσή σας. Ευχαριστώ. Εμείς ε, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ε, κύριε Σιγητά, ε, χαίρομαι πάρα πολύ για τις ε, εισηγήσεις ε, που είχαμε μέχρι τώρα. θα γίνει και άλλη μια συζήτηση και θα επανέλθουμε. Και εγώ ευχαριστώ, λέει ο Πρόεδρος. Είναι σαφές το χρονοδιάγραμμα. Θα ήθελα απλά να επισημάνω ότι κατά πόσον ε, θα αποφασίσουμε στην ε, πρώτη ανάγνωση όχι. Το είπα ήδη η Ισπανική Προεδρία, το επιθυμεί αλλά και εμείς ε, δεν πρέπει να επιδιώξουμε πρώτη ανάγνωση με κάθε τίμημα. Δεν είναι αυτή η πεπατημένη. θα δούμε πώς θα εξελιχθεί. Επόμενο θέμα, αν επιτρέπετε, δεν έχουμε και πολύ χρόνο στη διάθεσή μας, αλλά η κυρία Γκροστέτ είπε ότι ίσως για το δικό της θέμα να μην χρειαστούμε και πάρα πολύ χρόνο. Η κυρία Νίπλα, διαδικαστικό. Κύριε Πρόεδρε, Κοιτάξτε, έχουμε ε, λάβει αλλαγή της ημερήσιας διάταξης και μετά την έκθεση Γκλάντε είναι η έκθεση του Σενόφσκι που θα προχωρήσουμε και εκεί πολύ γρήγορα. Δεν γίνεται. Μα πώς δεν γίνεται. Εγώ περίμενα γι' αυτό το σύνορα και αλλάξατε πάλι την ημερήσια διάταξη. Μα δεν γίνεται αυτό. Κάθενες από εμά ε, έχει υποχρεώσει σε το απόγευμα. Ε, θα πρέπει να πω στην νομική επιτροπή. Εγώ είμαι αρμόδια για την έκθεση αυτή και παρακαλώ να τηρήσουμε τη μέση διάταξη. Ε, Πρόεδρο, ο κύριο Τουχανόφσκι μου είπε ότι είχε κάποιε δυσκολίε. Ε, Α, ήρθε τώρα. Ναι, εντάξει, ήρθατε, αλλά είχατε πει ότι δεν θα αρχόσταν λόγω αεροπλάνου και γι' αυτό σήμερα το πρωί σε 9 αλλάξαμε τη μέση διάταξη. Πρόεδρος, ε, Τώρα δεν μπορώ να αλλάζω τη μέση διάταξη ανά 5 ανά 10 λεπτά. Ε, τα πράγματα γίνονται όλο και πιο δύσκολα, γιατί από ό,τι φαίνεται ε, δεν ισχύει πλέον το να είμαστε εδώ. Μάλλον η εξαίρεση γίνεται αυτό. Κύριε Μπιτεχόφερ, αφήστε μας ε, να είμαστε λιγάκι αυθόρμητοι και ας αντράξουμε την ευκαιρία που παρίσταται εδώ ο κύριος Τιχανόφσκι. τότε ίσως να έχει πρόβλημα η κυρία Γκροστέτ Τώρα, αν έχουμε να συζητάμε γι' αυτό, δεν θα κάνουμε ούτε το ένα ούτε το άλλο, τη μία την άλλη έκθεση. Α αποφασίσουμε στα γρήγορα, θα εξετάσουμε μία μόνο από τι ε, δύο εκθέσει. Ε, κυρία ε, Γκροστέτ, θέλετε να το συζητήσουμε ω πρώτο θέμα σήμερα το απόγευμα. Κυρία Γκροστέτε, κοιτάξτε και εγώ έφυγα από την Επιτροπή Περιβάλλοντος ε, για να έλθω εδώ. Είμαι εδώ, εδώ και κάποια ώρα και περιμένω. Έτσι λοιπόν ε, και εγώ ζητώ να το δούμε τώρα γιατί σήμερα το απόγευμα θα πρέπει να φύγω στις 3.30. Πρόεδρος, ε, αν προσπαθήσετε και οι δύο, ίσως μπορέσουμε να εξετάσουμε και τις δύο εκθέσεις. Επτά λεπτά στον καθένα για την έκθεσή σου. Σας φτάνει για την έκθεσή του αλλά θα πρέπει να είστε πάρα πολύ σύντομοι. Λοιπόν, η κυρία Γκροστέτ, δύο, δύο μόνο λεπτά ε, για την ε, εκθεσή της. Μετά θα έχουν δυνατότητα να μιλήσουν άδελφοι και μετά θα περάσουμε στο επόμενο θέμα. Θα είμαι πολύ σύντομη, Πρόεδρε. Θέλουμε να δημιουργήσουμε μια Ευρωπαϊκή Σύμπραξη για το 2009-2013 ε, για να υπάρχει ένα συντονισμό για την καταπολέμηση του καρκίνου, γιατί δυστυχώ εξακολουθούν να υπάρχουν πολλέ αποκλήσει και αντιλαμβανόμαστε Ό,τι τέτοιο. Ε, το 1 τρίτο των καρκίνων θα μπορούσαν να αποφευχθούν. Ε, όμως ε, δεν είναι ενδιαφέροντα αυτή τη στιγμή τα αποτελέσματα γιατί υπάρχουν καρκίνε όπως ε, της μήτρας ή του στήθους που θα έπρεπε να εξελιχθούν αν είχαμε μια καλή σύμπραξη καταπολέμηση του καρκίνου σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης. Έτσι λοιπόν ευχαριστώ τους συναδέλφους και κυρίως τον κύριο Κάμπος που μου έκανε μια σειρά προτάσεων για την εκθέση αυτή. Λυπάμαι που δεν υπάρχει προσθέτη χρηματοδότηση για τη σύμπραξη αυτή έτσι λοιπόν θα πρέπει να κάνουμε με τα κονδύλια προτείνονται στο 7ο πρόγραμμα πλαίσιο. Τώρα με το 6ο πρόγραμμα πλαίσιο και με τις ε, δύο πρώτες προσκλήσεις υποβολής προκτήσεως ε, του 7ου ε, προγράμματος έχουμε 750 εκατομμύρια που καλύπτουν όλα τα μεγάλα είδη καρκίνου και συμμετέχουν οι μικρές και μεσές επιχειρήσεις, τα πανεπιστήμια και σημαντική βιομηχανική εταίρεια. Αλλά πρέπει να χρησιμοποιήσουμε καλύτερα τους σπόρους και να καταβάλουμε μεγαλύτερε προσπάθειες για την καταπολέμηση του καρκίνου. Έχουν αναλυφθεί πολύ σημαντικέ προσπάθειε δυστυχώ ο όγκο των εξετάσεων ανείχνευση δεν φτάνει ε, στο ίμιση του αριθμού των εξετάσεων που θα έπρεπε να υλοποιήσουμε. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προτείνει μία δομή ε, που μου φαίνεται πραγματικά πολύ επαχθή. Ε, εφιστώ την προσοχή σας σε αυτό. Ζητά να δημιουργηθεί ένα φόρουμ με ομάδες ε, καθοδήγησης, με ομάδα εργασία. Θα ήθελα να πω στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή να μην ε, δημιουργήσουμε κάτι που θα μας φρενάρει. Θα πρέπει να ενθαρρύνουμε περισσότερο τι συμπράξει ιδιωτικού τομέα για να δώσουμε κίνητρα στην έρευνα και στην ανείχνευση σε ό,τι αφορά την ιατρική επικόνηση κυρίω. Θα πρέπει να συνεργαστούμε πιο στενά με το Διεθνέ Κέντρο Ερευνών για τον Καρκίνο, όπω προτείνουν κάποιοι συνάδελφοι και αυτό είναι πολύ καλή ιδέα. Θα πρέπει επίση να μην ξεχνάμε την πρόληψη σε δευτερογενέ και σε πρωτογενέ επίπεδο, αλλά και τον έλεγχο των νόσων που μπορούν να εξελιχθούν ω καρκίνο και κυρίω ε, για το θέμα τη έρευνα, Εκτιμώ ουσιαστικό να υπενθυμίσουμε πόσο επιτακτικό είναι να συστήσουμε ένα ευρωπαϊκό δίπλωμα ευρωστεχνία. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Merci beaucoup. Πολύ ωραίο. Κύριος Χατζή Μαρκάκης, παρακαλώ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ε, θα ήθελα να υποστηρίξω τη συνάδελφο σε όλα αυτά που είπε. Πράγματι, είπε τα σημαντικότερα. Ε, χρειαζόμαστε καλύτερο συντονισμό. Η έρευνα για τον κακίνο είναι μεγάλο πρόβλημα και για την Ευρωπαϊκή Ένωση και για ολόκληρο τον κόσμο. Πρέπει να συντονίσουμε καλύτερα τα ερευνητικά προγράμματα. Ε, διεξάγονται και παράλληλε έρευνε. Αυτό δεν είναι απαραίτητο πλέον στην Ευρώπη, γιατί απαιτεί και περισσότερα κονδύλια. τα προγράμματα ΣΔΙΤ ενδείκνυνται ιδιαίτερα και τούτο το γνωρίζουμε και από άλλες πρωτοβουλίε όπου ε, μπορούμε να αποκτήσουμε ακόμη περισσότερο ιδιωτικά κονδύλια. Και τέλος ε, το Ευρωπαϊκό Δίπλωμα Ευρεσιτεχνία αποτελεί ένα περαιτέρω κίνητρο. Εδώ λοιπόν καλούνται τα κράτη-μέλη επιτέλους να επιταχύνουν. Ο κύριος Κορέα Δεκάμπους. Ναι, Πρόεδρε, ευχαριστώ. Πρόεδρε, α, συγγνώμη έχουμε μία θέση θετική απέναντι στο έγγραφο και ήδη συνεισφέρεμε με πολλές σκέψεις ε, και σχόλια στα οποία αναφέρθηκε η κυρία Γκρουστέτ προλίγου. Έχω ένα γενικό σχόλιο. Εμείς ε, θα θέλαμε να αναπτυχθεί περισσότερο στο έγγραφο το ε, θέμα ότι ε, μπορούμε να έχουμε πλεονεκτήματα από τη σύγκριση η καταπολέμηση του καρκίνου είναι πρόβλημα των κρατών μελών, είναι θέμα επικουρικότητα βασικά, αλλά υπάρχουν ε, προφανή ωφέλη αν υπάρχει ευρωπαϊκή οργάνωση και ε, μπορούμε να πούμε ότι είχαμε ε, πάνω και κάτω σε όλο αυτό το εγχείρημα. Στο παρελθόν είχαμε ε, κάποιες πρωτοβουλίες που είχαν αναλυφθεί όπως ένα ακρονίμιο, όμως τώρα βρισκόμαστε σε πολύ χαμηλή άλλα επίπεδα, σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Εμείς θα προσπαθήσουμε πάντως τις επόμενες ημέρες να στείλουμε τα σχολιά μας. Ευχαριστώ. Σας ε, ευχαριστώ. Η προθεσμία είναι 2 Φεβρουαρίου. Έτσι λοιπόν κλείνει αυτό το θέμα της ημερήσιας διάταξης. Παρακαλώ την Κομισιόν να δείξει κατανόηση ότι σήμερα επειδή έχουμε έτσι μια ε, πιεσμένη διαδικασία δίνω προτεραιότητα περισσότερο στο Κοινοβουλίο. Πάμε στο επόμενο θέμα που είναι το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Πλοήγησης. Ε, ζητώ συγγνώμη, λέει ο κύριο Τσενόφσκι, ο εισηγητής ε, για το ότι επικράτησε αυτό το χάος. Καθυστέρησα να έρθω. Αλλά ξέρετε, εμεί είχαμε στην Πράγα μείον 20 και κόλλησε εκεί και δεν μπορούσε να φύγει το αεροπλάνο. Το ε, πρόγραμμα λοιπόν της δορυφορικής πλοήγησης. Αυτό το συζητήσαμε σε πάρα πολλές συνεδριάσεις με τους συναδέλφους, με εισηγητές και Έχω λάβει 15 τροπολογίες. Προσπαθούμε λοιπόν ε, ή δυνατόν να βρούμε κάποιες ε, λύσεις ε, για τις τροπολογίες αυτές, γιατί ορισμένες εξ αυτών επικαλύπτονται. Αφορούν κατά κύριο λόγο τρεις τομείς. Πρόκειται για τη συμμετοχή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στις εργασίες του Ευρωπαϊκού Οργανισμού κατά πόσον ε, οι υπάλληλοι θα έχουν το καθεστώς του παρατηρητή, ε, κατά πόσον θα μπορούν να ψηφίσουν ή όχι. Το δεύτερο πρόβλημα είναι το εξής. Ε, πρέπει να προσπαθήσουμε να αναζητήσουμε ισορροπίες στο Συμβούλιο γιατί η Κομισιόν έχει σημαντικό ρόλο, φέρει την ευθύνη για το σύνολο του προγράμματος και εμείς προσπαθούμε να αναζητήσουμε μια τέτοια λύση η οποία αφενός θα μας δίνει τη δυνατότητα ουσιαστικής ε, παρέμβασης για την ε, περίπτωση κατά την οποία οι προτάσεις ε, των εκπροσώπων των κρατών μελών ξεπερνάνε το δημοσιονομικό πλαίσιο. Αφετέρου όμως θα πρέπει να διατηρήσουμε την ενεργό συμμετοχή των κρατών μελών έτσι ώστε να μπορούν και τα κράτη-μέλη να δείξουν το ενδιαφέρον τους. Και τα κράτη-μέλη θα πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να επιβάλλουν τις προτάσεις τους. Είμαστε στο 30 ε, μέχρι 40 της ε, εκατό ε, της διάθεσης της Κομισιόν. Αυτά είναι ποσοστά που αφορούν τη διάθεση, γιατί απλά θέλω να δείξω ότι όλοι ενδιαφέρονται. Το τρίτο που θέλω να πω αφορά την ε, ε, θέση μας σχετικά με την διαπίστευση, τη διασφάλιση διαπίστευσης ε, των υπαλλήλων. Αυτό με ενδιαφέρει εμένα πάρα πολύ. πρόκειται για το πώς θα λειτουργήσει αυτή η διαδικασία διαπίστευση. Από την άλλη, θεωρώ επίσης ότι θα κατορθώσουμε το συντομότερο δυνατόν να καταλήξουμε σε συμβασμό. Ε, θα έχω ακόμα περισσότερες συναντήσεις με τους ε, σκιώδεις εισηγητές και νομίζω ότι πλησιάζουμε σε μια καλή ε, λύση. Θα ήθελα λοιπόν να ευχαριστήσω τους συναδέλφους για την συνεργασία, την αγαστή συνεργασία, γιατί η συνεργασία αυτή θα μας επιτρέψει ε, στο να προχωρήσουμε ταχύτατα. Ευχαριστώ ε, πάρα πολύ κύριε Πρόεδρε. Νομίζω ότι τήρησα το χρονικό διάστημα που μου είχατε διαθέσει. Η κυρία Νίπλε, Ευχαριστώ πολύ κύριε ε, Πρόεδρε. Ε, θα ήθελα να ευχαριστήσω και τον ε, κύριο Τουσινόφσκι, ο οποίος κάλεσε όλους τους σκιώδης για να καταλήξουν σε μια συμβαστική πρόταση. Το θέμα που τίθεται είναι ο οργανισμός, αυτό είναι το ένα, και δεύτερον πώς θα εκπροσωπείτε το Κοινοβούλιο στο Διοικητικό Συμβούλιο και πώς θα σταθμίζονται οι ψήφοι επεξεργαζόμεθα μια συμβαστική πρόταση που να μπορεί να τη στηρίξει και η δική μας η πολιτική ομάδα. Δεν θέλω να μπω σε λεπτομέρειες, νομίζω όμως ότι είμαστε σε καλό δρόμο και μέχρι αύριο θα μπορέσουμε να έχουμε βρει καλές συμβαστικές προτάσεις και να ε, καταλήξουμε στο συμβασμό. Επόμενος ο κύριος Γκλάντε. Πρόεδρε, υπογραμμίζω ανεπιφύλακτα αυτά που είπε η συνάδελφο κυρία Νίπλα. Και η δική μου η πολιτική ομάδα θα είναι παρούσα στι ε, συμβαστικέ ε, προτάσει πρέπει να δούμε λιγάκι πώς θα σταθμιστούν οι ψήφοι, ε, ποιο θα είναι το βάρος ε, της ε, ψήφου της Κομισιόν. Οι εκπρόσωποι του Κοινοβουλίου πρέπει να επαγρυπνούν. Πάντως είχαμε πολύ καλή συνεργασία και για άλλη μια φορά ευχαριστούμε τον κύριο Κοζανόφσκι. Συνάδελφος κυρία Εκ, και εμείς θα θέλαμε να εκφράσουμε την ικανοποίησή μας για την έκθεση, την ποιότητα της έκθεσης και προσβλέπουμε στο συμβαστικό κείμενο. Σας ευχαριστώ. Πρόεδρος, πάρα πολύ ωραία. Ε, πολύ γρήγορα τα είπατε, αλλά ομολογώ με εντυπωσιάσατε. Ε, 17 Μαρτίου θα ψηφίσουμε και νομίζω ότι δεν πρέπει να δεσμευθούμε ότι ε, θα ολοκληρώσουμε τη διαδικασία σε πρώτη ανάγνωση. Το επαναλαμβάνω, αυτή δεν είναι υπεπατημένη. Υπάρχει άλλη υπεπατημένη. Στις 17 Μαρτίου θα ψηφίσουμε για όλα και θα δούμε μετά πώς θα προχωρήσουμε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που με βοηθήσετε, ειδικά τώρα στο τέλος, να παραμείνω μέσα στο χρονοδιάγραμμά μου. Βέβαια, ο Υπουργός δεν έχει έρθει ακόμα ή μήπως ήρθε.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 ή όχι. Αν ήρθε παρακαλώ να περάσει. Yeah? Uh, no, no, no. We are in time and then we can start. <laughs> Herzlich willkommen. Σας καλωσορίζω εγκαρδιότατα κύριε Υπουργέ στην Επιτροπή μας εδώ. Θα ήθελα να παρουσιάσω τον κύριο Σεμπαστιάν, Υπουργό Βιομηχανία Εμπορίου και Τουρισμού τη Ισπανία, που θα ασκεί την Προεδρία του Συμβουλίου. Χαίρομαι που έχουμε την ευκαιρία να σα δούμε. Είσαστε ο πρώτο Ισπανό Υπουργό που έρχεστε εδώ στη συνεδρίασή μα. Θα έχουμε και κάποιου άλλου επαφέ και χαίρομαι που έχουμε σήμερα τη δυνατότητα να συζητήσουμε μαζί σα. Μια μισή ώρα έχουμε προβλέψει περίπου. Θα σας δώσω καταρχήν δυνατότητα να μας κάνετε μια γενική παρουσίαση των στόχων της Προεδρίας. Μετά οι συνάδελφοι μπορούν να υποβάλουν ερωτήσεις. Λοιπόν, δεν θα μακρηγορήσω εγώ τώρα. Σας χαιρετίζω, σας καλωσορίζω και σας δίνω το λόγο κύριε Υπουργέ. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Αξιότιμε Πρόεδρε, μέλο τη Επιτροπή Βιομηχανία, Έρευνα και Ενέργεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Για μένα είναι τιμή να παρευρεθώ ενώπιόν σα και να παρουσιάσω τις προτεραιότητε ε, που θέσπισε η Ισπανική κυβέρνηση για τον τομέα τη αντιγωνιστικότητα για το ξάμεινο τη Προεδρία. Ε, επιτρέψτε μου επίσης να εκφράσω την αναγνώρισή μου στην ε, προκατοχό μας, ε, τη Σουηδική Προεδρία, για το εξαιρετικό έργο που επιτέλεσε σε στενή συνεργασία με όλους εσάς στους ε, τομείς της αρμοδιότητας αυτής της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής. Η πρόθεσή μας είναι να συνεχίσουμε αυτή την οδό και μάλιστα περισσότερο τώρα που ως συνέπεια της θέσης ισχύ της Συνθήκης Λισαβόνας οι αρμοδιότητες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου έχουν ενισχυθεί καταλήλως. Είμαστε η πρώτη Προεδρία η οποία θα σκίσει τις αρμοδιότητές της ε, υπό ε, τη συνθήκη της Λισαβόνας και ε, θεωρούμε ότι το να παγιώσουμε τις διοργανικές σχέσεις αποτελεί βασική προτεραιότητα για αυτό το πρώτο εξάμεινο του τρίου των Προεδριών όπως επίσης και όχι σε μικρότερο βαθμό είναι προτεραιότητα να θέσουμε σε εφαρμογή αυτό που ζητούν οι Ευρωπαίοι πολίτες και οι επιχειρήσεις από τα ευρωπαϊκά όργανα για να ε, ανακτήσουμε ε, την οικονομική μας δραστηριότητα. Σε συνεργασία με το Βέλγιο και την Ουγγαρία έχουμε εκπονήσει ένα πρόγραμμα εργασίας για το επόμενους 18 μήνες που έχει ως στόχο φαινός και βραχυπρόθεσμα να συνεισφέρει ε, στο να δημιουργήσει τις απαραίτητες προϋποθέσεις έτσι ώστε οι ευρωπαϊκές οικονομίες να ξεπεράσουν το συντομότερο τη σημερινή κατάσταση οικονομικής τελμάτωσης ε, οθώντας, προωθώντας μια ταχύ ανάκαμψη και μακροπρόθεσμα να θέσουμε τις βάσεις έτσι ώστε η ευρωπαϊκή οικονομία να αποκτήσει τα απαραίτητα στοιχεία για να δημιουργηθεί ένα βιώσιμο, ισορροπημένο και ανταγωνιστικό μοντέλο. Το πρόγραμμα της Ισπανικής Προεδρίας θα προσπαθήσει να δώσει απάντηση σε αυτές τις δύο προκλήσεις σε ό,τι αφορά στον τομέα της ενέργειας, ο πρώτος μας στόχος είναι το επόμενο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, ε, το ΕΡΙΝΟ, να υιοθετήσει το σχέδιο δράσης 2010-2014, ένα σχέδιο στο οποίο η ουσιαστική ολοκλήρωση της αγοράς ενέργειας θα είναι ένα από τα ε, θεμελιώδη στοιχεία. Ε, γι' αυτό θα πρέπει ειδικά να εστιαστούμε στην ε, αύξηση των διασυνδέσεων και στη ρυθμιστική εναρμόνιση. Σε ό,τι αφορά την πρώτη πτυχή, θα εργαστούμε έτσι ώστε η ικανότητα διασύνδεσης μεταξύ των κρατών μελών να φτάσει, η δυναμικότητα να φτάσει το 10% των ε, αντίστοιχων ε, ισχύων. Ε, όπως, επίσης, ε, συνάπτοντας τις απαραίτητες συμφωνίες, ε, θα προσπαθήσουμε το νέο μέσο ενεργειακής ασφάλειας ε, να υλοποιηθεί το συντομότερο και θα δημιουργήσουμε προγράμματα ηλεκτρικών διασυνδέσεων στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού Δικτύου Ενέργειας. Επίσης, ε, από τη σκοπιά της εσωτερικής αγοράς ενέργειας είναι πολύ σημαντικός ο ρόλος που η ρυθμιστική εναρμόνιση θα διαδραματίσει για το μελλοντικό οργανισμό συνεργασίας ρυθμιστικών αρχών ενέργειας. Κατά το εξάμεινο της δικής μας Προεδρίας ε, θα προωθήσουμε να τεθεί σε εφαρμογή, σε λειτουργία το συντομότερο δυνατόν. Σε ό,τι αφορά την ασφάλεια του εφοδιασμού θα εργαστούμε έτσι ώστε ο κανονισμός ε, για τον ενεργειακό φυδιασμό σε αέριο να υιοθετηθεί η Ποσπενική Προεδρία και για στο, τις εξωτερικές σχέσεις θέλουμε να ενισχύσουμε το διάλογο με τις τρίτες χώρες ε, διέλευσης, ε, προμήθειας και κατανάλωση ενέργειας. Θα εργαστούμε για να προλάβουμε πιθανές κρίσεις ενεργειακού εφοδιασμού στην Ευρώπη και θα δώσουμε ιδιαίτερη προσοχή στις σχέσεις με τους κύριους ενεργειακούς προμηθευτές και τις χώρες ε, διέλευση. Όλοι γνωρίζουν ότι η ασφάλεια του εφοδιασμού βελτιώνεται με την ενεργειακή αποδοτικότητα και την προώθηση των ενώσιμων πηγών ενέργεια. Προ την κατεύθυνση αυτή, ο στόχο τη βελτίωση ε, τη ενεργειακή αποδοτικότητα ε, θα αποτελέσει ένα στοιχείο σημαντικό μέσα στο σχέδιο δράση 2010-2014 για την Ισπανική Προεδρία, εν ώψη του Ευρωπαϊκού Σχεδίου του 6 για την ενεργειακή αποδοτικότητα. Σε ό,τι αφορά τι καθαρέ πηγέ ενέργεια, εμεί ε, έχουμε ω προτεραιότητα το να μεταφερθεί η κοινοτική νομοθεσία στο ιστορικό δίκαιο τη κάθε χώρα. Γι' αυτό θα θέσουμε σε εφαρμογή τα σχέδια εθνική δράση ε, και έχουμε ως στόχο την 30 Ιουνίου θα αφιερώσουμε προσπάθειες ε, στις ενεργειακές τεχνολογίες με χαμηλές εκπομπές άνθρακα, όπως είναι το σχέδιο SET. Ε, στην κατεύθυνση αυτή θέλουμε να υιοθετήσουμε συμπεράσματα στο Συμβούλιο του Μαρτίου που θα σας επιτρέψουν να έχουμε νέες πρωτοβουλίες βιομηχανικές και να επιτραπεί και η χρηματοδότησή του. Στο παρελθόν, ε, οι ορυκτές πηγές ενέργειας αποτέλεσαν ε, πηγή συγκρούσεων και πολέμων με περασμένος χαρακτήρας τους οδήγησε σε οικονομικές και πολιτικές εντάσεις ε, που δυσκόλεψαν τη συνεννόηση μεταξύ των χωρών. Πρέπει να τεθεί τέλος στην τάση αυτή η εμφάνιση νέων ενεργειακών πηγών ε, καθαρών και ανεξάντλητων ανοίγει νέες προοπτικές βιωσιμότητας αλλά και συνεργασίας και ειρήνης. Και με το πνεύμα αυτό και στο πνεύμα αυτό, ε, μία από τις προτεραιότητες που έχουμε θέσει για το εξάμεινο της Προεδρίας μας είναι να προωθήσουμε το Μεσογειακό Ηλιακό Σχέδιο. Η Ισπανική Προεδρία έχει την πρόθεση να οργανώσει στη Βαλένσια 11 και 12 Μαΐου 2010 μια συνδιάσκεψη για το σχέδιο αυτό. τα συμπεράσματα θα μπορέσουν να εγκριθούν στη σύνοδο Euromed που θα λάβει χώρα τον Ιούνιο στη Βαρκελόνη. Η ενέργεια θα είναι ένα σημαντικό στοιχείο στην ικανότητα την ανταγωνιστική της Ευρωπαϊκής Ένωσης όπως ήδη είναι και θα πρέπει να συνεχίσουν να είναι οι τεχνολογίες τεχνολογιών και πληροφοριών αξιότιμοι κύριοι βουλευτέ, στον τομέα των λεπικοινωνιών και στην ανάπτυξη τη κοινωνία, τη πληροφόρηση, η στρατηγική μα περνά από την ανάπτυξη αυτού του τομέα, το τομέα των χειρολογικών επικοινωνιών και πληροφοριών, ε, οι οποίε ε, είναι απαραίτητε για να δημιουργηθεί μια ανταγωνιστική και σταθερή Ευρώπη. Καθώ είναι πολύ σημαντικό αυτό ο τομέα, κατά τη διάρκεια του εξαμήνου τη Προεδρία μα θα ξεκινήσουμε μια νέα στρατηγική για την περίοδο η οποία θα λέγεται για μια ψηφιακή Ευρώπη, στρατηγική της Γρανάδα, ε, τεχνολογίες, ποιότητας της ζωής, παραγωγικότητας και η στρατηγική αυτή θα αντικαταστήσει την ε, στρατηγική I 2010 και θα εγκριθεί στο άτυπο Συμβούλιο Υπουργών Τηλεπικοινωνιών που θα λάβει χώρα στη Γρανάδα 19 και 20 Απριλίου φέτος και θα λάβει υπόψη τις ε, προτάσεις της έκθεσης ε, της Σουηδικής Προεδρίας. Το κεντρικό στοιχείο της στρατηγικής της Γρανάδα 2010-2015 θα είναι δημιουργηθεί μια νέα ψηφιακή αγορά μια νέα ψηφική αγορά που θέλουμε να ε, θεωρηθεί ως η πέμπτη ελευθερία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η σύστασή της θα επιτρέψει αφενός ε, να εντοικοποιηθεί η ίδια το διασυνοριακό ηλεκτρονικό εμπόριο και να προωθήσει αφετέρου τη βιομηχανία των ε, ψηφιακών αγαθών και υπηρεσιών και κυρίως των ψηφιακών περιεχομένων. Για να εκμεταλλευτούμε το δυναμικό της ενιαίας ψηφιακής αγοράς πρέπει να καταργήσουμε τα εμπόδια για την επίτευξή της. Ε, αναφέρομαι στο να υπάρχουν δίκτυα νέας γενιάς, προσβασιμότητα και προστασία των δικαιωμάτων των χρηστών ε, των ηλεκτρονικών μέσων επικοινωνιών. Και γι' αυτό η στρατηγική της Γρανάδας στη στρατηγική της Γρανάδα καταρχήν θα θέσουμε στόχους και μέσα και εργαλεία έτσι ώστε να κλείσει το δεύτερο ψηφιακό χάσμα και θα προωθήσουμε την ανάπτυξη δικτύων νέας γενιάς μέσω του καθορισμού ενός ευνοϊκού νομικού πλαισίου και της απαραίτητης Δημοσιονομική στήριξης ε, θα ε, εκπονήσουμε σε ευρωπαϊκό επίπεδο ένα, μια ευρωπαϊκή χάρτα των χρηστών, των ηλεκτρονικών επικοινωνιών, σύμφωνα με αυτό που υθετήσαμε πρόσφατα στην Ισπανία η απασχόληση και η ανταγωνιστικότητα είναι οι πυλώνε στου οποίου βασίζεται η οικονομική ανάπτυξη, αλλά στον 21ο αιώνα η ανάπτυξη αυτή καθ' ε, δεν φτάνει για να πετύχουμε την αηφορία. Πρέπει να υπάρχει και σεβασμό στο περιβάλλον σε ένα ουσιαστικό στοιχείο τη οικονομική ανάπτυξη. Προ την κατεύθυνση αυτή, τεχνολογίε τεχνολογίες επικοινωνιών και πληροφοριών ε, αποτελούν ένα σημαντικό παράγοντα για την επίτευξη των περιβαλλοντικών στόχων που έχουμε θέσει για το 2020 Τεχνολογίε, αυτέ πρέπει να διαδραματίσουν ένα θεμελιώδη ρόλο στην παγίωση ενιών όπω είναι η ενεργειακή αποδοτικότητα και η οικολογική αποδοτικότητα. Θα προωθήσουμε τι βιντεοσκέψεις, το ηλεκτρικό αυτοκίνητο, τη τηλεεργασία, τα έξυπνα δίκτυα, smart nets και τους έξυπνους μετρητές smart meters μεταξύ άλλων και γι' αυτό ο ρόλος ε, των TPE ε, ε, θα είναι μαζί με την ενιαία ψηφιακή αγορά τα δίκτυα τα νέα δίκτυα και την υπέρβαση του δεύτερου ψηφιακού χάσματος και το χάρτη των δικαιωμάτων των χρηστών θα είναι ο πέμπτος πυλών στρατηγικής της Γρανάδας. Τώρα, για τι τεχνολογίε αυτέ θα προωθήσουμε δύο ακόμα δράσει. Θα εργαστούμε αφενό για να ενισχύσουμε την εμπιστοσύνη και την ασφάλεια στα δίκτυα, και την προστασία των δικαιωμάτων πνευματικής διοκτησίας στο διαδίκτυο. Και αφετέρου θα προσπαθήσουμε να συνάψουμε μια συμφωνία που να επιτρέπει την εκπόνηση ενός συναρμονισμένου πλαισίου για την παραγωγή δικτών της κοινωνίας ε, της πληροφορίας. Κυρίε και κύριοι, η πρόσφατη οικονομική κρίση είχε πολύ μεγάλο αντίκτυπο στην βιομηχανική δραστηριότητα όλων των κρατών μελών. Ε, συνέπεια είναι ότι σε πολλέ χώρε ελήφθησαν μέτρα στήριξη για το βιομηχανικό τομέα. Θα πρέπει να σκεφτούμε ως ποιο σημείο αυτά τα μέτρα ε, σήμαιναν αλλαγή της βιομηχανικής πολιτικής των ευρωπαϊκών χωρών ταυτόχρονα. Όπως επίσης πρέπει να αναλύσουμε την αποτελεσματικότητα των μέτρων αυτών και το ρόλο της βιομηχανικής πολιτικής ε, με ορίζοντα το 2020. Η δική μας πρόθεση είναι ο προβληματισμός αυτός να γίνει στο πλαίσιο της Ισπανικής Προεδρίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, συνεισφέροντας έτσι στο να τεθούν οι βάσεις για τη μελλοντική βιομηχανική πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μια βιομηχανική πολιτική που θα πρέπει να είναι ικανή να προωθήσει την αηφορία και την ε, ε, ικανότητα καινοτομία της βιομηχανίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης για να είμαστε ανταγωνιστικοί στις παγκοσμίες αγορές. Μια προώθηση της αηφορίας και της ε, ικανότητας της καινοτομίας στο ε, στον τομέα της αυτοκινητοβιομηχανίας ε, έχει ένα κύριο σύμμαχο μέσω του ηλεκτρικού αυτοκινήτου. Είμαι πεισμένη κύριε βουλευτέ, ότι η Ευρώπη όχι μόνο εδώ με το ηλεκτρικό αυτοκίνητο ουσιαστικά διακυβεύει το μέλλον της, το ενεργειακό μέλλον, αλλά και την τεχνολογική ανάπτυξη. Το να στοιχηματίσουμε υπέρ του αυτοκινήτου, ηλεκτρικού αυτοκινήτου σημαίνει ότι θα έχουμε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, χρησιμοποιούμε ενώσιμε πηγέ ενέργεια, θα εξαρτώμαστε λιγότερο από το πετρέλαιο και το, θα μειώσουμε την εξαρτησή μας από το πετρέλαιο και αν το πράξουμε αυτό και προωθήσουμε ταυτόχρονα τι ανανεώσιμε πηγέ ενέργεια, θα κάνουμε ένα ποιοτικό άσμα σε ό,τι αφορά την ανταγωνιστικότητα, την ασφάλεια και το σεβασμό του περιβάλλοντο και την ευημερία. Ε, το 2008 η Ευρωπαϊκή Ένωση χρειάστηκε να εισαγάγει περίπου το 90% ε, των αναγκών κατανάλωση πετρελαίου, δηλαδή 4,4 δις ε, βαρέλια πετρελαίου. Αν για την επόμενη δεκαετία οι προβλέψει υλοποιηθούν για το πετρέλαιο, η τιμή του πετρελαίου θα αυξηθεί κατά 30 ευρώ δηλαδή, ε, τότε αυτό σημαίνει ότι στις ε, χώρες εξαγωγής ε, πετρελαίου θα μεταφέρουμε 132 πρόσθετα δισεκατομμύρια κέρδος ετησίως. Και αυτό ισοδυναμεί με όλο τον κοινοτικό περιπροσωπικό για το 2010 το ηλεκτρικό αυτοκίνητο όχι μόνο αποτελεί μια βιομηχανική και ενεργειακή ευκαιρία, αλλά και μια τεχνολογική ευκαιρία. Ε, η εφαρμογή του ηλεκτρικού αυτοκίνητου σημαίνει ότι θα αναπτυχθεί software για ε, το φορτισμό των μπαταριών και θα αναπτυχθεί ε, και ένα δίκτυο έξυπνο και έξυπνοι μετρητές. Η εφαρμογή του ηλεκτρικού αυτοκίνητου χρειάζεται επίσης ε, χρήζει ενό διατομεακού διαλόγου μεταξύ του βιομηχανικού τομέα, του ενεργειακού τομέα και του τομέα των ΤΠΕ. Κυρίε και, και κύριοι, κύριε Πρόεδρε, εμείς ε, πιστεύουμε στο ότι η χρήση του ηλεκτρονικού αυτοκινήτου μπορεί να ε, οδηγήσει στο να παγιώσει ένα νέο μοντέλο ανάπτυξης που χρειάζεται η ευρωπαϊκή οικονομία. Γι' αυτό η, ευρωπαϊκή Ισπανική Προεδρία θα προωθήσει σε ευρωπαϊκό επίπεδο μια συζήτηση για τα πιθανά μέτρα που μπορεί να θετηθούν για την προώθηση ε, τη χρήση του ηλεκτρικού αυτοκινήτου, τη παραγωγή του ηλεκτρικού αυτοκινήτου από την ευρωπαϊκή βιομηχανία και θα προωθήσει και τη χρήση του. Θέλουμε να προωθήσουμε τη συζήτηση και τον προβληματισμό επί του θέματο αυτού. Έτσι λοιπόν θα προτείνουμε την υιοθέτηση μιας ευρωπαϊκής στρατηγικής για το ηλεκτρονικό αυτοκίνητο που θα προσεγγιστεί ως κεντρικό θέμα στο άτυπο Συμβούλιο ανταγωνιστικότητα που θα λάβει χώρα το Φεβρουάριο στο Σαν Σεμπαστιά. Τέλος, ε, επιθυμούμε το Συμβούλιο Ανταγωνιστικότητας ε, που θα λάβει η χώρα το Μάιο να θετήσει συμπεράσματα και να συμπεριλαμβάνει τις δεσμεύσεις που θα αναλάβουν τα κράτη-μέλη για την πρόθεση τέτοιων αυτοκινήτων. Επίσης, στα πλαίσια της βιομηχανικής πολιτικής ε, προτιθέμεθα να εργαστούμε στα ακόλουθα. Καταρχήν, θα προωθήσουμε την εφαρμογή του νόμου των μικρών, για τις μικρές επιχειρήσεις, δηλαδή το Small Business Act και δεύτερον, θα προωθήσουμε την εκπόνηση μιας μελέτης για τις προοπτικές ε, του, ε, της κοινωνικής, του, κοινωνικού, του ευρωπαϊκού με συγχωρείτε σήματος, της ευρωπαϊκής μάρκας, ε, προκειμένου να προστατεύσουμε τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας. Πρόεδρε, αξιότιμοι κύριοι βουλευτέ, η κυβέρνηση τη Ισπανία ό,τι αφορά την πολιτική τη ανταγωνιστικότητα ε, έχει μια πολύ μεγάλη ημερησία διάταξη για το θέμα τη ανταγωνιστικότητα ε, και λαμβάνουμε υπόψη τι προκλήσει που τίθεται στο ορίζοντα του 2010, έναν ορίζοντα που ε, μπορεί να είναι υποσχόμενο και με ελπίδα παρά του κακού ιονού, αν όλοι συμφωνήσουμε επί των οδών που οδηγούν στην καινοτομία, την ανταγωνιστικότητα και τη βιωσιμότητα ε, με ε, την ε, δέσμευση που αξίζουν οι πολίτες μας και οι επιχειρήσεις μας. Έτσι λοιπόν σε αυτό έχετε τη στήριξη της Ισπανικής κυβέρνησης. Σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Υπουργέ. Ευρύ φάσμα θεμάτων. Αυτό οδήγησε ότι πολλοί συνάδελφοι ζητούν το λόγο. 15 ονόματα έχω ήδη καταγράψει. Θέλει κάποιο άλλο το λόγο. Θα τον κλείσουμε. Εδώ. Να. Und hier Dann Κλείνω ο κατάλογος εδώ. Και θα ήθελα να σας παρακαλέσω να συμφωνήσουμε όλοι να αρκεστούμε σε δύο λεπτά για ερώτηση για να μπορεί να υπάρξει και μια αναλυτική απάντηση μετά που είναι πάρα πολύ σημαντικό. Και να βάλουμε το ρολόι να τρέχει νομίζω γιατί είναι καλό να βλέπει κανένας ότι περνάει ο χρόνος του. Και τελειώνουμε στις 12.30 έτσι κι αλλιώς. Κύριε Δικαστήριο, η πρώτη θα υποβάλει ερώτηση. Ε, Ευχαριστώ Πρόεδρε. Ευχαριστώ κύριε Υπουργέ, εξ ονόματος της ομάδας μου. Θα ήθελα να σας καλωσορίσω στην Επιτροπή αυτή και να σας ευχαριστήσω για την παρουσία σας εδώ. Μεταξύ των πολλών θεμάτων που δείξατε, γιατί το Υπουργείο σα καλύπτει πολλού τομεί, όπω και αυτή η Επιτροπή, εγώ θέλω να αναφερθώ στο ενεργειακό θέμα. Γνωρίζετε πολύ καλά ότι οι πυλώνες τη ενεργειακή πολιτική τη Ευρωπαϊκή Ένωση είναι να εγγυηθούμε την ασφαλεία του εφοδιασμού, την ανταγωνιστικότητα και την αηφορία. Δηλαδή, με άλλα λόγια, πρόκειται για το να μην εξαρτώμαστε από το εξωτερικό συνεργειακό επίπεδο. Δεύτερον, να είναι βιώσιμο το κόστος τη ενέργεια. Και τρίτον, να έχουμε καθαρές πηγές ενέργειας, δηλαδή ώστε να το χαμηλότερε εκπομπέ διοξιδίου του άνθρακα. Δεν υπάρχει εμβολία ότι η πυρηνική ε, ενέργεια είναι η μόνη αυτόχθονη ενεργική πηγή που πληρεί ταυτόχρονα αυτούς τους τρεις ε, στόχους. Είναι προφανές ότι στο ενεργειακό μείγμα η απόφαση για το ποσοστό της πυρηνικής ενέργειας είναι μια απόφαση που πρέπει να ληφθεί ανάλογα με τις αρμοδιότητες του κάθε κράτος μέλους. Αλλά εγώ θα ήθελα να αναφερθώ σε ένα θέμα για το οποίο η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει αρμοδιότητες και έχει να κάνει με την ασφάλεια ή πυρηνική ενέργεια σύμφωνα με το Ευρωβαρόμετρο 2008 χέρι μεγαλύτερη υποστήριξη και τώρα υπάρχει ε, σχεδόν υποστήριξη από το 50% ε, των πολιτών. Όμως υπάρχει ένα πολύ ενδιαφέρον θέμα που είναι το θέμα της ε, ασφάλειας και της διαχείρισης των αποβλήτων. Όταν ε, τίθεται ερώτηση για το θέμα αυτό αυξάνεται το ποσοστό αυτών που λένε ότι αν υπάρχει ένα σίγουρος τρόπος για τη διαχείριση και την αποθήκευση των αποβλήτων. Οι πολίτε που είναι υπέρ τη ελληνική ενέργεια αυξάνονται πάνω από το 60%. Όμω υπάρχει ένα, προσ... ένα πρόσθετο πρόβλημα ότι δεν υπάρχει πολύ μεγάλη πληροφόρηση για το θέμα αυτό. Υπάρχουν δύο χώρε, Βουλγαρία και Ουρμανία, νέα κρατημέλη. Αλλά υπάρχουν και δύο κράτη-μέλη πολύ παλιά, όπω είναι η Αυστρία και η Ισπανία, στην περίπτωση της Ισπανίας, ε, η πληροφόρηση που υπάρχει για το θέμα αυτό είναι ιδιαίτερα ελλειπής. Και καθώς η πληροφόρηση είναι βασικός πυλώνας για την ελευθερία λήψης αποφάσεων, τι θα κάνει η Ισπανική Προεδρία, δηλαδή εσείς τι θα κάνετε για να ε, βελτιώσετε την ενημέρωση για το θέμα της πυρηνικής ενέργειας και για τη διαχείριση ε, και αποθήκευση των πόρων. Η κυρία Μαδουρέλ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ κύριε Υπουργέ, εκ μέρους της ομάδας μου. Θα ήθελα και εγώ να σας καλωσορίσω στην Επιτροπή αυτή και να σας ευχαριστήσω και να σας συγχαρώ για την παρουσίαση του προγράμματος της Ισπανικής Προεδρίας. Ε, μας παρουσιάσετε και τι αρμοδιότητε του Υπουργείου σα, που είναι πολλέ και φυσικά αφορούν ε, τα μάλα της εργασίας αυτής της Επιτροπής. Ένα πρόγραμμα της Ισπανικής Προεδρίας που θεωρεί ε, η ομάδα μου φιλόδοξο και πολύ συναφές με τις αναγκαιότητες της Ευρωπαϊκής Ένωση, αυτή τη στιγμή. Βρισκόμαστε σε ένα πολύ συγκεκριμένο πλαίσιο που περιγράψατε πολύ καλά. Βρισκόμαστε μέσα σε μια πολύ μεγάλη οικονομική κρίση αναθεωρούμε την καθολική μας στρατηγική για την Ευρωπαϊκή Ένωση και θέτουμε σε εφαρμογή μια νέα συνθήκη που μεταξύ άλλων δίνει περισσότερες αρμοδιότητες στο Κοινοβούλιο αυτό και τη νομική βάση για να καθορίσουμε κοινέ πολιτικές σε απαραίτητου τομεί όπως ο ενεργειακός και σε σχέση με την ασφάλεια του ενεργειακού εφοδιασμού ε, έχει να κάνει η πρώτη μου ερώτηση μπροστά σε μια κρίση που ζούμε με την ε, Ρωσία και την Ουκρανία πρέπει να εντατικοποιήσουμε τα διπλωματικά ε, μέτρα αλλά ε, όταν βρεθήκαμε σε μια επίγουσα κατάσταση είδαμε ότι τελικά πρέπει να υπάρχουν εσωτερικά μέτρα αλληλεγγύης που να μας επιτρέπουν τον εφοδιασμό των υπόλοιπων κρατών μελών και έτσι λοιπόν γι' αυτό, αυτό που χρειάζεται μεταξύ άλλων είναι να υπάρχει μια ροή ενέργεια σε όλη την επικράτεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης και φτάνουμε λοιπόν στα θέματα της διασύνδεσης μεταξύ των κρατών μελών που αναφέρετε εσείς και αυτό είναι ένα θέμα που ανησυχεί πάρα πολύ αυτή την Επιτροπή. Εμείς ε, καταλάβαμε ότι αυτό θα αποτελέσει προτεραιότητα της Προεδρίας. Μπορείτε να εμβαθύνετε στο θέμα αυτό, γιατί όπως σας είπα είναι κάτι που το συζητούμε και μας απασχολεί εδώ και καιρό. Και πολύ σύντομα μια δεύτερη ερώτηση κύριε Υπουργέ. Αναφερθήκατε στην ενιαία ε, ψηφιακή αγορά κάθε φορά που προσπαθήσαμε να προχωρήσουμε προς την κατεύθυνση αυτή εμφανίστηκαν πάρα πολλά εμπόδια ε, στα κράτη-μέλη για το να υπάρχει πραγματική διασυνορική αγορά των ψηφιακών προϊόντων αναφέρατε ορισμένες από τις αιτίε των δυσκολιών αυτών. Αλλά τι θα κάνετε για να πείσετε το Συμβούλιο και ποιες δράσεις προτεραιότητα σκέφτεστε να θέσετε σε εφαρμογή για να καταστεί αυτό πραγματικότητα τα επόμενα έτη. Ευχαριστώ. Danke sehr. Εγώ σας ευχαριστώ. Κυρία Εκ. Also I want to welcome you on behalf. Και εγώ θα ήθελα να σας ευχαριστήσω, να σας καλωσορίσω κύριε Υπουργέ, εξ ονόματος της ομάδας μου, των Φιλελευθέρων. Και να σας ευχαριστήσω για την ωραία συζήτηση που είχαμε στη Μαδρίτη πριν από κάποιες μέρες θα ήθελα να αναφερθώ στο θέμα τη ενέργεια και της αποτελεσματική χρήση της ενέργειας. Ξέρουμε πόσο σημαντικό είναι αυτό. Ξέρουμε ότι θα πρέπει να έχουμε σύντομε προθεσμίε για να μπορέσουμε να δράσουμε σε αυτό το τομέα. Και το πρώτο τμήμα τη ερώτησή μου είναι το εξή. Τι θα λέγατε να κάνετε προτάσεις στη διάσκεψη κορυφής για το 2020 σχετικά με θέματα αποτελεσματικής χρήσης ενέργειας. Στη συνέχεια της ε, ε διάσκεψης Κοπεχάης θα πρέπει να σκεφτούμε και μια πολιτική που θα προχωρήσει την Ευρώπη ένα πρόγραμμα δράσης για θέσεις απασχόλησης, επίσης μέσα στα πλαίσια ε, του 2020. Και εδώ θα μπορούν να βρεθούν πολλές ε, λύσεις. Τέλος, την εφορία που η κυρία Καστέλο. Εσείς είσαστε εταίρος για την αηφορία, ιδίως εν ώψη των προτάσεων που υποβάλλει η Ισπανία αυτή τη στιγμή, που δεν είναι και πολύ αηφόρες από ό,τι το βλέπουμε εμείς. Ευχαριστώ. Φεμπράντ. Ναι, σας ευχαριστώ πρόεδρε. Θα ήθελα και εγώ να σας ε, καλωσορίσω θα ήθελα να σας πω ότι αυτή η Επιτροπή θα σας υποστηρίξει και εσάς και τις φιλοδοξίες σας γιατί, για την ενέργεια και εγώ από μια βόρεια χώρα. Ενδιαφερόμαστε ιδιαίτερα για την ελοική ενέργεια στην Βόρεια Θάλασσα και επίσης ε, θέλουμε να υποστηρίξουμε την ηλιακή ενέδρα. Ένα πολύ επίκαιρο θέμα που θα ήθελα να θίξω είναι το εξής. Επισκέφτηκα χθες είναι το κοντά στην Αμβέρσα. Ξέρετε φαντάζομαι τι θα πω. Ξέρετε ότι γίνεται πάρα πολύ αναδιάρθρωση εκεί και πρόκειται να κλείσει μια ε, επιχείρηση και λέγεται ότι δεν σχετίζεται αυτό με την απόδοση ή την παραγωγικότητα αλλά ότι η επιχείρηση αυτή, το εργοστάσιο μάλλον αυτό της επιχείρησης, κλείνει για πολιτικούς λόγους. Και γι' αυτό οι εργαζόμενοι στην Όπελ εκεί εξετάζουν προσεκτικά τι θα κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Κομισιόν πάντα ήταν φιλόδοξη στην οθέτηση μέτρων για την εσωτερική αγορά, αλλά δεν είναι και τόσο φιλόδοξη όταν πρέπει να εξασφαλίσει και οι επιχειρήσεις να αναλάβουν τις δικές τους ευθύνες μέσα στα πλαίσια αναδιορθώσεων. Από ό,τι ξέρουμε, η Όπελ πρόκειται να ζητήσει κρατικές ενισχύσεις ε, για τα εργοστάσια της και θα πρέπει η Κομισιόν να φροντίσει να γίνει αυτό σύμφωνα με όλους τους κανόνες του παιχνιδιού. Αυτό το θέμα είναι η σημασία διάταξη επίσημη ε, ε, συνόδου του Συμβουλίου. Τι πρόκειται να κάνετε για να υπάρχει ομοιομορφία στην εφαρμογή των κανόνων. Και τέλος, οι εργαζόμενοι του Στενόπελτ δείχνουν αλληλεγγύη μεταξύ τους και τι θα κάνετε εσείς για να σας υποστηρίξετε. Και τέλος, Πρόεδρε, αναφέρονται όλοι στην ελεύθερη στην ε, σύμβαση συγγνώμη ελευθερών συνολογών με την Νότιο Κορέα που συμπεριλαμβάνει διάφορε βιομηχανίε, παραδείγματο χάρη και την αυτοβιομηχανία, παραδείγματο χάρη και την όπλη. Τι θα κάνει η Κομισιόν και το Συμβούλιο για το θέμα αυτό. Ευχαριστώ, ε, Ευχαριστώ κύριε Φανιάν. Ευχαριστώ, Πρόεδρε, κύριε Υπουργέ. Και εγώ θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για την ε, ευρεία παρουσίαση της των προτεραιοτήτων της Ισπανικής Προεδρίας, ε, των θεμάτων που εμπίπτουν στην αρμοδιότητά σας, αλλά θα αλλάξω θέμα. Θα ήθελα να σας ρωτήσω κάτι για τις τεχνολογίες ε, επικοινωνιών και πληροφοριών. Όπως ξέρετε, τον Νοέμβριο στο Σάλμα στην Αίγυπτο έλαβε χώρα το Φόρουμ ε, Διαχείρισης του Διαδικτύου. Ένα από τα κύρια θέματα ήταν ε, η ασφαλεία στον χώρο Και εδώ εντάσσεται το θέμα της ασφάλειας του διαδικτύου για τα παιδιά μπορέσαμε να συζητήσουμε με πολλές οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών που είχαν αυτή την ανησυχία. Και με ικανοποίηση διαβάζω ότι μία από τις προτάσεις της Προεδρίας σας είναι η υιοθέτηση της χάρτας για τις ΤΑΦΠΕ, για την ασφάλεια των χρηστών. Και θα ήθελα να μου πείτε αν η Προεδρία σας ε, σκέφτεται να αναλάβει κάποια συγκεκριμένη δράση για να αποφευχθούν οι κίνδυνοι του διαδικτύου για τα παιδιά, γιατί όπως ξέρουμε ε, κάθε μέρα είναι όλο και μικρότερη ηλικία χρήστες ε, του διαδικτύου. Αυτό έχει να κάνει με την εκπαίδευση των παιδιών, την παιδεία των γονιών και των εκπαιδευτικών. Θα ήθελα να ξέρω, έχετε προβλέψει κάποια πρωτοβουλία προς αυτήν την κατεύθυνση. Ευχαριστώ. Συνάδελφος Κέδεκ. Σας ευχαριστώ, Πρόεδρε. Κύριε Υπουργέ, εδώ και πολλά χρόνια ε, βλέπουμε από την Ευρώπη να φεύγουν διάφορα εργοστάσια και να μετατοπίζονται. Για λόγους οικονομικούς πολλά προϊόντα δεν παράγονται πια στην Ευρώπη, αλλά κάπου. Στην Ασία. Αυτό αφορά την ε, προστοϊφωνική βιομηχανία, αλλά και άλλους κλάδους βιομηχανίας. Και επίκειται ένα άλλο κύμα μεταδοποίησεων ε, επιχειρήσεων ε, λόγω του υψού των τιμών της ενέργειας. Και αυτό θα είναι κάτι που θα μας απασχολήσει σίγουρα. Και φανερόμαστε ότι τελικά δεν θα είναι μόνο οικονομική αυτή η μετατόπιση, θα είναι και πολιτική. Η συνάδελφος αναφέρθηκε στην Όπελ, στην Αμερικανία παραδείγματο χάρη. Fiat, το Fiat το πολωνικό λέγεται για πολιτικούς λόγους, όχι για οικονομικούς, για πολιτικούς λόγους θα μεταφέρει πάλι την παραγωγή εν μέρη στην Ιταλία. Το ίδιο ισχύει και για την Χαλιβουργία γενικά. Τι σκοπεύει να κάνει η Ισπανική Προεδρία, πώς θα το αντιμετωπίσει, πώς θα αντιμετωπίσει αυτά τα προβλήματα που δεν είναι καθόλου σχετικά με την ανταγωνιστικότητα. Ευχαριστώ. Θα κάνουμε μια διακοπή και θα έχει τη δυνατότητα ο Υπουργός να απαντήσει στι ερωτήσει. Παρακαλώ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Σας ευχαριστώ για το καλό όρισμα. Ευχαριστώ τα μέλη της Επιτροπής σας που μου καλωσόρισαν. Για τις πρώτες ερωτήσεις από την κυρία Δεκαστήγιο. Η ενεργειακή πολιτική σε ό,τι αφορά την πυρηνική ενέργεια είναι απόφαση των κρατών μελών. Και επομένω η Προεδρία λογικά θα είναι ουδέτερη έναντι των προτάσεων είτε για διεύρυνση είτε για ανανέωση που θα θετήσουν τα κράτη-μέλη. Τώρα, σε ό,τι αφορά την ασφάλεια της πυρηνικής ενέργειας και τη διαχείριση των αποβλήτων, εργαστήκαμε στο εσωτερικό της Ισπανίας, τη μεταφορά των οδηγιών των στο εσωτερικό δίκαιο και Κατά τη διάρκεια της Προεδρίας μας αναμένουμε να παρουσιάσουμε ένα πρώτο σχέδιο ε, για τα ενεργά απόβλητα και τη διαχείριση των αποβλήτων αυτών, ένα σχέδιο οδηγίας που θα θέσουν ε, τις ε, ομοιόμορφες προϋποθέσεις έτσι ώστε να υπάρχει ασφαλής διαχείριση των ε, καυσίμων αυτών και των πυρηνικών αποβλήτων. Εγώ δεν συμφωνώ με αυτό που είπατε ότι η πυρηνική ενέργεια είναι μόνο η καθαρή και αυτοθόνα ενέργεια που μπορούμε να έχουμε στην Ευρώπη. Έχουμε και άλλε εναλλακτικέ πηγέ ευτυχώ. Μία από αυτέ είναι οι ανανεώσιμε πηγέ ενέργεια. Άλλες ε, είναι εξοικονόμηση για ενεργειακή αποδοτικότητα. Σκεφτείτε την Ισπανία ως παράδειγμα. Εμείς έχουμε 20% ε, παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από την πυρηνική ενέργεια και το να εξοικονομήσουμε το 20% στην κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας μπορούμε να το κάνουμε με μέτρα εξοικονόμησης θα σήμαινε ότι ε, θα διπλασιάσουμε τις ε, πυρηνικές εγκαταστάσεις με δύο πλεονεκτήματα. Καταρχήν ε, δεν κοστίζει τίποτα, είναι δωρεάν και όχι μόνο αυτό, μάλιστα κερδίζει κανείς και χρήματα γιατί ουσιαστικά αντικαθιστούμε εισαγωγές ενέργειας και ε, δεν έχουμε μεταφορά κέρδους. Απλώς ε, δημιουργείται κέρδος στο εσωτερικό και θέσεις απασχόλησης. Και επίσης δεν υπάρχει και πρόβλημα αποβλήτων. Έτσι λοιπόν η ενεργειακή εξοικονόμηση είναι μία από τις κύριες πηγές ενέργειας που πρέπει να εκμεταλλευτούμε στην Ευρώπη. Αλλά επίσης και η διανθεσιμότητα και οι υποδομές και θα απαντήσω έτσι στην απάντηση της ε, κυρίας Βιέρα για τις ε, διασυνδέσεις ε, στο εσωτερικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης αλλά και των διευρωπαϊκών δικτύων, των διασυνδεσμικών δικτύων. Αυτό αποτελούν ένα στοιχείο που ευνοούν, αγγιώνται την ασφάλεια του εφοδιασμού και ευνοούν και την ανταγωνιστικότητα. Σκεφτείτε το αέριο που θα έρθει από την Αλγερία μέσω της Ισπανίας, μέσω από τη MedGas, ε, μπορούμε αντί για 8 να έχουμε αμέσως 16 ε, κυβικά μέτρα, 10 κυβικά μέτρα αν σκεφτούμε ότι ε, θα φτάσει το αέριο αυτό στη Βόρεια και Ανατολική Ευρώπη έναντι του αερίου που προέρχεται από τη Ρωσία. Και αντίθετα, αν το αέριο από τη Ρωσία φτάσει στις χώρες του Νότου, αυτό θα μειώσει το κόστος της τιμής του αερίου. Έτσι λοιπόν, ε, οι διασυνδέσεις δεν είναι μόνο καλές για την ασφάλεια του εφοδιασμού, αλλά είναι καλές και για την ανταγωνιστικότητα, γιατί μειώνουν το κόστος, την τιμή της ενέργειας. Ε, είναι καλές για να έχουμε διαπραγματευτική δύναμη με τις χώρες προμηθευτές. Ε, δηλαδή είναι σημαντική συνιστόσα η μείωση της τιμής και φυσικά συνεισφέρουμε και στην ανταγωνιστικότητα και στην ευημερία των πολιτών μας με τις διασυνδέσεις αυτές και με τα διασυνοριακά δίκτυα. Απαντώ λοιπόν στην κυρία Ριερέτση. Η προτεραιότητά μας είναι να ενδυναμώσουμε τα διευρωπαϊκά δίκτυα για τη μεταφορά ενέργειας, αλλά και τις διασυνδέσεις στο εσωτερικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει έξι μεγάλα σχέδια διασύνδεσης και εξωτερικής σύνδεσης που είναι ουσιαστικά για να εγγυθούμε την ενεργειακή ασφάλεια και ελπίζουμε ότι η Κομισιόν φέτος θα παρουσιάσει τα απαραίτητα μέτρα για τη θέση σε εφαρμογή σε λειτουργία τέτοιων ε, έργων, τέτοιων project. Φυσικά η Ισπανική Προεδρία θα στηρίξει ανάλογα. Επίσης, για την προώθηση των ενεργειακών υποδομών, η Προεδρία έχει το στόχο να συνάψει μια συμφωνία επί της ρύθμισης της κοινοποίησης επενδυτικών σχεδίων σε ενεργειακές υποδομές. Ελπίζουμε ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα συμφωνήσει με την ε, γνωμοδότηση του Συμβουλίου το συντομότερο, έτσι ώστε το Συμβούλιο να μπορέσει να λάβει υπόψη αυτή τη γνωμοδότηση και να θετήσει την κατάλληλη νομοθεσία. Επιπρόσθετα, η Κομισιόν φέτος θα μπορούσε να παρουσιάσει ένα νέο νομοθετικό μέσο για τις ε, υποδομές, για την ασφάλεια του εφοδιασμού. Η πρόταση αυτή θα μπορούσε να συμπεριλαμβάνει την αναθεώρηση ε, της ρύθμισης TNC. Και επίσης και η αποθήκευση είναι σημαντική για την ε, ασφάλεια ε, του εφοδιασμού σε ό,τι αφορά το πετρέλαιο. Ξέρετε, ε, το Νοέμβριο τέθηκε σε ισχύ η οδηγία ε, για την ε, ελάχιστη υποθήκευση πετρελαίου ή πετρελαϊκών προϊόντων. Το σημαντικό είναι η δημιουργία ομάδας συντονιστών για το πετρέλαιο και τα πετρελογικά πετρελαϊκά προϊόντα, παρόμοιο με τον Gas Coordination Group, την ομάδα των συντονιστών για το αέριο. Σε ό,τι Μάλλον θα συνεχίσω με το θέμα της ενέργειας και κατόπιν θα δούμε τα ψηφιακά θέματα. Ε, η κυρία Εκ ε, αναφέρθηκε στο θέμα της ενεργειακής ε, αποδοτικότητας, όπως σας είπα είναι ζωτικό θέμα, γιατί για μας είναι ένα από τα μεγάλα εργαλεία, από τις μεγάλες πηγές ενέργειας που έχουμε στην Ευρώπη. Θεωρούμε ότι στο πρόγραμμα της Προεδρίας καταρχήν πρέπει να προσεγγίσουμε το σχέδιο δράσης ενέργειας 2010-2014, δηλαδή το σύνολο, και κατόπιν να έχουμε την αναθεώρηση του σχεδίου ενεργειακής αποδοτικότητας που πρέπει να αποτελεί τμήμα αυτού του καθολικού σχεδίου ενέργειας. Όμως το σχέδιο δράσης ενέργειας πρέπει να περιλαμβάνει τις κυρίες γραμμές ε, βάσει των οποίων θα πρέπει να εργαστούμε η Ισπανία, ανάλογα και με το χρονογραφείο τη Κομισιόν, οι υπόλοιπε προεδρίες, ε, Βέλγιο ή Ουγγαρία θα ασχοληθούν με το θέμα αυτό που όπως σας είπα είναι πολύ σημαντικό για την ενέργεια στην Ευρώπη. Και επίσης ε, έχουμε και τον ε, Οργανισμό των Ρυθμιστικών Αρχών που φυσικά υποστηρίζουμε και θέλουμε να προωθήσουμε. Σε ό,τι αφορά τώρα στο θέμα του άνθρακα, αναφερθήκατε στο θέμα του άνθρακα, ο Ευρωπαϊκός Κανονισμός ε, για τον Άνθρακα λύγει στα τέλη του 2010. Έτσι λοιπόν πρέπει να εκπονήσουμε ένα νέο κανονισμό. Θεωρούμε ότι οι προϋποθέσεις που επέτρεψαν την έγκριση το 2002 συνεχίζουν να ισχύουν οι συνθήκε αυτές και δεδομένου ότι οι συνθήκε του ενεργειακού τομέα στην Ευρώπη δεν έχουν αλλάξει ουσιαστικά από την έγκριση του τελευταίου κανονισμού το 2002, φαίνεται λογικό να σκεφτούμε επέκταση, επιμήκυνση του κανονισμού. Ε, θα μπορούσαν να τα συζητηθούν τα στοιχεία ε, της επέκταση του κανονισμού με τα κράτη-μέλη, αλλά η Ευρώπη θα πρέπει να έχει στοιχεία που θα μπορούν να εγγυηθούν την ασφάλεια του εφοδιασμού. Δηλαδή έχουμε το θέμα της ασφάλειας του εφοδιασμού που θα πρέπει να χρησιμεύει και σαν ένα backup με τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας γιατί ξέρουμε ότι η διαχείριση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας ενώ δεν έχουμε τεχνολογικά, ε, τεχνολογικές εξελίξεις, δηλαδή αν δεν έχουμε αναπτύξει το ηλεκτρικό αυτοκίνητο που θα μας βοηθήσει να διαχειριστούμε ε, και το ηλεκτρικό σύστημα χρειαζόμαστε ένα backup και αυτό το backup ε, θα πρέπει να το έχουμε είτε με τη μορφή πυρηνικής ενέργειας που είναι πιο δύσκολο να το διαχειριστούμε ή θα έχουμε το backup του άνθρακα. Έτσι λοιπόν ε, πρέπει να έχουμε ένα backup, αν και φαίνεται κάπως παράδοξο. Θα πρέπει όμως αυτό να συνοδεύεται πάντα με την ανάπτυξη των ε, ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Μόνο από αυτή τη σκοπιά θεωρούμε ότι είναι απαραίτητη διεύνηση ή επέκταση του κανονισμού για τον άνθρακα. Κύριε Βαν αναφερθήκατε στο θέμα της Όπελ. Εμείς ως κράτος μέλος καταρχήν και τώρα ως Προεδρία πάντοτε υπερασπιζόμασταν ότι το πρόβλημα της Όπελ είναι ευρωπαϊκό πρόβλημα και επομένως θα πρέπει να δοθεί μια ευρωπαϊκή λύση. Γι' αυτό ευνοήσαμε και θα συνεχίσουμε να το πράττουμε, θα συνεχίσουμε να βρούμε το διάλογο μεταξύ ευρωπαϊκών χωρών και με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή προκειμένου να συζητήσουμε μια ευρωπαϊκή λύση για την Όπελ. Η όπελ μπορεί να είναι κερδοφόρος, μπορεί να είναι ένα σχέδιο για το μέλλον. Αλλά φυσικά θα πρέπει να υπηρεσίσουν τα κριτήρια της ανταγωνιστικότητας, τα βιομηχανικά κριτήρια και ποτέ εθνικά κριτήρια κριτήρια χώρα. και έτσι λοιπόν η Ισπανική Προεδρία πάντοτε θα υποστηρίζει την ευρωπαϊκή διάσταση του προβλήματο Όπελ αλλά χωρίς να ξεχνάμε ότι η Όπελ πρέπει να είναι ανταγωνιστική και αποδοτική επιχείρηση. Έτσι λοιπόν οι αποφάσεις αναδιάρθρωσης θα πρέπει να συμπεριλαμβάνουν και αυτή τη συνιστόσα ανταγωνιστικότητα και κερδοφορία. Για τη Συμφωνία Ελευθερου με την Κορέα με την Νότια θα προωθήσουμε την προσωρινή εφαρμογή αυτής της συμφωνίας ε, σε στενή συνεργασία με τους κύριους βουλευτές και με την Κομισιόν σε ένα πλαίσιο διαφάνειας και συμμετοχής σύμφωνα με τις συνθήκες. Η συμφωνία λαμβάνει υπόψη το ψήφισμα του Κοινοβουλίου του 2007 για την αυτοκινητοβιομηχανία προβλέπει ουσιαστικά σταδιακή μείωση των δασμών, περίοδος 3 και 5 ετών ανάλογα με το μέγεθος των αυτοκινήτων και η Κορέα προσχέθηκε να άρει τα εμπόδια με την αποδοχή της ισοδυναμίας των ευρωπαϊκών κανόνων ασφαλείας Πρωτύπων ασφαλείας. Δεσμεύτηκε η Κορέα να ερμηνεύσει ε, τα πρότυπα αυτά, τους κανόνες αυτούς για να μην υπάρχουν προβλήματα πρόσβασης στην αγορά. Και το θέμα της Ευρωπαϊκής Βιομηχανικής Πολιτικής, στο οποίο αναφέρθηκε ο κύριος Γέρεκ. Θα αναφερθώ σε αυτό πρώτο και κατόπιν ε, θα αναφερθώ στο ψηφιακό ζήτημα για τη βιομηχανική πολιτική. Η Ισπανία έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον να δημιουργηθεί μια συζήτηση που θα αναλύσει τα αποτελέσματα των βιομηχανικών πολιτικών που υλοποιήθηκαν στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ένας Ισπανός πολιτικός είπε ότι η καλύτερη βιομηχανική πολιτική είναι αυτή που δεν υπάρχει. Όμως εμεί δεν συμφωνούμε με την άποψη αυτή. Θεωρούμε ότι πρέπει να υπάρχει βιομηχανική πολιτική μια βιομηχανική πολιτική που να έχει στο, ως στόχο την καινοτομία και την ανταγωνιστικότητα σε ένα κόσμο γεμάτο με προκλήσεις, σε ένα παγκοσμιοποιημένο κόσμο. Έτσι λοιπόν αναμένουμε ότι για να δημιουργηθεί η συζήτηση αυτή, να ξεκινήσει η συζήτηση αυτή, να εκπονηθεί ένα έγγραφο για το Συμβούλιο Ανταγωνιστικότητας του Μαρτίου. Εκπόνηση του εγγραφού αυτού γίνεται σε συνεργασία της Προεδρίας με τη ΓΑΜΑ Επιχειρήσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Βέβαια, η στήριξη στην ε, ευρωπαϊκή βιομηχανία θα πρέπει να γίνει από τη σκοπιά της στήριξη ε, στην ποιότητα, της, ε, στην ανταγωνιστικότητα, στο σχεδιασμό και στην ύπαρξη προϊόντων προστιθέμενης αξίας που μας επιτρέπουν να είμαστε ανταγωνιστικοί. Αυτή η ευρωπαϊκή βιομηχανική πολιτική μας επιτρέπει να, είμαστε, να είναι ένας από τους άξονες της στρατηγικής για το 2020 δηλαδή τη στρατηγική, κατόπιν της στρατηγικής της που θα πρέπει να συζητηθεί από τους υπουργού στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και τους πρωθυπουργούς στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. Σε ό,τι αφορά την νέα ψηφιακή αγορά, στην οποία αναφέρθηκε η κυρία Ριέρα. Θεωρούμε ότι εξακολουθούν να υπάρχουν πολλά εθνικά κολλήματα που εμποδίζουν ε, την ε, αποτελεσματική λειτουργία της αγοράς ε, λόγου χάρη τα δικαιώματα της πνευματικής δεξίας και οι άδειε που συνεχίζουν να είναι βασικά εθνικές. Πιστεύουμε ότι θα ήταν καλή μια εναρμόνιση σε ευρωπαϊκό επίπεδο να έχουμε και τη δυνατότητα να δίνονται άδειε που να ισχύουν σε πολλές επικράτειες. Επίσης, ε, να προωθήσουμε τη διαλειτουργικότητα διαφόρων συστήματων πληρωμής, ε, εφόσον βέβαια θα έχουμε σίγουρες οικονομικές συναλλαγές και προστασία των δεδομένων των καταναλωτών και των επιχειρήσεων. Όπως ξέρετε, μόνο το 7% των επιγραμμικών συναλλαγών είναι διασυνοριακές και θεωρούμε ότι εδώ υπάρχει πρόβλημα ασφάλειας στον χώρο που πρέπει να αντιμετωπίσουμε η απαραίτητη προστασία των καταναλωτών θα πρέπει να αποφύγει μέτρα που να κατακαιρματίζουν την αγορά. Επίσης πρέπει να αναλύσουμε τις ζημίες ε, που, επιφέρει, ε, που επιφέρουν οι προμήθειες ε, που ζητούνται όταν υπάρχουν παραδείγματος χάρη συναλλαγές επιγραμμικές, όταν λόγω χάρη αγοράζει κάποιο εισιτήρια στο διαδίκτυο για να παρακολουθήσει κάποια θεάματα. Ε, σε αυτά που αναφέρθηκε η κυρία Βαλία μας ε, ε, ανησυχεί η πρόσβαση των παιδιών στο διαδίκτυο. Χρειαζόμαστε συμφωνίες που να διασφαλίζουν την ασφάλεια στο ίντερνετ. Η προστασία των παιδιών μας φαίνεται πάρα πολύ σημαντική και θεωρούμε ότι πρέπει να ενδυναμώσουμε διαδικασίες εντοπισμού των ιστοσελίδων που δεν είναι κατάλληλες για παιδιά και σε ό,τι αφορά την εκπαίδευση πρέπει στο σχολείο να μαθαίνουν πώς να γίνεται μία ε, ασφαλής πλοήγηση τόσο τα παιδιά όσο και οι γονείς και θα πρέπει η Ευρωπαϊκή Ένωση ε, να παρακολουθεί αυτές τις σελίδες που δεν είναι κατάλληλες για τα παιδιά. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ πολύ. 11 έχουν ακόμα ζητήσει το λόγο. Μπορούμε να είμαστε ακόμη πιο σύντομοι για να προφτάσουμε να δώσουμε το λόγο σε όλους. Γιατί δεν έχουμε πάνω από μισή ώρα. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για την παρουσίασή σας. Äh, και Ασκήσατε λοιπόν κριτική και είπατε ότι θα πρέπει να υπάρχει ένα ε, βιώσιμο μοντέλο της ε, εφόρου ανάπτυξης. Η πρακτική όμως ε, που ακολουθεί η Ισπανική Προεδρία δεν ταιριάζει με αυτά. Η Αντιπρόεδρος, κυρία Φερνάντες Τελαβέγκα, σήμερα ανακοίνωσε στην Ισπανία ότι μία από τις προτεραιότητες της Ισπανικής Προεδρίας είναι το να εγκριθούν, ε, να αποκτήσει τη συνένεση για νέες επιδοτήσεις, νέες ενισχύσεις για τον άνθρακα, που ήδη επιδοτείται σε μεγάλο βαθμό στην Ισπανία. Εγώ λοιπόν θεωρώ ότι αυτό δεν έχει καμία απολύτως σχέση με την αεφορία, τη βιώσιμη ανάπτυξη και την κλιματική αλλαγή. Και προστίθηκε κάτι άλλο. Ε, πρόκειται και για μια ιδιαίτερα δυσάρεστη μορφή προστατευτισμού. Γιατί ποιοτικά καθαρά ο ισπανικός άνθρακας είναι πολύ χειρότερος από τον πολωνικό που είναι και πιο φτηνός. Και ο ισπανικός άνθρακας ως ισπανικός άνθρωπος, άνθρακας επιδοτείται για να ε, βγάλει από την αγορά τον πολωνικό άνθρακα. Τι σχέση έχει αυτό με την αλληλεγγύη ή με την αηφορία. Σας ερωτώ ειλικρινά, είσαστε εν πάση περιπτώσει πρόθυμοι ως ισπανική κυβέρνηση να τηρήσετε την υποχρέωσή σας ε, για αλληλεγγύη και βιώσιμη ανάπτυξη. Δεύτερον, ε, εκφραστήκατε υπέρ της ε, κινητικότητας και με ενδιαφέρει η Ισπανική Προεδρία μέχρι το 2020 ποιο είναι το ποσοστό ε, που ε, επιθυμεί η ε, Ισπανική Προεδρία να επιτύχει σε ηλεκτρονική κινητικότητα ή mobility. Υπάρχει ένα συγκεκριμένο στόχος που θέλετε να επιτύχετε με αυτή την νομοθετική πράξη για μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Η κυρία Κολόνα Καμπογκίνσκα. για μικρομεσαιες επιχειρησεις Κύριε κυρια Υπουργέ, σας εύχομαι το ιδιαίτερα φιλόδοξο και πλούσιο πρόγραμμά σας να μπορέσετε να το υλοποιήσετε. Αυτό θα είναι το σημαντικότερο. Μιλήσατε διαμακρών για την ενεργειακή ασφάλεια, για τη διασφάνιση ε, εφοδιασμού με αέριο. Το πρόγραμμα Ναμπούκο είναι πάρα πολύ σημαντικό για πολλές χώρες όσον αφορά την ενεργειακή ασφάλεια. Όμως αυτό το πρόγραμμα δεν προχωρεί, διότι οι προμήθειες από το Αζερβαϊτζάν δεν μπορούν να διασφαλιστούν. Η Ρωσία ασκεί πίεση στο Αζερβαϊτζάν και επιθυμεί να ελέγχει τις πηγές αερίου που υπάρχουν ε, στη χώρα αυτή. Όμως το πρόγραμμα Ναμπούκο είναι πρόγραμμα κλειδί. Εσείς λοιπόν, η Ισπανία, τι πιστεύουν για όλα αυτά, τι προτίθεστε να κάνετε κατά τη διάρκεια της Προεδρίας σας για να αλλάξει η κατάσταση, μήπως ε, προτίθεστε να λάβετε κάποια μέτρα έτσι ώστε το ε, πρόγραμμα Ναμπούκο να ολοκληρωθεί ταχύτερα, μήπως προτίθεστε παραδείγματο χάρη να επισκεφτείτε το Αζερβαϊτζάν. Σας ευχαριστώ και που ήσασταν και σύντομοι. Επόμενη ομιλήτρια. Κυρία Καρβάλιο, ευχαριστώ Πρόεδρε, ευχαριστώ κύριε Υπουργέ. Θα ήθελα να αφαιρθώ στη σημασία της εσωτερικής αγοράς ανέργειας και στο θεμελιώδη ρόλο ενός ηλεκτρικού δικτύου σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Θα ήθελα να ρωτήσω για το πώς προωθούνται συγκεκριμένα σχέδια για την Βυρική Χερσόνησο, συγκεκριμένα έργα. Είναι πάρα πολύ σημαντικά αυτά για την Πορτογαλία, όπως η σύνδεση μεταξύ Πορτογαλίας και Ισπανίας και Ισπανίας και Γαλλίας σε ό,τι αφορά το ηλεκτρικό δίκτυο. Το δεύτερο σχόλιο και ερώτησή μου έχουν να κάνουν ε, με το ηλεκτρικό αυτοκίνητο. Είναι μία λύση μεταξύ άλλων ε, με πλεονεκτήματα ε, που βασίζονται στην μείωση των εκπομπών διοξιδίου του άνθρακα Επίσης υπάρχουν τεχνολογικά προβλήματα που έχουν να κάνουν με τη φόρτιση των μπαταριών και προβλήματα μελητίας που έχουν να κάνουν ε, με την ε, προμήθεια, με τον εφοδιασμό. Τώρα, για την ανταγωνιστικότητα θα διατηρήσει η Ευρώπη την ανταγωνιστική της ικανότητα έναντι ε, Κίνας και Ρωσίας για το ηλεκτρονικό αυτοκίνητο. Η Ευρώπη έχει ουσιαστικά ένα προβάδισμα. Είμαστε ε, σε πολύ καλή θέση σε σχέση με τις υποστημονικές έρευνες. Μήπως θα έπρεπε εδώ να θέσουμε και την εναλλακτική της ε, ε, χρήσης εσωτερικής καύσης με υδρογόνο. Θα ήθελα λοιπόν να μου πείτε ποια είναι η στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το ηλεκτρονικό αυτοκίνητο. ηλεκτρικό αυτοκίνητο. Ευχαριστώ. Ο κύριος Τσιμάνσκι. Ευχαριστώ πολύ. Θα ήθελα να θίξω και εγώ κάποια θέματα. Οι κρατικές επιδοτήσεις ε, για τον ισπανικό άρθρακα οδηγούν σε στρεβλώσεις ε, στην ε, αγορά της Ευρωπαϊκής Ένωσης και δεν υπάρχει και κανένα επιχείρημα, κανένας λόγος Εδώ παραβιάζεται η ευρωπαϊκή νομοθεσία. Και κάτι άλλο που αφορά στην ε, ηλεκτρονική αγορά. Από τη διεύρυνση, από το 2004, πολλοί πολίτες από την κεντρική και ανατολική Ευρώπη δεν μπορούν πλέον να απολαμβάνουν ε, υπηρεσίες ε, που προσφέρονται ηλεκτρονικά. Τι μπορεί λοιπόν να γίνει έτσι ώστε η ηλεκτρονική αγορά να είναι ανοιχτή και να προσφέρει τα, τα ίδια σε όλους τους πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ, κύριε Υπουργέ. Πολύ φιλόδοξο το πρόγραμμα που ανακοινώσατε και σας εύχομαι καλή επιτυχία κατά την εφαρμογή του. Εμένα με ενδιαφέρει ένα θέμα που συζητήθηκε διαμακρών. Ξεκινήσατε με την ολοκλήρωση των ε, δικτύων ηλεκτρικού ρεύματος ε, και αυτό δεν είναι ίσως τυχαίο γιατί ενδιαφέρει πάρα πολλούς. Εγώ έχω να υποβάλω μια σύντομη και συγκεκριμένη ερώτηση όσον αφορά στο θέμα αυτό. Δηλαδή, για την ολοκλήρωση των ε, ενεργειακών δικτύων ηλεκτρικού ρεύματος ε, και αερίου. Υπάρχει ενεργειακή νησίδα αλλά πολλές φορές δεν ε, προσελκύονται επενδύσεις γιατί ε, δεν είναι αποδοτικές, ε, δεν θα αποφέρουν κέρδος. Πρέπει λοιπόν να καλύψετε διάφορα στοιχεία, αλληλεγγύη, ασφάλεια, κέρδος. Σας ερωτώ λοιπόν, ως Προεδρία θεωρείτε ότι τέτοιου προγράμματα θα πρέπει να στηριχθούν περαιτέρω σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Οντί. Σας ευχαριστώ πρόεδρε. Σας ευχαριστώ κύριε Υπουργέ και σας καλωσορίζω. Δύο ερωτήσει. Ε, Μία θεσμική. Αναφερθήκατε στο ότι είσαστε η πρώτη ε, προεδρία μετά την ε, θέση ισχύ της σύνδεξης Λισαβόνας. Θα ήθελα να σας πω ότι υπάρχει κάποια διαφορά ανάμεσα στα χαρτοφυλάκια των επιτρόπων Εμείς εργαζόμαστε με δύο υπουργούς, με τέσσερις ε, επιτρόπους. Δεν θα υπάρχει κάποια στιγμή να υπάρχει κάποια συνοχή μεταξύ των χαρτοφυλακίων των υπουργών στα κράτη-μέλη, των ε, επιτρόπων και των κοινοβουλευτικών επιτροπών. Όσον αφορά τη δυνατότητα επίδραση ε, ε Ισπανία. Εγώ μου άρεσε πάρα πολύ η ομιλία του Πρωθυπουργού, αλλά απογοητεύτηκα σε ένα σημείο όσον αφορά το θέμα τη επίδραση που δεν μπορεί να έχει η Ισπανία στην ε, Αμερικανική Ήπειρο, εκτός Καναδά και ε, ΗΠΑ. γιατί έχουμε την Ιβυρική Χερσόνησο επικεφαλής και του Συμβουλίου και της Επιτροπής αυτή τη στιγμή όσον αφορά το εμπόριο, το τουρισμό, δεν μπορείτε κάτι να κάνετε προς όφελος της Ένωσης. Κολλήγη Τόμσον. Τόμσον. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Καλώς ορίσατε κύριε Υπουργέ. Θα τα πω τα υπόλοιπα στα αγγλικά. Ε, στα δανέζικα. Ε, ε, κοιτάξτε, όσον αφορά την ε, βιώσιμη ενέργεια και την ενεργειακή αποδοτικότητα, Έχουμε επιτυχεί πάρα πολλούς ε, στόχους εδώ στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Συμφωνήσαμε για το στόχο του 2020. Συμφωνήσαμε να μειώσουμε τις εκπομπές διοξιδίου του άνθρακα και υπάρχουν και δεσμευτικά όρια. Όσον αφορά όμω την ενεργειακή απόδοση, εκεί δεν υπάρχουν δεσμευτικοί στόχοι. Στι διαπραγματεύσει, λοιπόν, όχι κυβερνήσει, το Κοινοβούλιο έστειλε μια επιστολή στον κύριο Μπαρόζο και τον ρώτησε «Μα δεν μπορούμε να έχουμε ε, δεσμευτικούς στόχους ε, όσον αφορά στην ενεργειακή απόδοση. Δηλαδή, στη Δανία είχαμε μάρα πολύ καλή εμπειρία όσον αφορά άλλα θέματα. Γιατί δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι έτσι ώστε να μην είμαστε αναγκασμένοι να παράγουμε συνεχώς όλο και περισσότερη ενέργεια. Πρέπει οι στόχοι για την ενεργειακή απόδοση να είναι δεσμευτικοί, κυρίως μεσούσες της κρίσης. Γι' αυτό λοιπόν θέλω να γνωρίζω κατά πόσον η Ισπανική ε, Προεδρία είναι ε, διατεθειμένη να ορίσει δεσμευτικούς στόχους ε, για την ενεργειακή απόδοση. Και όσον αφορά ε, το ΙΚΑΤΕ, το διαδίκτυο, δεν είναι πάντα ε, περιεκτικό, αλλά πολλές φορές ε, δημιουργεί και αποκλεισμό. Πώς είναι δυνατόν να υπάρχει τεχνολογική εξέλιξη εάν οι άνθρωποι δεν έχουν τα προσόντα, τη δυνατότητα να συμμετέχουν και αυτοί. Πρόκειται κυρίως για την ανταγωνιστικότητα και για την απόκτηση προσόντων, πώς είναι δυνατόν να διασφαλίσουμε ότι όλοι οι Ευρωπαίοι θα έχουν πρόσβαση στο ίντερνετ. Μήπως αυτό μπορεί να γίνει μέσα από δωρεάν ε, ίντερνετ. Κύριε Υπουργέ, πριν από λίγα ε, χρόνια στο Eurosport υπήρχε η εξής ε, διαφήμιση. Spain, in Spain everything is under the sun. Όλα υπό τον ήλιο στην Ισπανία. Και νομίζω αυτό ισχύει κατά κάποιον τρόπο σε αλληγορία και για τη δική σας την εισήγηση. Ο άνθρακας, ο ε, καθαρός άνθρακας ε, θα πρέπει να προάγεται. Εσείς είπατε να ξεχάσουμε τα ορυκτά καύσιμα, όμως ε, μεσοπρόθεσμα δεν μπορούμε να τα ξεχάσουμε όλα αυτά. Και ως εκ τούτου εδώ υπάρχει μια αντίφαση. Μιλήσατε για ενεργειακή απόδοση στην Ισπανία, ανταυτού όμως ε, λέτε ότι δεν θέλετε να χρησιμοποιήσετε την πυρηνική ενέργεια, αλλά την αιωλική, παρότι η πυρηνική είναι πολύ πιο καθαρή ε, και δεν υπάρχει ιδιαιτερότητα ως προς το μέλλον της πυρηνικής ενέργειας. Ερωτώ λοιπόν, η Ισπανική Προεδρία θα αυξήσει τα κονδύλια με τα οποία μπορεί κανείς να διασφαλίσει την ασφάλεια της πυρηνικής ενέργειας και την ασφάλεια της διάθεσης των αποβλήτων. Αυτό είναι ένα πολύ συγκεκριμένο ερώτημα και θέλω να μάθω αν συμφωνείτε ή όχι. Ο κύριος Χατζημαρκάκης, κύριε Πρόεδρε, ε, καταρχήν συγχαρητήρια για αυτό που είπατε, που προβάλλατε ε, την ε, ηλεκτρονική, την ηλεκτρική κινητικότητα ηλεκτρική κινητικότητα. Εγώ ήμουν εισηγητής. Η ηλεκτρική κινητικότητα, χαίρομαι που έχει γίνει ένα κεντρικό σημείο των προσπανθιών σας. Σήμερα το πρωί είχαμε ανταλλαγή απόψεων με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και η Προεδρία θα πρέπει να ε, δώσει ιδιαίτερο βάρος στην ε, τυποποίηση. Να έχουμε τις ίδιες μπρίζες για τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα, τους ίδιους μετασχηματιστές ε, και την ίδια τάση σε ολόκληρη την Ευρώπη. Αυτό που μου κάνει εντύπωση είναι ότι σε αυτό το κόκκινο έντυπο που διανύμαται αποδίδεται ιδιαίτερη σημασία στο θέμα της επικοινωνίας, στην πληροφορική και στην επικοινωνία. Καλό αυτό ε, με την ενεργειακή πολιτική θα είμαστε πιο αποτελεσματικοί μόνο εφόσον ε, συνδυάσουμε την ηλεκτρονική αποτελεσματικότητα και η ΚΑΤΕ. Βεβαίως, θα ήθελα να επισημάνω ότι σε σχέση με την εφορία μας δεν πρέπει να είμαστε τυφλοί και να προσπαθούμε πάση θυσία να επιβάλλουμε αυτή την αυτοματοποίηση. Τελική ανάλυση δεν βλέπετε και ότι η κρίση αυτή ε, οδήγησε στο να χαθούν κάποια κονδύλια εις βάρος των πολιτών. Όλοι βέβαια αποσύρονται, λένε ότι το πρόβλημα ήταν ε, λογιστικό περισσότερο. Δεν πιστεύετε λοιπόν ότι παρότι υπάρχει κάποια εφορία θα πρέπει πολύ προσεκτικά και συνετά να ε, συνεχίσουμε συνεχίσουμε να διατηρούμε τον ε, έλεγχο στο διαδίκτυο προς του ανθρώπου. Ο κύριος Κορέδα Κάμπορ, κύριε Υπουργέ, μας άρεσε πολύ η παρουσίασή σας και ε, καθώς εγώ ήμουν ο τρίτος που ρώτησα για το ηλεκτρικό αυτοκίνητο, αυτό δείχνει το συμβολικό χαρακτήρα της ε, παρέμβασης του Πρωθυπουργού σας όταν αναφέρθηκε στο θέμα αυτό το ευρωπαϊκό ηλεκτρικό αυτοκίνητο αυτή τη στιγμή, αν δούμε το ε, θέμα της εισαγωγής στην αγορά, έχει καθυστερήσει εδώ και δύο χρόνια σε σχέση με τα ευρυδικά δηλαδή ε, αυτοκίνητα που έρχονται από τρίτες χώρες. Ε, τώρα η φιλοδοξία, ο στόχος για την Προεδρία σας ε, είναι να προβείτε σε ρύθμιση και να προσπαθήσετε να δώσετε κίνητρα στην ευρωπαϊκή βιομηχανία έτσι ώστε να παράξει καινοτόμο ηλεκτρικό αυτοκίνητο ή ε, φτάνετε και μέχρι το σημείο να δώσετε κίνητρα στις διαπραγματεύσεις ε, με τα κέντρα όπου υφίσταται ήδη αλλά οι εγκαταστάσεις βρίσκονται σε τρίτες χώρες. Κύριε Πρόεδρε, αγαπητέ Υπουργέ, θα ήθελα να σας ε, συγχαρώ για αυτό το φιλόδοξο πρόγραμμα που μας ε, παρουσιάσετε. Σας εύχομαι καλή επιτυχία στην εφαρμογή του προγράμματος και εύχομαι επίσης να συμβάλλετε στην ε, αύξηση της ανταγωνιστικότητας στον τομέα της βιομηχανίας και της ενέργειας. Μια άλλη ερώτηση. Πιστεύω ότι η χρηματοπιστωτική κρίση έπληξε κυρίως τις χώρες της Ανατολικής Ευρώπης. Κλείνουν η μία μετά την άλλη οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις, οι επενδύσεις ε, είναι όλο και πιο περιορισμένες και αυτό συμβάλλει στην αύξηση της ε, ανεργίας σε αυτές τις ε, περιοχές. Εσείς λοιπόν τι μέτρα προβλέπετε για να αντιμετωπιστεί αυτή η κατάσταση έτσι ώστε οι πραγματικά μικρές επιχειρήσεις να έχουν έστω κάποια ευκαιρία να ανταπεξέλθουν στον ανταγωνισμό. Πρόεδρος, αυτές ήταν οι ερωτήσεις κύριε Υπουργέ και έχετε την ευκαιρία σε 15 λεπτά να, πατήσετε, να απαντήσετε κατά το μάλλον ήτον σε όλες τις ερωτήσεις. Ευχαριστώ. Λοιπόν, να προσπαθήσουμε να είμαστε αποτελεσματικοί και αποδοτικοί και στον χρόνο, όχι μόνο σε ό,τι αφορά την ενέργεια. Τώρα θα μου δοποιήσω όλε τι ερωτήσει που έγιναν για το ηλεκτρικό αυτοκίνητο και πάλι σα ευχαριστώ για την υποδοχή του σχεδίου αυτού που είναι ένα πράγματι δύσκολο σχέδιο για το ηλεκτρικό αυτοκίνητο. Δεν θα αποτελέσει επιτυχία γιατί το θέλουν κυβερνήσει. ούτε γιατί το θέλουν όλε οι κυβερνήσει ε, ή το κοινοβούλιο ή η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, όχι το ηλεκτρικό αυτοκίνητο ούτε θα αποτελέσει επιτυχία για το θέλει βιομηχανία, η αυτοκίνητο βιομηχανία, η ενεργειακή βιομηχανία, η βιομηχανία των τεχνολογιών πληροφοριών και επικοινωνιών ή όλες τις τεχνολογίες μαζί. Όχι. Το ηλεκτρικό αυτοκίνητο θα αποτελέσει επιτυχία αν το θέλουν οι πολίτες. Έτσι λοιπόν, ε, αυτός πρέπει να είναι ο στόχος, να το θέλουν οι πολίτες. Και για να το θέλουν οι πολίτες, ε, καταρχήν πρέπει να υπάρχει καταλληλή ενημέρωση για τα πλεονεκτήματα ε, που ε, προϋποθέτει για την τσέπη τους, για την αποδοτικότητα, την κερδοφορία της χώρας τους, για την κερδοφορία της Ευρώπης, για τη δημιουργία θέσεων εργασίας και για τον πλανήτη. Καλό λοιπόν για την τσέπη, καλό για τη χώρα, καλό για την Ευρώπη, καλό και για τον πλανήτη. Και θα υπάρχουν ε, λίγα βιομηχανικά και οικονομικά στοιχήματα που να έχουν αυτό το πόκερ με τους άσους, δηλαδή και τους τέσσερις άσους που σας ανέφερα. Ε, είμαστε λοιπόν ενεκτοί στο να ε, βρούμε και ε, άλλα πλεονεκτήματα για να προσθεθούν σε αυτούς τους άσους και Βεβαίως ε, θα πρέπει να είναι προσβάσιμο στους πολίτες, θα πρέπει να είναι διαθέσιμο και θα πρέπει να είναι και άνετο και θα πρέπει να είναι και εύκολη και η επαναφόρτιση. Όμως ε, πέρα από τα περιβαλλοντικά πλεονεκτήματα που θα έχει το, το ηλεκτρικό αυτοκίνητο, εμείς ε, αν κάποια μέρα όλα τα αυτοκίνητα που χρησιμοποιούνται στην Ισπανία ήταν ηλεκτρικά, τότε σε ό,τι αφορά τις εκπομπές θα είχαμε ισοδυναμία με το να φυτευτούν 4,5 ε, δισεκατομμύρια δέντρα. Ποτέ δεν θα γίνει αυτό στην Ισπανία, δεν χωράνε όλα αυτά τα δέντρα. Αλλά αν κάποια μέρα, μια ουτοπική μέρα, σε 60, 70, 100 χρόνια φτάσουμε στο να είναι ηλεκτρικά όλα μας τα αυτοκίνητα, τότε θα μπορούσαμε να μιλάμε για κάτι τέτοιο. Μιλάμε για ένα πολύ μακροπρόθεσμο στόχο που μπορεί να έχει αποτελέσματα για το περιβάλλον που καμία άλλη πολιτική που να γνωρίζουμε σήμερα ε, μπορεί να πετύχει. Γιατί επιπρόσθετα το ηλεκτρικό αυτοκίνητο έχει πάρα πολλά πλεονεκτήματα ως προς την ενεργειακή ασφάλεια και πολλά πλεονεκτήματα σε ό,τι αφορά τη βιομηχανική ανάπτυξη για μια Ευρώπη που θα πρέπει ε, τελικά να φορτίσει τις μπαταρίες της στο βιομηχανικό τομέα. Αν ε, δεν θέλει τελικά να την υπερνικήσουν οικονομικά άλλες χώρες όπως χώρες από την Ασία που στοιχηματίζουν σημαντικά στη βιομηχανική ανάπτυξη με την καινοτομία γιατί το ηλεκτρικό αυτοκίνητο επιπρόσθετα θα έχει και σημαντικές εφαρμογές ε, στις ε, νέες τεχνολογίες πληροφοριών και επικοινωνιών ε, και αυτό θα σημαίνει ότι θα έχουμε και ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα για την Ευρώπη. Δηλαδή όσο περισσότερα διαβάζουμε για το ηλεκτρικό αυτοκίνητο τόσο περισσότερο μας αρέσει, αλλά τελικά τόσο θα βγούμε... Τελικά θα προσπαθήσουμε και να το προσπαθήσουμε μπορούμε να μιλάμε για 7 εκατομμύρια ηλεκτρικά αυτοκίνητα χωρίς να δαπανίσουμε τον ευρώ σε ηλεκτρικές υποδομές. Πώς δούμε να τα φορτίζουμε τη νύχτα. Έτσι λοιπόν έχουμε μια τεχνολογία που μπαίνει στην πρίζα. Δεν έχουμε τίποτα κατά του υβριδικού αυτοκινήτου, αλλά αν μπαίνει στην πρίζα μπορούμε να εισαγάγουμε όχι μόνο τεχνολογία επαναφόρτησης, αλλά και τη συνήθεια της επαναφόρτησης τη νύχτα και αυτό θα μειώσει ε, το κόστος ε, της ενέργειας για όλους τους πολίτες, ε, για όλους όσους χρησιμοποιούν το ηλεκτρικό αυτοκίνητο. Δηλαδή από τους εχθρούς, μέχρι και οι εχθροί του ηλεκτρικού αυτοκινήτου θα επωφεληθούν από το χαμηλότερο κόστος της ενέργειας, γιατί θα μειωθεί έτσι το ενέο κόστος στο σύστημα της παραγωγής και διανομής της ενέργειας. Έτσι λοιπόν ε, θα πρέπει να χρησιμοποιήσουμε αυτό το δυναμικό στην Ευρώπη. Πρέπει ε, να το αξιοποιήσουμε για να μην χάσουμε την ηγετική μας θέση στις τεχνολογίες επικοινωνιών και πληροφοριών. Πρέπει να κάνουμε μια προσπάθεια εναρμόνισης όχι μόνο στο θέμα της τεχνολογίας επαναφόρτισης, αλλά πρέπει να καταβάλουμε και μια προσπάθεια εναρμόνισης της πολιτικές ε, στήριξης ενίσχυση του ηλεκτρικού αυτοκινήτου. Πρέπει να υπάρχει συντονισμό ανάμεσα στι βιομηχανίε. δηλαδή ε, πρέπει η ενεργειακή βιομηχανία να καθίσει μαζί με την αυτομηχανία και με τη βιομηχανία τεχνολογιών και πληροφοριών και ε, να επικοινωνήσουν, γιατί σήμερα δεν επικοινωνούν και πολύ μεταξύ του. Πρέπει να επικοινωνήσουν για να καταστεί πραγματικότητα το ηλεκτρικό αυτοκίνητο. Φυσικά, λογικά μιλάμε και για κινδύνου, ασφάλεια ε, του εφοδιασμού, γιατί σήμερα δεν έχουμε την άμεση δυνατότητα να κατασκευάσουμε ηλεκτρικές μπαταρίες στην Ευρώπη. Όταν, επομένως υπάρχει ουσιαστικά μια συνιστός ενεργειακής εξάρτησης, ε, πρέπει να το δούμε και το θέμα αυτό. Όλα αυτά τα θέματα θα συζητηθούν στο Σαν Σεμπαστιάν. Θα παρουσιάσουμε ένα πρώτο έγγραφο που ελπίζουμε κάποιες γενικές γραμμές που ελπίζουμε ότι θα μπορεί να μεταφραστεί από την Κομισιόν σε μία ανακοίνωση για το Συμβούλιο Ανταγωνιστικότητα. Τώρα, σε ό,τι αφορά το θέμα του άνθρακα, μάλλον υπήρξε κάποια σύγχυση όταν μιλάμε για αυτόχθον άνθρακα για αυτόχθονα άνθρακα, μιλάμε για ευρωπαϊκό. Δεν κατάλαβα λοιπόν πολύ καλά να αναφερθήκατε στο άνθρακα από την Πολωνία, από την Ισπανία. Για μας δεν υπάρχει καμία διαφορά. Γιατί εμεί όταν μιλάμε για αυτόχθονα άνθρακα, μιλάμε για ευρωπαϊκό. Εμεί ε, θέλουμε να υπάρχει ένα ορθό στοίχημα. μέσω της Ευρωπαϊκής Οδηγίας. Πάντα προσεγγίζουμε από αυτή τη σκοπιά το θέμα του άνθρακα. Αναμένουμε την πρόταση της Κομισιόν, να κατανοούμε ότι υπάρχουν απαιτήσει ως προς τις δεμεύσεις ε, και η Ισπανία αλλά και άλλες χώρες ε, θέλουμε να διερευνήσουμε το θέμα του CCS, της δέσμευσης και αποθηκεύσης του άνθρακα και είμαστε ε, φυσικά ευαίσθητοι απέναντι στις κοινωνικές επιπτώσεις που θα προκύψουν από τον νέο κανονισμό. Όμως περιμένουμε την πρόταση της Κομισιόν βάσει τις οποίες θα εργαστούμε. Κύριε Οντή, αναφερθήκατε σε πιθανές ε, ασυνάφειες. Εμείς δεν πιστεύουμε ότι υπάρχει κάτι τέτοιο, αλλά υπάρχει διαφορά διαλόγου μεταξύ των διαφορών τομέων. Είναι δύσκολη η εναρμόνιση των ε, Υπουργικών Χαρτοφυλακίων όλων των κρατών μελών. Θα ήταν πολύ αποτελεσματικό, αλλά είναι πολύ δύσκολο να γίνει όλοι. Δυστυχώς βιώνουμε τις αρνητικές συνέπειες από αυτές τις αποκλήσεις. Ε, εγώ έχω, μπορεί να έχω ε, δύο ή τρεις ε, διαφορετικούς υπουργού άλλε χώρε με του οποίου θα πρέπει να συνδιαλεχθώ γιατί το δικό μου χαρτοφυλάκιο περιλαμβάνει και τον τουρισμό και τη βιομηχανία και το εμπόριο. Ε, βέβαια, μπορούμε να ευνοήσουμε το διάλογο, γιατί εγώ νομίζω ότι να μην τελματώνουμε είναι κάτι καλό για όλους. Εγώ πάντως συμφωνώ με αυτά που είπατε για τις ε, δυσκολίες ε, που υπάρχει σε ό,τι αφορά το διάλογο. Δεν ξέρω, Πρόεδρε, πόσο χρόνο έχω ακόμα. Κύριε Καρβάλιο, αναφερθήκατε στην Ιβυρική Χερσόνησο και στη σχετική αγορά. Εμείς είμαστε ικανοποιημένοι για το πώς λειτουργεί η Ιβυρική αγορά λειτουργεί σαν ενιαία αγορά. Έγινε μια προσπάθεια, ένα εγχείρημα αριθμιστικής εναρμόνισης, πολύ σημαντικό. Και συνεχίζουμε να έχουμε ένα πρόβλημα ως Ευρική Χερσόνησον με τη διασύνδεση με την υπόλοιπη Ήπειρο, με τη Γαλλία, μέσω της Γαλλίας. Έχουμε μια νέα ηλεκτρική διασύνδεση με τη Γαλλία και θέλουμε να ευχαριστήσουμε τις προσπάθειες του Επιτρόπου Μόντι αλλά και τη γαλλική πλευρά, τις προσπάθειες που κατέβαλαν για αυτή τη διασύνδεση. Είναι η πρώτη διασύνδεση που έχουμε την Ισπανία από την εποχή του Φράνκο. Μιλάμε για μια διασύνδεση που θα συμβάλλει στο να ε, έχει η Βυρική Χερσόνησο 6% από 3% ε, σε ό,τι αφορά την ε, διασύνδεση. Εμείς δηλαδή προσπαθούμε να αυξήσουμε το, διασυνδέσει. και γι' αυτό σας είπα ότι η βελτίωση των διασυνδέσεων ε, είναι όχι μόνο ένα εργαλείο για την ε, πρόθεση της νέα ευρωπαϊκής αγοράς του με αλλά ε, έχει και ως στόχο να βελτιώσει την ανταγωνιστικότητα της βιομηχανίας μας και την ευημερία των καταναλωτών. Σε ό,τι αφορά τις διασυνδέσεις με την Πορτογαλία, είναι υποκατασκευή οι γραμμές που έχουν σχεδιαστεί και ελπίζουμε να ολοκληρωθούν το 2014 και στο τομέα του αερίου μελετάμε τη διασύνδεση ε, με το βορρά, δηλαδή να περάσει ένας νέος ε, αγωγός αερίου από το βορρά. Και στα λίγα λεπτά μου μένουν θα ήθελα να φερθώ στον Αμπούκο. Όπως ξέρετε, στόχος του Ναμπούκο είναι να υπάρχει διαφοροποίηση των διαφορών οδών εφοδιασμού. Αυτός ο νέος ε, αγωγός αερίου θα εγγυηθεί την ασφάλεια του εφοδιασμού. Επομένως, θα το υποστηρίξουμε εμείς ως Προεδρία. Για τα θέματα των τεχνολογιών, πληροφοριών και επικοινωνιών. Το δίκτυο είναι μια καθολική, μια παγκόσμια δομή. Αναφερθήκατε στο ότι δεν μπορούν όλες οι χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης να έχουν πρόσβαση σε όλες τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες. Εμείς θεωρούμε ότι το δίκτυο είναι ε, ένα παγκόσμιο, μια παγκόσμια δομή. Κάθε φορά είναι και πιο δύσκολο να μπλοκαριστούν οι προσβάσεις και ο στόχος μας είναι να προωθήσουμε την ανάπτυξη μιας ενιαίας ψηφιακής αγοράς, ανοιχτής ψηφιακής αγοράς σε σχέση με αυτό που είπε η κυρία Τόμσεν σε ό,τι αφορά το δικαίωμα που έχουν οι πολίτες για καθολική υπηρεσία. Εμείς ε, είμαστε υπέρ ε, να χρησιμοποιείται καθολικά στην Ευρώπη ε, η ευρεία ζώνη. Στην Ισπανία έχουμε ένα μεγαμπάιτ ανά δευτερόλεπτο από το 2011 και πιστεύουμε ότι αυτό είναι ένα πολύ κατάλληλο εργαλείο που πρέπει να συμπεριλάβουμε στη στρατηγική της Γρανάδας. για τους προσωπικούς στόχους ενεργειακής αποδοτικότητας. Είναι πολύ δύσκολο να επιτευχθούν, κυρία Τόμψεν. Γιατί είναι διαφορετικά τα επίπεδα εφετηρίας κάθε χώρας. Τι πρέπει να κάνουμε, να ενδυναμώσουμε τις επιχειρήσεις ενεργειακών υπηρεσιών σε όλη την Ευρώπη, οι οποίες επιχειρήσεις θα είναι πολύ σημαντικές γιατί θα ε, βοηθήσουν τον τομέα των κατασκευών να γίνει ένας τομέας εφορίας ή ανάπτυξη των υπηρεσιών των επιχειρήσεων υπηρεσιών ε, ενέργειας στις ΗΠΑ, ε, στα με επιτυχία και εμείς θεωρούμε ότι αυτό το στοίχημα λοιπόν είναι πάρα πολύ σημαντικό και θα πρέπει να το υλοποιήσουμε στην Ευρώπη. Τώρα σε ό,τι αφορά τους προσωπικούς στόχους, με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον θα μελετήσουμε οποιαδήποτε πρόταση, αλλά είναι δύσκολα τα πράγματα, καθώς υπάρχουν διαφορετικά σημεία φετηρίας. Αλλά πρέπει και οι δημόσιες διοικήσεις αλλά και οι πολίτες και οι βιομηχανία να καταλάβουν ότι έχουμε ένα μεγάλο δυναμικό και ότι η καλύτερη ενέργεια του μέλλοντος είναι να προβούμε σε εξοικονόμηση ενέργειας. Συνεχίζουμε να εργαζόμαστε από αυτού και έτσι η Ισπανική Προεδρία μέσα στο σχέδιο δράση 2010-2014 ε, θα θέσει σε πρωταρχική θέσει το θέμα της ενεργειακής αποδοτικότητας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε Πρόεδρε, σας ευχαριστώ πάρα πολύ όλους για την υποδοχή σας, για τα σχόλια, τις ερωτήσεις σας και για τις παρεμβάσεις σας. Και εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ και σας ευχαριστώ που μας βοηθήσετε να κρατήσουμε και τα όρια χρόνου που έχουμε. Είμαι σίγουρος ε, κύριε Υπουργέ ότι θα ξαναειδωθούμε θα έχουμε κάτι να προετοιμάσουμε και να ολοκληρώσουμε μαζί. Και θα ήθελα να σε ευχηθώ και σε εσά και στην Ισπανική Προεδρία. Καλή δουλειά, καλή συνεργασία. Σας ευχαριστώ.